Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στη συνεδρίαση. Την πρωινή μας συνεδρίαση. Το πρώτο σημείο είναι κάτι που όλο και περισσότερο θα γίνεται σημαντικό. Ποια θα είναι η βιομηχανική πολιτική στην εποχή της παγκοσμιοποίησης, Ποιο θα είναι ο μελλοντικός ρόλος της Ευρώπης. Έχουμε δρομολογήσει μία έκθεση ίδιας πρωτοβουλίας και θέλουμε μια πρώτη και θελω μια σήμερα και θα ήθελα να καλωσορίσω το Γενικό Διευθυντή της Γενικής Διευθύνσεως για τη Βιομηχανία, τον κύριο Ζούρεκ και σίγουρα θα θέλει και αυτός να συμμετάσχει στη συζήτηση αλλά πρώτα απ' όλα θα ήθελα να δώσω στον εισηγητή τον κύριο Λάγκε το λόγο δώστε μας μια, δώστε μας μια γενική εικόνα κάντε μια παρουσίαση παρακαλώ Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Συνάδελφοι, κύριε Ζούρεκ. Η μηχανική πολιτική τα τελευταία χρόνια έχω δει, έχω διαπιστώσει ότι η εστίαση σε συντονισμένη βιομηχανική πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ήταν πάρα πολύ μεγάλη, δεν ήταν πολύ πετυχημένη. Σήμερα τονίζεται η ανταγωνιστικότητα, γενικά η ανταγωνιστικότητα και θεσπίζεται η σχετική νομοθεσία. Αλλά στατηγική, βιομηχανική πολιτική δεν έχουμε δει πάρα πολύ και δοθήσεις της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης νομίζω ότι έχει αλλάξει κάπου το επίκεντρο της προσοχής. Βεβαίως υπάρχει προστιθέμενη αξία όσον αφορά τη βιομηχανία. Τα τρία τέταρτα των εξαγωμένων προϊόντων είναι βιομηχανικά προϊόντα. 22% ε, ΦΠΑ προέρχεται από αυτή την, ε, τα έσοδα ΦΠΑ προέρχονται από αυτό τον τομέα και νομίζω ότι πρέπει να εστιαστούμε περισσότερο σε αυτό τον τομέα και χαίρομαι που μία από τις κατευθύντριες γραμμές όσον αφορά τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2020 σχετίζεται με την βιομηχανική πολιτική και δεν είχαν αναφερθεί τόσο ξεκάθαρα αυτά τα ζητήματα κάτω παρελθόν. Είναι επίσης σαφές ότι αντιμετωπίζουμε σημαντικές και συγκεκριμένες προκλήσεις που δημιουργήθηκαν τα τελευταία χρόνια. Βλέπουμε ότι η πίεση της παγκοσμιοποίησης έχει αυξηθεί σημαντικά, πιέζεται η ευρωπαϊκή βιομηχανία και υπάρχουν κάποιες περιοχές στον κόσμο, άλλα μέρη στον κόσμο που αναπτύσσονται και λαμβάνονται οι ανάλογες επενδυτικές αποφάσεις. Οπότε πρέπει πραγματικά να εστιάσουμε την προσοχή μας επί διατηρήσεως του βιομηχανικού μας πυρήνα στην Ευρώπη. Βλέπουμε ότι υπάρχει μεγαλύτερη παγκόσμια και διεθνή συνεργασία, παραδείγματο χάρη βιομηχανία σε παγκόσμιο επίπεδο και μηχανολογία σε παγκόσμιο επίπεδο και υπάρχει περισσότερη γνώση και μπορεί κανείς να ηγηθεί μόνο αν προβεί σε στενές ανταλλαγές γνώσεων με, με τον επιστημονικό κόσμο. Περνάμε λοιπόν από το φυσικό κεφάλαιο στο κεφάλαιο γνώσεων που αποτελεί τη βάση της βιομηχανικής ανάπτυξης. Οπότε βλέπουμε πρώτα απ' όλα μια αύξηση της παγκοσμιοποίησης, αυτό είναι το πρώτο, και δεύτερον έχουμε τις προκλήσεις τις οικολογικές. Πώς μπορούμε να ανανεώσουμε τον βιομηχανικό μας πυρήνα δοθήσεις της προκλήσεως της αλλαγής του κλίματος και των στόχων που έχουμε καθορίσει το φθινόπωρο του 2008 και υπάρχει και η άλλη πρόκληση της παραγωγής προϊόντων με τρόπο ε, φιλικότερο προς το περιβάλλον και με πιο αποδοτικό τρόπο στον αφορά πηγές που θα μας οδηγούσε σε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και βέβαια πρέπει να ανταποκριθούμε και στις δημογραφικές ε, αλλαγές. Η δημογραφική κατάσταση αλλάζει στην Ευρώπη και προφανώς η βιομηχανία θα πρέπει να ανταποκριθεί δεόντως. Πρέπει να δούμε και το πώς εξασφαλίζουμε ότι θα έχουμε επαρκές εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό στο μέλλον. Και υπάρχουν κενά όσον αφορά τις γνώσεις και τις δεξιότητες. Και αγαπητοί συνάδελφοι, η τέταρτη πρόκληση είναι η αναπτυσσόμενη ε, αστική ανάπτυξη που συνεπιφέρει νέες προκλήσεις όσον αφορά τα κτίρια, την οργάνωση, την επιμελητεία. Και, τη, και οι ίδιες οι παραγωγικές διαδικασίες αντιμετωπίζουν νέες προκλήσεις. Λοιπόν, θα πρέπει να ανανεώσουμε την βιομηχανική μας πολιτική και αντιμετωπίζουμε σημαντικές προκλήσεις και δεν είναι καθόλου εύκολο το έργο μας. Εδώ ακριβώς είναι το πρόβλημα. Η βιομηχανική πολιτική δηλαδή αντιμετωπίζει το εξή πρόβλημα. Δεν υπάρχει επαρκή συνεργασία. Έχουμε 307 κρατημέλη βεβαίω. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως διαπραγματευτή και πρωταγωνιστή, αλλά συντονισμένη δράση δεν υπάρχει. και βλέπω ότι είναι λογικό το συμπέρασμα στο οποίο καταλήγει το Συμβούλιο το Μάρτιο ότι πρέπει να ε, ξεπεράσουμε τα χάσματα και τις διαφορές μεταξύ των κρατών μελών. Περιμένω να δω βέβαια στην πράξη πώς θα ε, εφαρμοστεί αυτό. Ίσως το άρθρο 173 πρέπει να ενεργοποιηθεί και να αξιοποιηθεί πιο αποτελεσματικά και ίσως θα ήταν καλό να έχουμε μια στρατηγική καλή αλλά και ταυτόχρονα λειτουργική γιατί το να έχουμε μια καλή πολιτική η οποία δεν είναι λειτουργική δεν προσφέρει πολλά στη βιομηχανική πολιτική. Αγαπητοί συνάδελφοι λοιπόν, βλέπω ότι χρειάζεται μια νέα και ολοκληρωμένη προσέγγιση ε, για την βιομηχανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ολοκληρωμένη σημαίνει εν προκειμένου κοινέ θέσει για τους διάφορους τομείς πολιτικής που πρέπει να προσδιορίσουμε. Πολλές φορές έχουμε το πρόβλημα αυτό σε επιμέρους τομείς πολιτικής, περιβαλλοντική, εμπορική κτλ. Δεν, ε, η πολιτική η οποία αναπτύσσεται δεν συνάδει με τους βιομηχανικού μας στόχους. Αυτό λοιπόν πρέπει να εξασφαλιστεί αφενός, αφετέρου δε, οι διάφοροι ε, φορείς πρωταγωνιστής, πρωταγωνιστές της βιομηχανικής πολιτικής πρέπει να συμμετάσχουν στην πολιτική αυτή. Εάν δούμε λοιπόν τι είδους μέτρα απαιτούνται. Κάταρχας θα πρέπει να ενισχύσουμε την αλυσίδα της καινοτομίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η έρευνα η ανάπτυξη και και οι εφαρμογές με προσανατολισμό τη βιομηχανική εφαρμογή πρέπει να αναπτυχθούν πιο έντονα. Έχουμε εντυπωσιακά αποτελέσματα έρευνα συχνά με πολύ καλά πρότυπα εφαρμογών τα οποία όμως χάνονται στο δρόμο για τη βιομηχανική εφαρμογή. Δεν περνούν στην βιομηχανική εφαρμογή. Υπάρχει αυτή η ρήξη στην αλυσίδα δηλαδή της καινοτομίας. Και αυτό το γκρίκο θα πρέπει να αναπτύξουμε και πάλι, να επανασυνδέσουμε την αλυσίδα της καινοτομίας, ώστε να αναπτυχθεί η τεχνογνωσία στην Ευρώπη και πάλι και να εμφανιστεί ο στόχος βιομηχανικής πολιτικής σε κάθε τομέα ιδιαίτερα βέβαια στην έρευνα στις νέες τεχνολογίες όπως ανατεχνολογία και άλλες που θα πρέπει να ενισχύσουμε περαιτέρω. Δεύτερο σημείο, σχετικό με την αποτελεσματικότητα στη χρήση των πόρων. Από το 80 και έκτοτε έχουμε πλασιά στην αποτελεσματικότητα στην μηχανική μας παραγωγή. Όμως η αποτελεσματικότητα στην χρήση των πόρων δεν έχει αναπτυχθεί αντίστοιχα και η συμμετοχή του κόστου των πόρων στην βιομηχανική παραγωγή ανέρχεται σε 40%. Και γι' αυτό θα πρέπει, πιστεύω, να ενισχύσουμε την αποτελεσματικότητα της χρήσης των πόρων και ενεργειακά φυσικά, αλλά και στην χρήση των πόρων που χρειάζονται για την παραγωγή. Και έτσι εδώ αγαπητοί συνάδελφοι, ερχόμαστε στο εξή ότι εν γέννη οι πρώτες ύλε είναι περιορισμένες, σε παγκόσμιο επίπεδο είναι πεπερασμένες οι πρώτες ύλε, αφενός, αλλά και αφετέρου και βέβαια σχετικό, είναι πολύ μεγάλος ο ανταγωνισμός για το ποιο θα εξασφαλίσει την πρόσβαση στις πρώτες ύλε. Και ιδιαίτερα αν δούμε σε σχέση με την Κίνα, ε, η οποία αποτελεί μεγάλο ανταγωνισμό στην ε, διεκδίκηση πρώτων υλών, που φυσικά ενισχύουν ε, τις τιμές σε παγκόσμιο επίπεδο, ε, οθούν προς τα άνω τις τιμές σε παγκόσμιο επίπεδο. Έχουμε πολλά ακόμα να κάνουμε με συγκεκριμένα μέτρα. Και τρίτον, πιστεύω ακράδαντα ότι τα τομεακά συμφέροντα του βιομηχανικού κλάδου πρέπει να τα λαμβάνουμε πολύ πιο σοβαρά υπόψη. Είχαμε κάποιες προσεγγίσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Leadership, το STARS 21, το CARS 21, ε, μια Task Force ή άλλες Task Force ή υψηλού επίπεδου όργανα, τα οποία όμως μπορεί να προσέφεραν κάποια πλατφόρμα καινοτομίας χωρίς όμως στρατηγική ε, προσέγγιση και υλοποίηση των όσων συζητούσαν. Ή τουλάχιστον δεν έδιναν αρκετά σαφή εικόνα του τι, ποια θα έπρεπε να είναι η υλοποίηση αυτών που συζητούσαν. Και γι' αυτό νομίζω χρειάζονται σαφείς, ε, χρειάζεται σαφής διερεύνηση των αναγκών και των συμφερόντων του κάθε τομέα στη βιομηχανία ε, όσον αφορά την έρευνα και τις εφαρμογές να ακούμε δηλαδή τι έχει να πει η βιομηχανία και ταυτόχρονα να του αφήνουμε και ελεύθερου να επιλέγουν ε, πώς θα προχωρήσουν στι εφαρμογές. Για δε τα περιφερειακά πεδία δράσης ε, έχουμε πυρήνες βιομηχανικούς περιφερειακού χαρακτήρα οι οποίοι με μια καλή δικτύωση και με τον επιστημονικό χώρο μπορούν να προσφέρουν πολύ καλύτερα αποτελέσματα. Και νομίζω ότι εδώ έχουμε ένα κέριο ζήτημα της δικτύωσης της βιομηχανίας με την επιστήμη. Αυτά μπορούμε να τα ενισχύσουμε και αντίστοιχα να προσανατολίσουμε τις ε, επιλογές μας, τις αποφάσεις μας για επενδύσεις από πλευράς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ένα τελευταίο σημείο στο οποίο θέλω να φαρθώ, αγαπητοί συνάδελφοι, ήταν το να προκαταλαμβάνουμε τις εξελίξεις και την μεταλλαγή του βιομηχανικού τομέα, δηλαδή στους τομείς όπου έχουμε υπερβολική δυναμικό, υπερβολικές ικανότητες, θα πρέπει να προβλέψουμε την μετάλλαξη, χωρίς να θέλω να χρησιμοποιήσω τον όρο απεκβιομηχάνηση, θα ήθελα ψύχραμα να δούμε πώς μπορεί να μεταλλαγεί αυτός ο τομέας. Είτε πρόκειται για τα νέα κράτη-μέλη όπου έχουμε μεγάλες ε, και μαζικές ε, ε, δυνατότητες, πλεονάουσες δυνατότητες, είτε πρόκειται για τα παλαιά κράτη-μέλη, θα πρέπει να προ καταλάβουμε τις εξελίξεις, για να τις καθοδηγήσουμε και να μιλήσουμε ασφαλώς και για την αναδιάρθρωση εγκαίρως. Υπάρχει ένα μέσον, αλλά ασφαλώς θα πρέπει το ζήτημα της αναδιάρθρωσης να το εξετάσουμε με σοβαρότητα εγκαίρως και βέβαια συνοδευτικά θα πρέπει να έχουμε και μια πολιτική ε, ενσωμάτωσης, κοινωνικού χαρακτήρα δηλαδή πολιτική, που με δεδομένες και τις δημογραφικές εξελίξεις ε, σημαίνει ότι χρειαζόμαστε και υψηλής κατάρτισης και ειδίκευσης επιστήμονες και μια καλή πολιτική ενσωμάτωσης. Και ως γνήσιος δημοκράτης, ασφαλώς, εγώ τις εξελίξεις αυτές δεν μπορώ να τις δω ως ικανοποιητικέ παρά μόνο όταν υπάρχει επαρκής απασχόληση και αξιοποίηση, δηλαδή αυτός που έχει το δυναμικό, αυτός που έχει τη γνώση και την εξειδικεύση να απασχολείται εκεί ακριβώς όπου είναι χρήσιμο στη βιομηχανία. Ευχαριστώ πολύ. Ο Πρόεδρος, ευχαριστώ. Αν μου επιτρέπετε θα δώσω το λόγο στον εκπρόσωπο της Επιτροπής να ακούσουμε και τα δικά τους ε, σχόλια και μετά θα γίνει η συζήτηση. Ο κύριος Τσούρεκ, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Θα προσπαθήσω να σας ενημερώσω το δυνατόν πιο σύντομα για τις απόψεις επιτροπής στο θέμα αυτό. Καταρχάς βέβαια ευχαριστώ διότι το θέμα της παραγωγής και της βιομηχανίας είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να συζητήσουμε Όταν ανέλαβα εγώ τα καθηκοντά μου, είχαμε επιχειρήσεις οι οποίες θεωρούσαν ότι καλό θα είναι να μην εμπλέκεται η, η Επιτροπή, γιατί μας έβλεπαν ως old economy και ως ε, παλαιά φρουρά, ενώ τώρα βλέπουμε ότι θεωρούν χρήσιμη την παρουσία μας. Νομίζω λοιπόν ότι είναι σαφές για όλους ότι η οικονομική κρίση έχει ε, ιδιαίτερα ε, ορατά, ορατές συνέπειες στον από το χώρο της ε, παραγωγής προϊόντων, ιδιαίτερα στον κατασκευαστικό τομέα, που έχει υποχωρήσει κατά ένα πέμπτο μέσα σε ένα χρόνο και αυτή τη στιγμή φαίνεται ίσως μια αμυδρή ανάκαμψη, ίσως δηλαδή να τίνουν τα πράγματα προς βελτίωση, χωρίς βέβαια να ξέρουμε αν θα διατηρηθεί αυτή η τάση. Πάντως πέραν αυτού, η παραγωγή προϊόντων ε, είναι στο επίκεντρο της οικονομικής δραστηριότητας και ως εκ τούτου χρειάζεται να τη δώσουμε απόλυτη προσοχή και να ορίσουμε σαφείς στρατηγικές. Η αλήθεια είναι ότι η προστασία της βιομηχανικής παραγωγής, ε, η κατάσταση της βιομηχανικής παραγωγής στο τελευταίο καιρό ήταν λιγότερο στο επίκεντρο της προστοχής από ότι κάποιες ε, άλλες ανησυχίες όπως ε, παραδείγματι η περιβαλλοντική ρήπανση ή επιδείνωση της περιβαλλοντικής ποιότητας λόγω της βιομηχανικής παραγωγής και άλλες αντίστοιχες ανησυχίες. Ε, ωστόσο, η παραγωγή προϊόντων έχει πάρα πολύ ανησυχιες σημασία. Εμείς έχουμε ασχοληθεί από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τους επιμέρους τομείς. Παρακολουθούμε ποιες είναι οι μακροπρόθεσμες τάσεις τους και πώς, ε, τους, ε, πώς επηρεάζει τον κάθε τομέα η κρίση, καθώς επίσης και ποιες είναι οι κύριες δυσχέρειες που αντιμετωπίζουν οι τομείς αυτοί ή επιπλέον ποιες είναι οι εξελικτικές τάσεις που σημειώνονται ε, και που μπορούμε να υποστηρίξουμε ενδεχομένως και με νέα έρευνα στον τομέα. Υπάρχουν λοιπόν, διαπιστώνουμε ενδιαφέροντα φαινόμενα. Καταρχάς, η έννοια του τομέα έχει όλο και λιγότερο νόημα. Ο τομέας δηλαδή αναπτύσσεται αυτή τη στιγμή όλο και περισσότερο σε ε, συνάφεια με το τελικό προϊόν και ως εκ τούτου η δυσκολία την οποία έχουμε στην αυτοκινητοβιομηχανία Φερρυπίν με τις σημαντικές επιπτώσεις που είχαν εξελίξει αυτό το κλάδο ήταν ότι ήταν ορατές ε, οι δραστηριότητες όχι μόνο στην καθαρή ε, σύλληψη ή ε, κατασκευή ενός αυτοκινήτου αλλά και στη χημική βιομηχανία και σε πολλούς άλλους τομείς και ως εκ τούτου δεν μπορούμε να δούμε τον τομέα αυτόν αποκομμένο. Όταν μιλούμε δηλαδή για αυτοκίνητο βιομηχανία δεν μπορούμε να μιλήσουμε μόνο για έναν τομέα. Το ίδιο ισχύει και για άλλους αντίστοιχους τομείς. Δεύτερον, και αντίθετα από ό,τι γενικά πιστεύετε, ότι δηλαδή η βιομηχανία απασχολεί γενικά χαμηλής εξειδίκευσης εργαζομένους, στην πράξη η βιομηχανία έχει ιδιαίτερα εξελιχθεί ως προς την αξιοποίηση του εργατικού της δυναμικού και κατ' ουσίαν δεν προσδιορίζεται η βιομηχανία από χαμηλής εξειδίκευσης εργαζομένους εργάτες, αλλά από ιδιαίτερης εξειδίκευση εργάτες. Και γιατί, διότι κατά 20% ε, ε, γιατί έχει πέσει κατά 20% η προσφορά ενώ ε, έχει παραμείνει ένα υψηλό ποστό ζήτηση σε θέσει εργασίας και έτσι οι επιχειρήσεις ε, θέλησαν να διατηρήσουν κάποιους καλά εξειδικευμένους εργάτες στην απασχόλησή τους, φοβούμενος ότι σε περίπτωση ανάκαμψης ταχείας δεν θα έχουν επαρκές εργατικό δυναμικό στη θέσή τους για να ενισχύσουν γρήγορα την παραγωγή. Έτσι λοιπόν έχουμε ένα ζήτημα ανθρώπινου δυναμικού εδώ. Και επίσης τρίτον, βλέπουμε ότι δεν έχει νόημα να μιλούμε μόνο για τομείς, αλλά είναι καλό να χαράξουμε ένα τόξο μάλλον, δηλαδή να κάνουμε μια ανάλυση για τρεις-τέσσερις τομείς μαζί, ε, αναζητώντας ποιες είναι οι θετικέ του όψει, ποια είναι τα αρνητικά του, ποια είναι τα κοινά του στοιχεία πάνω απ' όλα. Αυτό είναι κάτι που ήδη κάνουμε εμεί και θα σα δώσω ένα παράδειγμα. Για τα επόμενα 10 χρόνια, Φερρυπίν, οι περισσότεροι, περισσότεροι από του μισού ε, μηχανολόγους που απασχολεί η βιομηχανία θα έχουν βγει στη σύνταξη και μόνο το 1 τέταρτο εξ αυτών θα αντικατασταθούν από τους νέους που τώρα σπουδάζουν και θα έχουν ακολουθήσει τον ίδιο αυτό κλάδο. Δηλαδή θα έχουμε έλλειψη σε υψηλής κατάρτισης ε, προσωπικό και αυτό δεν αφορά μόνο έναν τομέα, αλλά είναι ένα γενικευμένο φαινόμενο. Το ίδιο βλέπουμε και στο θέμα της περιβαλλοντικής νομοθεσίας ή της ε, πολιτικής για την καινοτομία ή για το εμπόριο και προσπαθούμε αυτές τις μεγάλες προκλήσεις ή και ευκαιρίες ίσως να τις ε, αναλύσουμε σε, κατά έναν τρόπο γενικό, να έχουμε δηλαδή μια γενική εικόνα της κατάστασης από την οποία θα μπορούσαμε να ε, παραγάγουμε μια γενική στρατηγική η οποία θα μπορούσε να εφαρμοστεί στον κάθε ένα τομέα χωριστά και έτσι βλέπουμε συγκεκριμένα ε, παραδείγματα μια σύγχρονης βιομηχανικής πολιτικής την οποία εκφράζει η Επιτροπή μέσα από την ανακοίνωσή της Φερρυπίν για το καθαρό αυτοκίνητο, όπου μιλούμε και για την παραγωγή αλλά και για την ε, πολιτική, για τις πρώτες ύλες και για τις επιδόσεις των αυτοκινήτων ή τις αποδόσεις. Αυτά λοιπόν τα εκφράζουμε εμείς μέσα σε στρατηγικές θέσεις με στόχο μια πιο ασφαλή, μια πιο παραγωγική και πιο ε, βιώσιμη θέση εργασίας, ανεξαρτήτως του τομέα ή της επιχείρησης στην οποία ε, απασχολείται ο εργαζόμενος. Όπως είπε και ο εισηγητής σας, είναι για μας αυτές οι κύριες γραμμές, ε, η καινοτομία, η αντιμετώπιση των προκλήσεων της παγκοσμιοποίησης, η αναδιάρθρωση, οι μεταλλαγές στις δομές του μηχανικού κλάδου που πρέπει να αντιμετωπίσουμε διαφορετικά. Ε, κινδυνεύουμε να μας κατηγορήσουν ότι σχολιάζουμε την ιστορία αλλά δεν την συνδιαμορφώνουμε. Ευχαριστώ πολύ για τα σχόλια. Η κυρία Γκροστέτα έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Να, που σήμερα το πρωί έχουμε αυτή την τόσο σημαντική συζήτηση για αυτό το θέμα το οποίο είναι τόσο σημαντικό στην Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί ακόμα περισσότερο σήμερα που βρισκόμαστε σε αυτή την συγκυρία της σημαντικής οικονομικής κρίσης και ήδη έχουμε χάσει έδαφος. Επομένω ε, θα πρέπει να σωθεί ό,τι απομένει για να δούμε πώς θα έχουμε μια σύγχρονη ευρωπαϊκή βιομηχανία. Επομένως, θα πρέπει να μην φανταζόμαστε την ευρωπαϊκή βιομηχανική πολιτική μόνο πάνω στη βάση της πράσινης οικονομίας. Το συζητήσαμε και το ξανασυζητήσαμε και όλοι λέμε ότι θα πρέπει να σωθεί η ευρωπαϊκή οικονομία με καινοτομία, με πράσινη οικονομία, όλα Είμαι πεπισμένη ότι αυτό δεν αρκεί. Γιατί έχουμε μεγάλους τομείς της βιομηχανίας, της κατασκευαστικής, που θα πρέπει να διασώσουν. Πρώτα-πρώτα, κύριε Διευθυντά, θα πρέπει να μας δώσει αυτή την ανακοίνωση Κομισιόν της 13ης Οκτωβρίου. Μας είπε τις βασικές γραμμές της μας είπατε το πλαίσιο στο οποίο κινείστε και μας αναφέρατε ότι η προσέγγιση δεν γίνεται ανατομέα γιατί αυτό θεωρείται τώρα λιγότερο σημαντικό αυτή η αντιμετώπιση. Χρειάζεται οριζόντια, εγκάρσια προσέγγιση. Αλλά δεν μπορούμε να την αποκλείσουμε και αυτήν την τομεακή προσέγγιση. Θα πρέπει να συνέχουμε εμπορική πολιτική, εμπορική ανταγωνισμού, καινοτομία, ε, γνώση, περιβάλλον, καταπολέμηση της ε, ενεργείας, τις μεταφορές και έτσι θα πρέπει να προωθήσουμε την ε, πολιτική μας με το να φροντίσουμε τα δίκτυα, τα μεγάλα δίκτυα και έχουμε εδώ το θέμα της χρηματοδότησης, πολύ βασικό θέμα Τώρα αντιμετωπίζουμε την κρίση, επομένω ε, δεν θα έχουμε νέα χρηματοδότηση, θα πρέπει να την αναζητήσουμε αλλού. Και έχουμε τις ε, συζητήσεις σε σχέση με τον προπολογισμό, τι θα γίνει με τις ε, ενισχύσεις, τι θα γίνει με το πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα. Θα δούμε πώς θα έχουμε κάποιους χρηματοδοτικούς μηχανισμούς. Το μεταλλητήσουμε καλύτερα τους τρεις τρόπους χρηματοδότησης. Κεφάλαιο κινδύνου, ήδη πόροι, εγγύησεις. Εσείς πώς βλέπετε τα θέματα αυτά. Και όταν μιλούμε για τον βιομηχανικό ιστό, μιλούμε για τις ΜΜΕ, δεν είναι μόνο οι μεγάλες βιομηχανίες. Φυσικά έχουμε αυτό, αλλά θα πρέπει οπωσδήποτε να τις υποστηρίξουμε. Η ΜΜΕ είναι το θεμέλιο. Αυτό να δούμε. Πώς θα τις βοηθήσουμε, θα τις υποστηρίξουμε. Να έχουν πρόσβαση στην χρηματοδότηση, στο πρόγραμμα πλαίσιο. Είναι δύσκολα τα πράγματα για αυτές τις και άρα θα πρέπει να δούμε πώς θα τους εγγυηθούμε τη θέση τους, πώς θα τους διευκολύνουμε το έργο. Για τον εξωτερικό ανταγωνισμό πολλές φορές θεωρούμε ότι προχωρούμε σε τραγμένα νερά, χρειάζεται υγιής, αμόλυντος ανώθευτος ο ανταγωνισμός, αυτό θα πρέπει να συνεχιστεί, να μην ε, τίθεται να αμφισβητήσει, να υπάρχει αμοιβιότητα. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχει ανταγωνισμός που να μην χρειάζεται από αμοιβιότητα. Να μην στριμώχνουμε τις δικές μας επιχειρήσεις σε σχέση με τις επιχειρήσεις των τρίτων χωρών. Για πέστε μας, τι συγκεκριμένα μέτρα υπάρχουν, γιατί αυτό που θέλουμε σήμερα δεν είναι ψευδής πόδι, θέλουμε συγκεκριμένα μέτρα, ούτω ώστε να μην μειονεκτούμε στη διεθνή σκηνή. Η Ευρώπη είναι η μόνη περιοχή στον κόσμο που υπάρχει έλεγχος επί των κρατικών ενισχύσεων. Γι' αυτό σας λέω. Τι θα γίνει τόσο ώστε να μην πλήσουμε τις ε, τεχνολογίες, όπως με τους σημειαγωγούς. Βοηθούνται επιχειρήσεις εκτός ένωσης. Όχι εδώ όμως. Γι' αυτό και έχουμε φυγή των επιχειρήσεων, έχουμε στρέβλος του ανταγωνισμού. Τι μέτρα εντάμικ μπορείτε να λάβετε, τι πιστεύετε όσον αφορά την προτυποποίηση. Αυτό το made in. Πώς είναι δυνατόν να προστατεύσουν τον αγωνισμό και να βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις. Έρευνα και καινοτομία. Ας πούμε κάτι πρέπει να γίνει για το διοικητικό άρθρο. Την γραφειοκρατία. Να βοηθήσουμε περισσότερο τα προγράμματα που έχουν σχέση με την επίδειξη. Πράσινες τεχνολογίες. Δεν αρκούν όμως αυτά. Κάτι πρέπει να γίνει να καλυφθεί το χαμένο έδαφος που ε, εκεί που έχουμε μείνει πίσω. Πρόσβαση στις πρώτες ύλες. Μίλησε γι' αυτό ο εισηγητής μας. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Για πολλέ πρώτες πρώτε δεν έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση ίδιου πόρου και όταν υπάρχουν είναι περιορισμένοι. Υπάρχει σπάνια αυτών των πόρων. Άρα τι θα πρέπει να κάνουμε, τι προτείνεται για την έρευνα όσον αφορά την αντικατάσταση αυτών των πρώτων υλών. Γι' αυτό θα πρέπει να επαγρυπνούμε όσον αφορά την εξωτερική πολιτική. Να δούμε τι θα γίνει με την Κίνα, η οποία πάει και εγκαθίσταται ανησυχητικά για μας στην Αφρική. Άρα κάτι θα πρέπει να γίνει ώστε να κερδίσουμε αυτά που χάσαμε, ας πούμε, στην Αφρική. Και βεβαίως να μην παραμελούμε το περιβάλλον, όπως είπε και ο εισηγητής, γιατί χρειάζεται πράσινη βιομηχανία, αλλά θα πρέπει με τρόπο αυτόματο στις αποφάσεις μας την υπόψη τα θέματα του περιβάλλοντος Φερρυπίν να καλύψουμε το θέμα των διαρών του διοξιδίου του άνθρακος. Θέλουμε να μας πείτε κάποιες συγκεκριμένες προτάσεις για να μπορέσουμε τελικά να αναχαιτήσουμε αυτή την κρίση που μας μαστίζει. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση να μην είναι απλά μια ήπειρος υπηρεσιών, αλλά να μπορέσουμε να διασώσουμε τη βιομηχανία μας. Κύριος Χατζημαρκάκης. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχά, θέλω να ευχαριστώ και τον εισηγητή για την πολιτιστική του παρουσίαση, αλλά και τον κύριο Ζωρεκ. Ήταν πολύ ενδιαφέρον και ευφιέ αυτό που μα παρουσιάσατε, κύριε Γενική Διευθυντά, αλλά αυτό περιμέναμε από εσά και περιμένουμε η βιομηχανική πολιτική να ενισχυθεί και πάλι. Όπως είπε ο συνάδελφος Λάγκε, όντω ζούμε σε ένα, βιομηχανό, σε ένα παγκοσμιοποιημένο κόσμο όπου αλλάζουν τα πράγματα και είτε μιλούμε για old economy ή για οτιδήποτε άλλο, πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι χρειάζεται ε, να είμαστε εκείνοι οι οποίοι θα μπορέσουν να τραβήξουν χάρη στη βιομηχανική παραγωγή τους υπόλοιπους που έχουν πέσει, περιέρθει σε κρίση λόγω της χρηματοπιστωτικής τους δραστηριότητας, ε, να τους βγάλουμε λοιπόν από την κρίση. Αυτή θα είναι η μεγάλη δύναμή μας. Εάν μιλήσουμε επίση για τι πρώτε ύλε και τη σχετική πρωτοβουλία, σε σχέση με του Κινέζου, έχουμε 20 χρόνια καθυστέρηση. Εχθέ είδαμε έναν συνάδελφο από το από τη βολή των αντιπροσώπων επικεφαλής ε, μιας μονάδας έρευνας, ο οποίος μίλησε για την πρωτοβουλία πρώτων υλών των ΗΠΑ σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί, διότι διαπιστώνει ότι οι Κινέζοι με τις μεθόδους που ακολουθούν, που βέβαια δεν ακολουθούν τα πρότυπα και τις αρχές της χρηστής ε, διοίκησης, ε, έχουν καπαρώσει όλες τις πρώτες ύλες ανά τον κόσμο. Έχουμε να συζητήσουμε θέματα τα οποία για χρόνια ε, θεωρούνταν ταμπού. Η βιομηχανική πολιτική Φερρυπέν στη Γερμανία δεν συζητούν για χρόνια γιατί λέγανε άμα είναι κάτι που ρυθμίζει αυτόματα η αγορά. Όχι, δεν είναι αλήθεια αυτό. Οι Γάλλοι, όπως ακούσαμε τώρα την κυρία Γκροστέτ να μιλάει, οι Γάλλοι μπορέσαν να φτιάξουν πρωταγωνιστές στη βιομηχανική παραγωγή και όπως και αυτοί θα πρέπει η ολόκληρη Ευρώπη να εξασφαλίσει Ευρωπαίους πρωταγωνιστές. Η Νόκια Φερρυπίν, μια μεγάλη εταιρεία που μπόρεσε να προαγάγει την ευρωπαϊκή βιομηχανική παραγωγή. Χωρίς όμως την μεγάλη πρωτοβουλία της φιλανδικής κυβέρνησης και την υποστήριξη Ευρωπαϊκής Ένωσης τότε που ξεκίνησε αυτή η ιστορία, δεν θα είχε καταστεί δυνατό αυτό. Πρέπει λοιπόν να ενισχύσουμε τους ισχυρούς και τα σημεία που είμαστε πιο δυνατοί. Και δυστυχώς στο παρελθόν η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είχε συνεπή πολιτική φερρυπίν στον τομέα των, της βιομηχανιας που να οι ε, ορισμοί Έχουμε διάφορους τομείς, για να το πω έτσι, με τον τομέα premium όπως ονομάζεται, όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει την πρωτοπορία με 86% της παραγωγής. Και έγινε μία πρόταση, την οποία ευτυχώς παρεμπόδισε το Κοινοβούλιο, η οποία όμως αν είχε περάσει, πρόταση Ευρωπαϊκές Επιτροπές, θα είχε για λόγους αυστηρής και άτεγκτης των αρχών του ανταγωνισμού οδηγεί σε κατάρρευση όλων αυτών των τομέα των premium. Το ίδιο το βλέπουμε τώρα και με τα light vehicles, τα ελαφρά οχήματα. Γι' αυτό λοιπόν παρακαλώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να έχει πιο συνεπή στάση από ό,τι μέχρι τώρα. Ας ακολουθήσει το Κοινοβούλιο. Εγώ προσωπικό συνεργάζομαι με τους αδέλφους από την άκρα αριστερά ακόμη, από την άκρα δεξιά, όταν θεωρώ ότι είναι κάτι θετικό και σκόπιμο για την βιομηχανική πολιτική. Είχαμε στο παρελθόν ε, αν όχι διελκυστίνδα, πάντως διαφορά μεγάλη την οποία ναι, εξέφρασαν ως αντίποδες ο κύριος Δήμας Αφενός και ο κύριος Φερχόγεν από την άλλη. Δεν μπορεί όμως η Επιτροπή να είναι διχασμένη σε αυτό το τομέα. Πρέπει να έχει μια ενιαία και συνεπίσταση. Το ίδιο ε, το ζήτημα το οποίο εσείς θίξατε των μηχανολόγων που θα αναζητούμε σε λίγο πρέπει να το δούμε ως ζήτημα και μεταναστευτικής πολιτικής. Οι ορδές ο κύριος Κόφερ κάνει ένα λογοπαίγνιο εκτός μικροφώνου. Οι ορδές λοιπόν των ε, Κινέζων ε, φοιτητών που βλέπουμε στα μεγάλα μας πανεπιστήμια που σπουδάζουν μηχανολογία κτλ. Αλλά που μετά θα πάνε στην Κίνα και θα τροφοδοτήσουν το εργατικό δυναμικό της Κίνας. Χρειαζόμαστε λοιπόν μια πολύ συγκεκριμένη μεταναστευτική πολιτική. Μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις επίσης που ενδιαφέρουν και την κυρία Γκροστέτ. Εδώ δεν μπορούμε να κάνουμε διαφοροποίηση. Τι θα κάνει μια μικρή επιχείρηση στην αυτοκίνητο-βιομηχανία χωρίς τη μεγάλη αυτοκινητο αυτοκίνητο-βιομηχανική ε, επιχείρηση. Είναι και οι δύο κλάσεις απαραίτητες. Επίσης τα θέματα της ευρεσιτεχνίας. Ας ακολουθήσουμε λίγο το παράδειγμα των Αμερικανών στο ζήτημα της ε, προστασίας της, της βιομηχανικής Το σύστημα first come, first serve, οποίο έρθει πρώτος ε, εφαρμόζει, έχει τα δικαιώματα. Ε, ε, ας δούμε από την άλλη ότι οι Κινέζοι εφαρμόζουν το πιο κλασικό γερμανικό σύστημα αλλά κατά τρόπο πολύ πιο επιθετικό και τελικά ανάμεσα στα δύο αυτά μεγάλα συστήματα εμείς θα συνθλιβούμε σαν να είμαστε ένα φιλαράκι μαρούλι μέσα σε ένα χάμπουργκερ. Γι' αυτό παρακαλώ η Ε, πρέπει λοιπόν να έχουμε μια στρατηγική θεώρηση. Η Επιτροπή πρέπει να έχει μια πιο συνεπή στάση και να προσανατολισόμαστε προς ε, τις τεχνολογίες εκείνες οι οποίες δεν θα, είναι, δεν θα κρυθούν μόνο με γνώμονα την περιβαλλοντική τους αξία, αλλά και την καινοτομία τους και την πρωτοπορία τους στον τομέα της χημικής βιομηχανίας. Πολλά πράγματα κινδυνεύουν τα τελευταία χρόνια λόγω των επιλογών μας λόγω επιλογών που σημαίνει ότι η βιομηχανία δεν θα μπορεί να, κάνει, να αξιοποιήσει κάποιες εφαρμογές. Ευχαριστώ πολύ. 15 λεπτά ακόμη. Για να ξεκινήσουμε ακριβώς τις 10 τις ψηφοφορίες. Έχω όμως 12 ε, συναδέλφους που έχουν στήσει το λόγο μπορούμε να διαλέξουμε. Είτε μιλάτε ως καθένας όσο θέλετε, και τότε μιλούν μόνο οι δυο τρει πρώτοι, είτε μιλάνε όλοι, αλλά από ένα λεπτό ο καθένας. Η κυρία Τσικά. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Η βιομηχανική πολιτική πρέπει όντως ε, να ληφθεί σοβαρά υπόψη, γιατί 80% της, των θέσεων εργασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση τις εξασφαλίζει βιομηχανική πολιτική. Δηλαδή βιομηχανική πολιτική σημαίνει και μέλλον τη Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και από τις τελευταίες μα στατιστικές βλέπουμε ότι στον χώρο της ε, αυτοκινητοβιομηχανίας έχουμε τα μεγαλύτερα ποσοστά. 30, 75% ε, εκεί, 30% ε, στα χημικά προϊόντα, ένα άλλο 15% στην μηχανουργία επίσης στη μεγάλη βιομηχανία, αεροπλάνα κτλ. και φαρμακευτική βιομηχανία. Αυτές είναι, αυτοί είναι οι συσχετισμοί σε παγκόσμιο επίπεδο και ε, εκεί που έχουμε την πρωτοπορία ακριβώς θα πρέπει να ε, προχωρήσουμε σε μέτρα τα οποία θα μας επιτρέψουν να την διαφυλάξουμε. Υπάρχουν λοιπόν και βιομηχανία, υπάρχουν και δεξιότητες και εξειδίκευση στα κράτη-μέλη και πιστεύω αυτά θα πρέπει να τα θέσουμε στο επίκεντρο των προσπαθειών μας και να αναζωογονήσουμε τους τομείς αυτούς. Ο κλάδος TIC επίσης είναι πολύ σημαντικό. Χωρί αυτόν δεν μπορούμε να πούμε. Κυρία Τρότμαν, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να θέσω ένα ερώτημα προ τον κύριο Διευθυντή. Όταν πήγαμε σε μία αποστολή στην Ισπανία, στην Ισπανική Προεδρία, συναντήσαμε πήγαμε στο Joint Research Center στη Σεβίλη και μας είπαν ότι ζητήθηκε μία μελέτη για μία βιομηχανία που θα δημιουργούσε απασχόληση. Το θέμα των πράσινων θέσεων απασχόλησης είναι βασικό θέμα. Η βιομηχανία θα πρέπει να συμβάλλει τα μάλα στη διατήρηση και δημιουργία της απασχόλησης. Το είπατε όσον αφορά μηχανικούς, αλλά υπάρχουν και άλλες θέσεις εργασίας, όχι μόνο αυτές που αποτελούν, α, απαιτούν υψηλές ε, γνώσεις υψηλού επίπεδου. Ε, πώς θα καταλήξουν αυτή τη λύση, τι συμπεράσματα έχετε συνάγει. Τώρα όσον αφορά το άλλο θέμα, σε κάποιες περιπτώσεις όσον αφορά τα συστήματα που χρησιμοποιούνται, τα TIC κλπ, έχουμε κάποια κενά όσον αφορά τις αξίες που επιδιώκουμε. Έχουμε ένα πρόγραμμα πλαίσιο, ε, το ΙΝΤΕΡ, και μικρά προγράμματα έρευνας. Στα πλαίσια των αυξήσεων των κονδυλίων του παρόντος προγράμματος πλαισίου θα μπορούσατε να επιλέξετε τα κενά να δημιουργηθούν ομάδες έρευνας εκεί. Και για να μην εισάγουμε τεχνολογία. Μα απειλεί με το σφυράκι ο Πρόεδρος, αλλά θα ήθελα να πω δύο μικρά πραγματάκια. Πρώτα απ' όλα όσον αφορά την Τράπεζα Επενδύσεων, χρειάζονται να υπάρχουν οτοστατικά προϊόντα που να παρακινούν στην ε, ε, δραστηριοποίηση και όσον αφορά την ε, ευφυή προσέγγιση για τα οικονομικά, Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να δημιουργήσει κατάλληλα εργαλεία. Είναι αδύνατο να προχωρήσουμε αφελώ έναντι των εξωτερικών ανταγωνιστών μας. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πραγματικά αυτό που μας είπε και ο κύριος Ζούρε και ο εισηγητής είναι πολύ σημαντικά και είπαν όσα πρέπει κανείς να καλύψουμε μια τέτοια έκθεση. Όμως, ακόμα υπάρχει ένα άλλο θέμα. Θα πρέπει να καλύψουμε την πολιτιστική βιομηχανία ή τις πολιτιστικές βιομηχανίες, γιατί η συνεισφορά τους είναι σημαντική στο ΑΕΠ. Πρόκειται για ένα κλάδο που είναι διτός, γιατί μετέχει και του πολιτισμού και της βιομηχανίας. Άρα θα πρέπει να προβληματιστούμε πώς και τι θα κάνουμε για αυτό τον ε, τομέα. Είναι ένας κλάδος που τον έχει χτυπήσει λιγότερο τώρα η κρίση, αλλά θα πρέπει να δούμε και σε αυτή την περίπτωση τι θα κάνουμε για την καινοτομία που επιβάλλεται. Κύριε Αγγέλεκ. Κύριος. Ευχαριστώ. Είναι πολύ φιλόδοξο το θέμα και τον ζηλεύω τον κύριο Λάγκε για τη δουλειά που έκανε και κάνει. Νομίζω ότι το βασικό θέμα και το βασικό ερώτημα που πρέπει να θέσουμε είναι το εξή. Ποιο είναι το μήνυμα που βγαίνει από αυτή την έκθεση, από αυτή τη δουλειά. Μια έκθεση αναλυτικότατη. Τι θέλουμε να κάνουμε, ποια είναι η βασική θέση Ποιο είναι το βασικό μήνυμα που θέλουμε να στείλουμε, διότι εγώ βλέπω δύο τοποθετήσεις. Η μία είναι πιο παθητική, δηλαδή να προσαρμοστεί η βιομηχανική πολιτική στην βιομηχανοποίηση, αυτή είναι η πρώτη φάση. Και εδώ ο βασικός παράγοντας που απορρέει από τον παγκόσμιο ανταγωνισμό που ξεκίνησε από το ελεύθερο εμπόριο και όχι σύμφωνα με θεμητό, κανόνες θεμητό ανταγωνισμού είναι ο πρώτος παράγοντας. Η Ευρώπη, εάν θέλει να ακολουθήσει τους άλλους, θα πρέπει να έχει χρόνο και θα πρέπει επίσης να μπορεί να προστατεύσει την ευρωπαϊκή αγορά. Αυτό είναι το μήνυμα που απορρέει από την πρώτη τοποθέτηση, την παθητική της έκθεσης. Η δεύτερη είναι ενεργητική τοποθέτηση, να δημιουργηθεί νέα βιομηχανική πολιτική μέσω ενός νέου μοντέλου κατανάλωσης. Πρέπει να βρεθούν νέες λύσεις, ε, υπολογιστές, πληροφορική, αυτό είναι σημαντικό και μετά η μελλοντική πόρη και αυτό είναι σημαντικό πολλά εξαρτώνται από τη μηχανολογία υλικών και από τις πράσινες τεχνολογίες που θα πρέπει να ερμηνευθούν σωστά. Ποιες είναι οι πράσινες τεχνολογίες. Κύριος Ρούμπιχ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ιδιαίτερα και στην περίοδο της παγκόσμιας αύξησης της δημοκρασίας η βιομηχανική πολιτική έχει μεγάλη σημασία γιατί θα μας απασχολήσει και το ζήτημα του πώς θα γίνονται οι ε, πληστηριασμοί των εκπομπών στο μέλλον. Σε σχέση λοιπόν με το θέμα αυτό και με τις προτάσεις της Επιτρόπου για φορολόγηση των προϊόντων με φόρο διοξιδίου του, του άνθρακα, μήπως θα ήταν σκόπιμο να ε, προτείνει η Επίτροπος να επιβαρυνθούν με ένα ποσοστό φορολόγηση τα προϊόντα τα οποία έχουν υψηλές, ε, υψηλή συμβολή στις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Ίσως όμως είναι η ώρα και ε, στο Συμβούλιο των Υπουργών Οικονομικών να συμμετάσχουν να συμμετέχουν οι αρμόδιοι για τα θέματα της βιομηχανίας έτσι ώστε να προσδιορίσουμε συγκεκριμένους στόχους για τη βιομηχανία μας από το 2020, συμμετοχή στην οικονομία μας, της βιομηχανίας κατά 20% και όχι μόνο των τραπεζών. Ευχαριστώ κύριο Σοντή. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ο πλανήτης τα πάει καλά. Η Κίνα αναπτύσσεται στους σωστούς ρυθμούς, η Αφρική αναπτύσσεται, όλα πάνε καλά εκτός από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και πιθανότατα η ενδεδειγμένη βιομηχανική πολιτική είναι από τα κλειδιά της ανάπτυξης που περιμένουμε όλοι. Έχω την εντύπωση και γενική διευθυντά ότι πρέπει να κολλήσουμε να εξετάσουμε σημείο. Αλλάζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εσείς μένετε, ίσως να έχετε ένα όραμα που είναι ενδιαφέρον. Το βασικό, το ισχυρό σημείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η ανταγωνιστικότητα, είναι το κλειδί της επιτυχίας. Και έχουμε δύο να στον την ανταγωνιστικότητα, κοινωνικές προδιαγραφές, έχουμε παράδοση ρυθμίσεων κοινωνικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ένα νέο στοιχείο που είναι η νομοθετικ... περιβαλλοντική νομοθεσία. Είναι, βοηθά την ανταγωνιστικότητα η κοινωνική νομοθεσία ή όχι. Διότι τώρα θεωρούσαμε ότι είναι υπέρ του ανταγωνισμού και όσον αφορά το περιβάλλον, ε, όσον αφορά τον άνθρακα, την νομοθεσία των άνθρακα, τι πιστεύετε, τι σημασία έχει αυτό αν δεν υπάρχει συμφωνία σε παγκόσμιο επίπεδο και όσον αφορά την εμπορική πολιτική μας είμαστε αφελείς και ας είμαστε πολύ απαιτητικοί όσον αφορά την αμοιβαιότητα έναντι των άλλων στον κόσμο, των άλλων εμπορικών φορέων στον κόσμο. Κύριος Χάναχαν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, ναι, α, δώστε μου και εμένα 12 λεπτά για να πω όλο αυτό το θέλω να πω, γιατί πάντα οι ίδιοι μιλάνε ένα, ένα λεπτό και υπάρχουν άλλοι που μιλάνε 12 λεπτά, γιατί αυτό το οποίο θέλουμε είναι να έχουμε την εποχή της παγκοσμιοποίησης μια βιομηχανική πολιτική, αλλά το πρόβλημα είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει μια βιομηχανική πολιτική και αυτό το οποίο άκουσα από του επιτρόπους εδώ, τους διαφορετικούς επιτρόπους, ότι δεν υπάρχει βιομηχανική πολιτική κοινή στην Ευρώπη, διότι Μόνο η αγορά θα πρέπει να αποφασίζει ποιος θα ζήσει και ποιος θα πεθάνει. Ε, από εκεί και πέρα υπάρχει θέμα ουσίας, γιατί αν δεν υπάρχει κοινή βιομηχανική πολιτική, πώς είναι δυνατόν να υπάρχει βιομηχανική πολιτική την εποχή της παγκοσμιοποίησης. Άρα θα πρέπει να αρχίσουμε από το Α. Η χρησιμότητα της βιομηχανίας στην Ευρώπη, η χρησιμότητα της βιομηχανίας για τον Ευρωπαίο. Τι κάνει η βιομηχανία όσον αφορά τους πόρους για το σύνολο της Επίρου. Τρία ερωτήματα. Αν δεν υπάρχει κοινή πολιτική και αποφασίζουν οι αγορές, τι θα κάνουμε. Δεύτερη ερώτηση. Πώς θα... Ε, τι θα κάνουμε για το ότι το, το, το, κέρδος είναι το μόνο κίνητρο. τρίτον, τι θα γίνει με την αποβιομηχάνηση στην Ευρώπη αφού δεν μπορούμε να έχουμε κάποιους κανόνες που να απαγορεύουν το, το ντάμικ, το κοινωνικό, το φορολογικό, το περιβαλλοντικό. Ευχαριστώ κύριε Χινάν τις ε, παρατηρήσεις σα για το χρόνο ομιλίας. Αλλά σα πω το εξή. Αυτοί μπορούσαν να μιλήσουν περισσότερο χρόνο, ήταν ο εισηγητή, οι δύο σκιώδει εισηγητέ και η Επιτροπή. Ναι. Προσπαθώ κατά τα άλλα να περιορίσω το χρόνο. Ο κύριο Βέμπερ έχει το λόγο. Βέμπερ, νομίζω ότι υποσχέται πολλά η έκθεση Λάγκε που είπε πολλά. Εγώ σε ένα λεπτό μόνο θα ένα, ένα πραγματάκι θέλω να θίξω ότι Εμεί δεν είναι δυνατόν να κάνουμε τίποτα όσον αφορά το θέμα της προστασίας. Διότι όλες οι μεγάλες εταιρείες, οι μεγάλες κοινωνίες και οι πιο ανοιχτές προστατεύονται. Οι προθελητές οι ε, συναλλαγές και ανταλλαγές είναι ύπαλο και αυτοί προστατεύονται. Επομένως τι θα γίνει κόντρα στον ντάμπινγκ, κόντρα στον αθήντο ανταγωνισμό και η Γερμανία το ίδιο και με, με, με αυτούς τους τεχνικούς κανόνες, μην πούμε για την, ε, για την Κίνα, κάθε είδους ντάμπινγκ ε, κάνει και ταυτόχρονα προστατεύεται. Τι θα γίνει με το χρηματοοικονομικό ντάμπινγκ. Ε, κυνηγάει τις ενισχύσεις η, Ένωση, ενώ η Κίνα κάνει ό,τι μπορεί και, και είπα. Ε, κόστος μηδέν για αυτούς. Ε, επομένως, εμείς τίποτα. Εγώ είμαι κατά του προστατευτισμού ως ε, δόγμα, ως αναρρίπλωση Είδαμε τι έγινε το, δεκαετία του 30 και σήμερα το ακόμα χειρότερα. Επίση είμαι κάθετα κατά του να είναι κανεί αθώο, σαν Άγγελο και, και, και Θα πρέπει κανεί να προστατεύεται κατά την τάμη και δεν το κάνει αυτό η Ευρώπη. Υπάρχουν ε, προστασίες θεμητέ. Να το κάνουμε όπω οι Αμερικάνοι. Έχουν ένα σωρό οι Αμερικάνοι και εμεί τίποτα. Ευχαριστούμε πολύ. Μπιτικόφερ. Ο κύριος Μπιτικόφερ. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ο αντιπρόεδρο Ταλιάνη, που ασχολείται με τη μηχανική πολιτική, μίλησε για μια fresh approach, καινούρια προσέγγιση και είμαι πεπισμένο ότι όπως και να έχει χρειαζόμαστε τουλάχιστον αυτή τη νέα προσέγγιση. Δεν μπορούμε να λέμε business as usual, δεν μπορούμε απλώς να ε, ξανά επαναλαμβάνουμε παλές προσεγγίσεις. Χρειάζεται με δεδομένη την παγκοσμιοποίηση να αναπτύξουμε μια ευρωπαϊκή βιομηχανική πολιτική φιλόδοξη όσο δεν την έχουμε δει ποτέ. Βιομηχανική πολιτική δεν σημαίνει ευρωπαϊκός, κεντρικός, κρατικός παρεμβατισμός. Χρειάζεται μια πραγματικά στοχευμένη βιομηχανική πολιτική που θα είναι και διατεθειμένη να στηρίξει τη βιομηχανία αλλά και να αγωνιστεί κατά του ντάμπινγκ. Βιομηχανική πολιτική σημαίνει ταυτόχρονα ότι η Ευρώπη δεν θα προσδιορίζει τις βιομηχανικές της επιλογές μόνο ε, με βάση τα εμπορικά κριτήρια, γιατί εκεί έχει πιο πολλές αρμοδιότητες, αλλά με βάση τις αρχές που είναι οι αρχές της νέας εποχής στην οποία ζούμε. Αυτές, αυτές τις αρχές περιέγραψε ο Τόμας Φρίντμαν στους New York Times λέγοντας ότι αυτός ο οποίος θα μπορέσει να έχει την τεχνολογία, την πράσινη τεχνολογία και την καινοτομία στον 21ο αιώνα θα είναι εκείνος που θα έχει τη διαφορά στήθους για να προχωρήσει στο μέλλον. Κύριε Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να θέσω δύο ερωτήσεις σύντομες. Πρώτον, ποια βιομηχανία θέλουμε να έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ποια είναι η επιθυμία μας, τι ρόλο θα παίξουν οι χώρες μας στο βιομηχανικό τομέα, ε, αυτή, για το παρόν και για το μέλλον. Αυτές είναι οι δύο ερωτήσει μου. Η χώρα μου έχει απίστευτο αριθμό μετεγκαταστάσεων επιχειρήσεων. Γίνονται ε, ομαδικές απολύσεις, πλήττονται εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενοι, διότι οι βιομηχανίες εγκαταλείπουν την ε, Πορτογαλία και πάνε σε άλλες χώρες. Στην Ασία, στη Βόρεια Αφρική. Εξαφανίζεται η βιομηχανία que eram tradicionais, como a Εξαφανίζονται όχι μόνο από τον παραδοσιακό τομέα όπως είναι η Φαντουργιά και τα υποδήματα, αλλά και η αυτοκινητοβιομηχανία. Ο ηλεκτρικός, ηλεκτρονικός εξοπλισμός. Από πολλούς ποικίλου τομείς, καθώς και από τομείς ε, εχμής. Ε, νομίζω ότι δεν υπάρχει στατική συγκεκριμένη σήμερα. Πώς θα καταπολεμήσουμε λοιπόν το φαινόμενο, πώς θα υπάρξει η βιομηχανική πολιτική που θα προστατεύσει τη βιομηχανία και την απασχόληση στην Ευρώπη. Καλό ήρθα, να θα ήταν για να κλείσουμε λίγο ο Πρόεδρο να δώσω το λόγο στον ε, κύριο Γενικό Διευθυντή, τον κύριο Τσούρεκ, παρακαλώ, να δώσει απαντήσει του. Και παρακαλώ του συναδέλφου να είναι προσεκτικοί και ήσυχοι. Ευχαριστώ πολύ. Σημειώνω από τα όσα είπατε ότι είναι ένα θέμα στο οποίο έχετε ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Σημειώνω επίσης ότι η βιομηχανική πολιτική είναι μόνο μία από τις δραστηριότητες μας, ε, γιατί ακούστηκε και η καινοτομία και άλλοι τομείς δράσης που θα πρέπει να δώσουμε έμφαση. Εγώ θα κάνω την πρόταση. Οι συνεργάτες μου που έχουν έρθει εδώ, ε, κυρία Διπλέμου και ο κύριος Μπέρκμαν, να ε, έρθουν σε επαφή διμερώς μαζί σας μετά την ψηφοφορία σας είναι στη θεσή σας εδώ για να σημειώσουν συγκεκριμένες παρατηρήσεις έτσι ώστε να έχουμε και συντομία χρόνου βέβαια και πιο αποτελεσματική συνεργασία. Ο Πρόεδρος, Καλώ οι συνάδελφοι που έχουν συγκεκριμένε ερωτήσει για την Επιτροπή μετά την ψηφοφορία παρακαλώ να έχουν υπόψη τους ότι η Επιτροπή είναι στη διάθεσή τους για να δώσουν απαντήσεις. Νομίζω ότι είναι πολύ καλή και πρακτική αυτή η συζήτηση. Ευχαριστώ Ολοκληρώνεται το σημείο αυτό για σήμερα. Και περνούμε στις ψηφοφορίες, αγαπητοί συνάδελφοι.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 συγκεντρωθούμε λίγο. Έχουμε αρκετές φοφορίες όχι πολλές, αλλά αρκετές σήμερα. Και σας παρακαλώ να ξεκινήσουμε με την πρώτη, το μέλλον της ευρωπαϊκής τυποποίησης και να δώσω το λόγο σύντομα στον κύριο Μπίτικόφερ. Χάρη στη βοήθειά του μπορέσαμε να κερδίσουμε χρόνο. Δεν έγινε κι άλλη συζήτηση σήμερα, αλλά πάντως το λόγο πρέπει να τον δώσω σήμερα. Κύριε Μπιτικόφερ. δεν θέλω να ευχαριστώ τον συνάδελφο Κοσούσνικ, που είναι επίσης εισηγητής από πλευράς της Επιτροπής ΙΜΚΟ, ε, συντάχτης νομοδότησης. Τον ευχαριστώ, έχει έρθει και εκείνο σήμερα εδώ. Και θα ήθελα επίσης να επισημάνω ότι στην έντυπη μορφή του η συμβαστική τροπολογία υπαριθμών 4 το κείμενο δεν είναι πλέον επίκαιρο, διότι εχθές ετοιμάσαμε μια νέα διατύπωση την οποία στην οποία συμφώνησαν οι ομάδες και παρακαλώ τους συναδέλφους ε, που ενδεχομένως έχουν διαβάσει την γραπτή μορφή να μην ενοχληθούν. Θα σας διαβάσω όταν έρθει η ώρα την ε, νέα μορφή της ευαστική τροπολογίας. Και ο κύριος και ε, αν δεν έχουν αντίρρηση οι συνάδελφοι, μπορεί να λάβει το λόγο για ένα λεπτό πολύ σύντομα. Είστε εδώ. Ε, ευχαριστώ Πρόεδρε. Δεν θέλω να κάνω μεγάλες συζητήσεις. Απλώς θέλω ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο εισηγητή, τον κύριο Μπιτικόφερ. Ήταν πολύ καλή η συνεργασία. Και περιμένουμε να δούμε τα δικά σας αποτελέσματα, αποτελέσματα της δικής σας ψηφοφορίας και εμείς από την ΕΜΚΟ θα καταθέσουμε τις δικές μας τροπολογίες φυσικά στην γνωμοδότηση. Με τη γνωμοδότηση ε, για το μέλλον της ευρωπαϊκής τυποποίησης πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε εκ της βάσεως προς τα άνω τη διαμόρφωση της, των, της τυποποίησης και των προδιαγραφών. Αυτό θα μας εξασφαλίσει καλύτερη ανταγωνιστικότητα ασφαλώς. Ο Πρόεδρος Καλός, περνούμε στην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 κατά εποχές Εγκρίνεται συμβαστική 4. Ο κύριος Κόφερ. Α, όχι, συγγνώμη, λέει ο πρόεδρος. 24, τροπολογία 24 της κυρίας Τσικά. Υπέρ. Κυρία Τσικάου παίρνει το λόγο. Πρόεδρε. Μια προφορική τροπολογία, αν μου επιτρέπετε, στην 24. In global competition. Θέλω να συμπληρωθεί στο κείμενο η φράση in global competition στον παγκόσμιο ανταγωνισμό. Καλώ λέει ο πρόεδρο. 24 με προφορική τροπολογία. Την ψηφίζουμε υπέρ. Κατά. Αποχές. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 4, κύριε Μπιτικόφερ, εσείς. Ναι, Πρόεδρε, θα ήθελα να σας διαβάσω το κείμενο για το οποίο θα ψηφίσουμε τώρα ζητεί κάθε μία από τις εμπλεκόμενες οργανώσεις να λάβουν το ρόλο που, τους που τις αρμόζει στη διαδικασία τυποποίησης και να τους δοθούν οι εξουσίες για τη συνδιαμόρφωση των ευρωπαϊκών προδιαγραφών στις οποίες έχουν ήδη συμβάλει για... Ε, και ζητού... ζητεί μία διαδικασία επίλυση διαφορών ταχεία έτσι ώστε να επιλύονται ε, γρήγορα οι διαφορέ ως προς την τήρηση των προδιαγραφών. Καλώ λέει ο Αυτή είναι συμβαστική 4 με τη ορθωμένη τη μορφή υπέρ κατά αποχέ, εγκρίνεται. Και τώρα μου λένε ότι όλες οι λοιπέ τροπολογίες πλην 2 μπορούν να ψηφιστούν συνολικά, εκτός από την 40 και τη 42. Συμφωνούν, ναι. Λοιπόν, τώρα, καταπληκτική η πρόταση, και με μεγάλο ενθουσιασμό προτείνω πλην τις 40 και 42 να ψηφίσουμε όλες τις λοιπές τροπολογίες μαζί. Υπέρ παρακαλώ. Ευχαριστώ κατά. Αποχές εγκρίνονται και έτσι μας μένουν η συμβαστική 5 Άλλη μια επιπλέον ε, ψηφοφορία. Η 5 συμβαστική. Ευχαριστώ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 40 Τροπολογία 40, χωριστά, υπέρ, κατά. Αποχές. Εγκρίνεται και 52, λέει ο πρόεδρος. 52, υπέρ, κατά. Αποχές. Εγκρίνεται και συμβαστική 6, παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία. Με το ηλεκτρονικό μας σύστημα άρχεται η ψηφοφορία. Ε, περισσεύουν τέσσερις από το ΕΛΚ. Δεν ξέρω πώς καταφέρετε να τους πολλαπλασιάσετε έτσι. Ρυθμίστε το. Πέρασε ψηφοφορία. Εντάξει τώρα. Δεν είμαι απαραίτητα κατά βέβαια τη συμμετοχή του, αλλά πα περιπτώσει. Λοιπόν, πέρα τη ψηφοφορία. Να επαναλάβουμε παρακαλώ γιατί έγινε ένα ασφάλμα από εδώ. Επαναλαμβάνουμε την ψηφοφορία για άλλη μια φορά. Η τελική ψηφοφορία, ψηφο ηλεκτρονική. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Και το αποτέλεσμα είναι σαφές. Mm. Συγχαρητήρια, σαφές το αποτέλεσμα για τον εισηγητή. Και ενώ ω πρόεδρο δεν πρέπει να κάνω τέτοιου είδου σχόλια, πρέπει να σα πω ότι μου άρεσε πάρα πολύ η κατάρτιση του καταλόγου των ψηφοφοριών. Πολύ με βόλεψε και θα ήθελα να το παραλαμβάνουμε για άλλε φορέ. Και τώρα πάμε σε μια εύκολη επίση ψηφοφορία, την ολοκλήρωση, την τελική μάλλον ψηφοφορία, για τη ρύθμιση, ε, την ασφάλεια εφοδιασμού με αέριο και ρωτώ ποιος είναι υπέρ της προτάσεως. Α, ηλεκτρονικά κατευθείαν καλύτερα. Ηλεκτρονική ψηφοφορία παρακαλώ. Άρχεται ψηφοφορία. Ένας σοσιαλιστής περισσεύει. Και? Α, και ένας από το ΕΛΚ, μάλιστα. Ξέρετε τι πρέπει να κάνετε. Πέρα στις ψηφοφορίες. Το αποτέλεσμα είναι σαφές. Σας ευχαριστώ πολύ. Και αυτές ήταν οι ψηφοφορίες μας. Ευχαριστώ πολύ. Και έτσι μπορούμε να προχωρήσουμε στο σημείο 13 της της διάταξης. Και μια και Κάποιοι εκ των συναδέλφων συνήθω αποχωρούν από την αίθουσα μετά τι ψηφοφορίε. Σα παρακαλώ να είστε στο δυνατόν πιο διακριτικοί και ήσυχοι για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε απρόσκοπτα τη συζήτησή μα. Έχουμε μια πληθώρα σχεδίων να συζητήσουμε. Και αν μας επιτρέπετε, περνούμε στο σημείο 13, απλούστευση της εφαρμογής των προγραμμάτων πλαισίου έρευνας. Αγαπητοί συνάδελφοί, σας παρακαλώ να είστε όσο το δυνατόν ήσυχοι και διακριτικοί για να μπορέσουμε να ακούσουμε τη συνάδελφο Καρβάλιο που θα λάβει το λόγο. Παρακαλώ, επιτρέψτε μας να ξεκινήσουμε τη δουλειά μας. Hans, αποχωρήστε ησύχως.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 Έχουμε ακόμα κάποια θεματάκια στην ημερήσια διάταξη, γι' αυτό καλό είναι να συγκεντρωθούμε και να προχωρήσουμε στη δουλειά μας. Η κυρία Καβάλιο παρακαλώ. Έχετε το λόγο. President, ladies and gentlemen, good morning. Κύριε Κυρία Καρβάλιο, καλημέρα σας για να ξεκινήσουμε. Να σας τονίσουμε ότι έγινε μια ευρύτατη διαβούλευση για αυτή την έκθεση. Τη... Ξεκίνησε τη διαδικασία και ήταν η ανταπόκριση πληθωρική. Σας ευχαριστώ όλους. The, report is of real interest to the... Πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η έκθεση αυτή και επίσης ε, ήρθε την ε, κέρια στιγμή, γιατί ήρθε η ώρα της αξιολόγησης του 7 προγράμματος για να προπαρασκευαστούμε για το επόμενο. Έχουμε τέσσερις πτυχές της έκθεσης που θα πρέπει να τις τονίσουμε. Πρώτα-πρώτα, διοικητική απλούστευση, βελτίωση σε προσβασιμότητα, διαφάνεια και ποιότητα. Επίσης, θα πρέπει να σας τονίσω ότι θα πρέπει να υπάρχει περισσότερη συνέργεια για τα μέσα και όργανα και εργαλεία πολιτικής που ε, χρησιμοποιούμε τώρα. Θα πρέπει να προετοιμαστούμε για το 8ο πλαίσιο και θα πρέπει επίσης να δούμε πώς θα έχουμε περισσότερη απλούστευση. Και εδώ έχουμε δύο πτυχές που φαίνονται από την έκθεση. Γενικές αρχές και συγκεκριμένες συστάσεις. για τις γενικές αρχές. Τονίζω ότι η απλούστευση ωφελεί όλους τους εμπλεκόμενους. Γιατί θα πρέπει να έχουμε σταθερότητα και ασφάλεια δικαίου. Ευέλικτη προσέγγιση χωρίς όμως να έχουμε μια διαδικασία μη στεγανή που θέτει την κινδύνο το δημόσιο χρήμα. Άρα θα πρέπει οι επιλέξιμοι να εφαρμόζουν τις κείμενες συνήθεις αρχές και διατάξεις. Για τις συστάσεις, ο σωστός είναι να έχουμε περισσότερη ασφάλεια και σαφήνεια. Αυτό τι σημαίνει. Να ξεκαθαριστεί το τι πρέπει να αλλάξει, πώς θα αλλάξει, πότε και με τι ρυθμό. οι διατάξει να προστευτούν όσον αφορά την ε, χρηματοδότηση και την σχετική μεθοδολογία. Μέθοδοι υπολογισμού θα είναι οι ίδιες για το κάθε εργαλείο πολιτικής ή όχι. Επίσης τελικά θα πρέπει να έχουμε σαφήνεια όσον αφορά τους ορισμούς, όσον αφορά επίσης τα εφάπαξ ποσά, τα, τα κατά αποκοπή ποσά, τους επιλέξιμους γιατί θα πρέπει να υπάρχει συνέπεια στην εφαρμογή των νομοθετημάτων για όλους και όλες τις διαδικασίες. Ποιότητα, διαφάνεια και προσβασιμότητα τώρα. Εδώ τονίζω τρία τεινά. Γενικώ είμαι υπέρ του να υπάρχει μία επιστημονική προσέγγιση αριστεία και ταυτόχρονα οικονομικός έλεγχος. Έχουμε επίσης την προσέγγιση βάσει των αποτελεσμάτων που έχει προτείνει η Επιτροπή. Υπάρχουν εδώ κάποια πλεονεκτήματα. Όμως, αυτή η προσέγγιση θα πρέπει να έπεται κάποιας πιλωτικής δοκιμής για να μπορούμε να διαπιστώσουμε τι ορισμός θα επικρατήσει όσον αφορά την έννοια του αποτελέσματος για επίδειξη και τεχνολογία, τέτοια προγράμματα. Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις συγκεκριμένων προκλήσεων επίσης προτείνω να υπάρχουν κάποια βραδεία. Αυτό που τα προτείνει και η Επιτροπή για περιπτώσεις όπως το Συμβούλιο Έρευνας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό τα κράτη-μέλη να συνεχίσουν έχουν την αρμοδιότητα του ελέγχου. Κυρίως όσον αφορά ασφάλεια και άμυνα και σε κάθε περίπτωση που υπάρχουν κάποια προγράμματα που έχουν τέτοιου είδους επιπτώσεις να υπάρχει διαδικασία δύο σταδίων και αυτό να οδηγεί σε μια πιο αποτελεσματική προετοιμασία και συνέχιση του έργου. Αυτά πάνω σε μια πλατφόρμα ευελιξίας. Και αυτό να ισχύει για όλες τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Συνέργεια θέλουμε για τα προγράμματα και για τα μέσα πολιτικής και να μειωθεί η πολυπλοκότητά τους. Άρα να έχουμε ενιαία ερμηνεία και εφαρμογή κανόνων και διαδικασιών. Εναρμόνιση για όλα τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τέλος, Όσον αφορά το επόμενο πρόγραμμα πλαίσιο, σας τονίζω τα εξής τρία. Διοικητική απλούστευση. Αυτό θα πρέπει να είναι η προτεραιότητα για το 8ο πρόγραμμα. Να μειωθούν τα εργαλεία πολιτικής και πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερο συντονισμός. Το 8ο πρόγραμμα πλαίσιο θα πρέπει να λάβει υπόψη κάθε περίπτωση καινοτομία, ε, έρευνα μεθοριακή, αξιοποίηση των αποτελεσμάτων και ταχύτερη ένταξη των αποτελεσμάτων στην αγορά. Και έτσι να πρέπει να, να μπορούμε να φτάσουμε σε ισορροπία της έρευνας είτε, είτε υπάρχει μέθοδος από πάνω προς τα κάτω είτε το αντίστροφο. εσωτερήκευση του κόστους για το 8ο πρόγραμμα πλαίσιο και αυτό επίσης να καλύπτει και τις αναπτυσσόμενες χώρες. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Καρβάιου. 12 συνάδελφοι έχουν ζητήσει το λόγο. Έχουμε και άλλα σημεία στην ημερήσια διάταξη. 13 έχουμε τώρα που έχουν ζητήσει το λόγο. Οπότε θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ σύντομοι. Καταρχάς θα ήθελα να δώσω το λόγο στους, στο σκιώδη εισηγητή και μετά στους άλλους. Παρακαλώ ε, να, να θυμηθείτε αυτοί που παίρνετε το λόγο πρώτοι και τελευταίοι θα έπρεπε να μπορούν να μιλήσουν. Η κυρία Ρία Ραμαδουρέλ πρώτα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όπως πάρα πολύ καλά μας τα εξήγησε η συγγήτρια, από το 1984 έχουμε διάφορα προγράμματα πλαίσια τα οποία έχουν εξελιχθεί και προχωρήσει σημαντικά και ε, αυξήθηκε και η προκοδότησή τους, έχουν ε, αυξηθεί οι τομείς που καλύπτονται και μιλούμε τώρα για το ότι τώρα θέλουμε να έχουμε κάποια πρόοδο χωρίς τους κινδύνους που συνεπάγονται τέτοια ανοίγματα. Πάντως να συγχαρώ την συντάκτρια της έκθεσης. Νομίζω ότι εξάντλησε το θέμα, είναι τέλεια η έκθεσή της όσον αφορά το τι ζητά η κοινότητα των επιστημόνων, το τι ζητάμε εμείς, για το τι κατευθύνσεις θα πρέπει να ακολουθήσουμε Έχουμε επίσης και το σχετικό σεμινάριο για την απλούστευση, ε, απλούστευση των διαδικασιών, κάτι το οποίο έγινε το Φεβρουάριο από την ε, Προεδρία. Και θα πρέπει να δούμε τι γραμμή πλέψης θα ακολουθήσουμε σε σχέση κιόλας με τον δημοσιονομικό κανονισμό, τις δημοσιονομικές προοπτικές για το πρόγραμμα πλαίσιο εκεί όπου έχουμε αντιμετωπίσουμε κάποιους στόχους και γι' αυτό και θα πρέπει να πούμε, όπως και η κυρία Καρβάλιο, ότι πέραν των μέτρων που θα ληφθούν στο μέλλον υπάρχουν και άλλα μέτρα απλούστευσης, έστω και μικρότερου βεληνικούς. Αυτά μπορούμε να τα εντάξουμε στο πρόγραμμα πλαίσιο και αυτό θα διευκόλυνε τους εμπλεκόμενους. Αλλά πέραν αυτού, νομίζω, αυτό θα ε, έφερνε μεγαλύτερη συμμετοχή. Πάρα πολύ πλήρης η έκθεση. Και μπράβο τους και πάλι σας λέω. Τώρα, εγώ είμαι σκιώδης εισηγητρία για την ε, πολιτική μου ομάδα. Έχω κατεβάσει κάποιες τροπολογίες και θέλω τώρα να σας πω ότι κάποιες παρατηρήσεις προφορικά γιατί νομίζω ότι είναι θεμητό το να θέλουμε να προστατεύσουμε τα συμφέροντα της Ένωσης. Αλλά αυτό δεν περιορίζεται μόνο στο περιθώριο του 2%. Θέλουμε αυτό να αφορά και την έρευνα, θέλουμε να δούμε πώς θα καλύψουμε για τους κινδύνους που εγκυμονούνται και που δεν είναι εύκολο πάντοτε να προβλέψουμε. Για όλους θέλουμε να κάνουμε κάτι και όχι μόνο για τους ερευνητέ, όπως θα είπε η κυρία Καρβάλιο και μας ανέφερε κάποια παραδείγματα, να σας πω και εγώ ότι θα άξιζε να δώσουμε έναν ορισμό ξεκάθαρο στην έννοια του λάθους. Τι γίνεται, πώς προκύπτουν τα λάθη. Να συμφωνήσουμε τι θα πει συνήθις λογιστική πρακτική των επιλεξίμων. Έλεγχη εκ των προτέρων. Για τους νεοεισελθόντες στο σύστημα, για αυτούς που εκτίθεται για πρώτη φορά μόνο στους κινδύνους ας κάτσει που να τα ξεκαθίσει αυτή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ας εφαρμόσει τους ίδιους κανόνες που ισχύουν για όσους είναι επιλέξιμοι για το πρόγραμμα πλαίσιο. Αυτό για τους οικονομικούς ελέγχους και ότι θα πρέπει σαν πλεονέκτημα να τους αναγνωρίσουμε το ότι μπορούν να έχουν ένα πιστοποιητικό για τον λογιστικό έλεγχο εκ των προτέρων. Όλα αυτά θα κάνουν πιο εύκολη τη δουλειά, πιο εύκολη τη συμμετοχή στους μελλοντικούς διαγωνισμούς και αυτά με ορίζοντα το 2013. Ευχαριστούμε, Πρόεδρε, και την Βελγική Προεδρία, γιατί από την πρώτη μέρα ασχολήθηκε με το θέμα. Έχουμε και εκείνο το σεμινάριο για την απλούστευση που είπαμε, οπότε θα βοηθήσουμε και εμείς όσο μπορούμε την βελική Προεδρία της προσπάθειάς της. Ευχαριστώ κ. Χατζημαρκάκης. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Δεν θα μπορούσαμε να βρούμε καλύτερη συγκήτρια από την κυρία Καρβάγιο γιατί το ξέρει το θέμα. Είναι πολύ καλά προετοιμασμένη, ξέρει και την παραμικρή λεπτομέρεια και πρέπει να είμαστε πολύ ευχαριστημένοι που έχουμε τη συγγήτρια. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνεργασία και για την προπαρασκευαστική εργασία. Η απλούστευση δεν είναι αυτός σκοπός. Θα πρέπει να εξυπηρετεί δύο σκοπούς. Πρώτα απ' όλα πρέπει να ενισχύσουμε την συμμετοχή στα προγράμματα πλαίσια, κυρίως των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και πρέπει να αυξηθεί και η ορατότητα της έρευνας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι πλέον ορατή. Δεν γνωρίζουμε τι παρέχει, ποια είναι το φέλη της ευρωπαϊκής έρευνας. Γιατί χρειαζόμαστε να δείξουμε στον κόσμο την έρευνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και μετά είναι η άλλη ιδέα της αλλαγής της προσέγγισης τονίζοντας περισσότερο την επιστημονική παρά την διοικητική πτυχή. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας έχει καθορίσει κάποιες αρχές. Νομίζω ότι υπάρχουν κάποιοι τομείς όπου πρέπει να σπρώξουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή παραπάνω. Ένας τομέας είναι η συνοχή χρησιμοποιούνται διάφορες ορολογίες, διάφορα λογιστικά συστήματα, διάφορες γενικές διευθύνσεις που ασχολούνται με διαφορετικούς τομείς, ενίο έλεγχος είναι σαφής έννοια, όλα τα τμήματα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως θα πρέπει να εργάζονται ως μία μονάδα για να κάνουν αυτή τη δουλειά. Χρειαζόμαστε ασφάλεια δικαίου, ε, νομική σαφήνεια, εκ των υστέρων δεν είναι αποδεκτές, κυρίως για τους μικρότερους συμμετέχοντες, δεν είναι αποδεκτό να αλλάζουν οι κανόνες εκ των υστέρων. Δεν είναι αποδεκτό αυτό. Η κυρία Καρβάγιο αναφέρθηκε σε καταποκοπήν ποσά και αυτό είναι σημαντικό θέμα. Ο χρονικός παράγοντας παίζει ρόλο. Πώς μετά από 200 μέρες παίρνουν τα χρήματά τους κάποιοι φορείς και άλλοι χρειάζονται 500 μέρες για να πάρουν τα χρήματά τους. Δεν είναι εύκολο να το καταλάβει κανείς. Χρειαζόμαστε υποστήριξη ε, της πληροφορικής. Αυτό είναι κάτι που αναφέρθηκε. Και όπως είπε και η κυρία Ριέρα Μαδουρέλ, πρέπει να εξετάσουμε και το ποσοστό σφάλματος, το περιθώριο σφάλματος. Δεν μπορούμε να θέτουμε ένα όριο σφάλματος 2% σε διοικητικό επίπεδο. Πρέπει να ακολουθήσουμε πιο ευφυή προσέγγιση. Βεβαίως υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός, κυρίως από την Ασία στον τομέα αυτό. Ευχαριστώ ο κύριος Λάμπερτς και εγώ όπως και οι συνάδελφοί μου θα συγχαρώ εκ νέου την εισηγήτρια. Έγινε αυτό δημοσία και κατηδίαν πολύ καλή έκθεση, θα επαναλάβω τα υποθέτα να εστιαστώ σε δύο πράγματα. Πρώτα απ' όλα ε, η προσέγγιση που προσανατολίζεται προς το αποτέλεσμα. Αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να προσπαθήσουμε να πετύχουμε. Όμως θα πρέπει να αποφύγουμε να, την παγίδα του καθορισμού εκ των, εκ των προτέρων τι αναμένουμε από την έρευνα. Διότι η έρευνα σε οδηγεί και σε απροσδόκητα αποτελέσματα και τομείς. Και αν μάλιστα θέλουμε να πετύχουμε συγκεκριμένα αποτελέσματα και να κινηθούμε ανάλογα, δεν ξέρω κατά πόσο θα ταιριάζει και ένα πρόγραμμα στο ITER. Διότι το αποτέλεσμα τέτοιου προγράμματο θα δώσει τι. Δεν γνωρίζουμε, ελπίζουμε βέβαια, αλλά δεν ξέρουμε. Και πότε, κανεί δεν γνωρίζει. Γι' αυτό λοιπόν, αν εφαρμόσουμε αυτή την αρχή, το ITER δεν θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί. Και έρχομαι στο δεύτερο. Στρεφόμαστε στο ΖΑΜΠΙΑ Οντί. Σίγουρα αντιδράσει αυτό θα πω. Έχουμε δύο βασικά προγράμματα τα οποία είναι εντελώς ανεξέλεγκτα δημοσιονομικά. Η κυρία Καρβάγιο αναφέρθηκε στο πρόγραμμα πλαίσιο 8. Α, θα έπρεπε να αναφέρουμε κάτι στην έκθεση για το 8ο πρόγραμμα πλαίσιο. Για να περιορίσουμε τις δυνατότητες τα προγράμματα να γίνονται ανεξάρτητα έχουμε το ΙΤΕΡ και το Γαλιλαίος. Το ΙΤΕΡ είναι τύπου 3. Το Γαλιλαίος δεν ξέρω ποιο είναι το ποσοστό όσον αφορά το κόστος και την αύξηση του κόστους. Ποιο είναι το πρόβλημα όμως. Συνήθως τα κράτη-μέλη λένε καλώς, δεν θέλουμε να δώσουμε και άλλα χρήματα, άρα θα πρέπει να χρηματοδοτήσουμε αυτά τα προγράμματα και την αύξηση των δαπανών κάνοντας περικοπές από άλλα σχέδια του ίδιου προγράμματος. Στην έκθεση θα έπρεπε να πούμε κάτι. Πώς θέλουμε να περιορίσουμε να συμβαίνει αυτό. Κάποια προγράμματα θα υποφέρουν λόγω Twitter και του Γαλιλαίος και αυτό δεν θα πρέπει να το δούμε με θετικό μάτι. Ίσως θα μπορούσαμε να βάλουμε μια παράγραφο. Θα προσπαθήσω να προτείνω κάτι σχετικό, διότι είναι θέμα κακής διαχείρισης. Και η Ευρώπη έχει τη φήμη ότι δεν χειρίζεται τα χρήματά της πολύ συνετά και εδώ έχουμε δύο σημαντικά παραδείγματα όπου η εικόνα που προβάλλουμε προς τους πολίτες δεν είναι καλή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κυρία Καρβάγιο, λέει κυρία Φόρντ. Ήταν επόλαυση, ευχαρίστηση να δουλεύουμε μαζί σας. Συγχαρητήρια λοιπόν. Να μπορεί να χρησιμοποιείται η συνήθις λογιστική προσέγγιση σημείο 10 και το 14 για τα μικρότερα κονσόρτσια. Εγώ ξέρω από την περιοχή μου ότι όσα προσθέτεις στα κονσόρτσια τόσο προσθέτεις στον περίπλοκο χαρακτήρα και στο κόστος δεν είναι μόνο ο αριθμός των συμμετοχών των φορέων παίζει ρόλο και οι γεωγραφικές αποστάσεις. Τούτων λεχθέντων, σας ευχαριστώ που συμπεριλάβατε και την ανάφορα στη διεθνοποίηση. Το συζητήσαμε αυτό και με κάποια πανεπιστήμια μας. Και χαίρονται που γίνεται αυτή η αναφορά. και ευχαριστώ που συμπεριλάβατε και το σημείο αυτό το σχετικά με το πλησίασμα των αγορών. Πολύ συχνά είμαστε σε μειονεκτική θέση ανταγωνιστικά στην Ευρώπη. Έχουμε πολύ καλή έρευνα που διεξάγεται. αλλά δεν πάμε το προϊόν στην αγορά. Αν πρέπει να το ταιριάξουμε και με άλλες προσπάθειες ε, που γίνονται στο Κοινοβούλιο, κρατικές προμήθειες, κεφάλαια κινδύνου κλπ. Ούτω ώστε να προωθούμε τα νέα προϊόντα, ίσως θα πρέπει να το εξετάσουμε. Δεν είναι μόνο το πρόγραμμα πλαίσιο 8 πρέπει να αναφέρεται, αλλά πώς συνδέεται η προσπάθεια με το επόμενο επίπεδο, την καινοτομία. Διότι αυτό είναι το κλειδί για το μέλλον της Ευρώπης. ήταν πολύ περίπλοκο, απίστευτα περίπλοκο το πρόγραμμα πλαίσιο, το 8ο πρόγραμμα πλαίσιο και υπήρξαν προβλήματα. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι η χρηματοδότηση που έχει σαν στόχο την εκροή, το αποτέλεσμα. Μου αρέσει η ανάλυση που κάνετε εκ των άνω προς τα κάτω και τον κάτω, από κάτω προς τα πάνω. Πάντα παραπονιόμουν για την έλλειψη διαφάνειας στα λογιστικά. Και νομίζω ότι είναι σημαντικό να έχουν περισσότερη διαφάνεια στα λογιστικά και πάντοτε θα πρέπει όφελο κόστο να λαμβάνονται υπόψη όσον αφορά τον λογιστικό έλεγχο και είδα ότι αυτό έχετε καλύψει αυτό και θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι θα πρέπει να υπάρχει σωστή, σωστή ε, εποπτεία. Και στη δική μου ε, εκλογική περιφέρεια είχαμε έναν φορέα που είχε φτάσει να υφίσταται ταυτοχρόνως τέσσερις οικονομικούς ελέγχους. Ευχαριστώ κύριε Ματίας, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Και εγώ να συγχαρώ την κυρία Καρβάλια για τα όσα έχει επιτελέσει για το, τη δουλειά της με την έκθεση αυτή που είναι υποδειγματική και όχι μόνο κάλυψε τα όσα θέλαμε οι σκιώδεις εισηγητές, αλλά γιατί πάρα πολύ δημοκρατικά δούλεψε και μας εκάλυψε. Είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε ότι ο τελικός στόχος είναι η απλούστευση. Και γι' αυτό οι προτάσεις της εισηγήτριας επιτυχώς καλύπτουν και με το παραπάνω την απλούστευση στα διοικητικά και στα οικονομικά. Πολύ σημαντικό αυτό. Τα εξής μου φαίνονται σημαντικά. Το σημείο 23 της έκθεσης όσον αφορά τα της χρηματοδότησης με βάση το αποτέλεσμα. Πολύ σημαντικό. Παρακαλώ συνάδελφοι να το λάβετε υπόψη. Έχουμε το παράδειγμα του ε, Έχουμε επίσης μια ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όπου όμως δεν δίνεται ούτε η χρονική διάσταση του πράγματος ούτε ο ορισμός του τι θα πει αποτέλεσμα. Τα είπε ο κ. Λάμπερς πριν από λίγο. Μεγάλη προσοχή να κάνουμε. Να δούμε πώς θα προστατευτούμε έναντι των κινδύνων της αλλαγής στο σύστημα χρηματοδότησης. Βάσει τα αποτελέσματα και με βάση την επιστήμη τώρα. Πάρα πολύ καλά τα λέει η κυρία και με έχει καλύψει. Έχω άλλες τρεις γενικές παρατηρήσεις να σας αναφέρω. Απλούστευση είναι ο τελικός στόχος και γι' αυτό θα πρέπει ευρωπαϊκός χώρος έρευνας να αναδειχθεί. Να εκμεταλλευτούμε όλες τις δυνατότητες του χώρου. Επομένως, βοηθούν τέτοιες εκθέσεις. Να υπάρχει ισότητα πρόσβασης από όλα τα θεσμικά όργανα και όλα τα κρατημέρη με εις, ε, τους πόρους που υπάρχουν. Να μην υπάρχει κεντροκατευθυνόμενη διαχείριση όσον αφορά την διαχείριση των πόρων. Επίσης κάτι άλλο, πολλές φορές ξεχνούμε ότι ο ευρωπαϊκός χώρος και ας λέγεται ευρωπαϊκός δεν σταματά στα σύνορα της Ευρώπης. Θα πρέπει να σκεφτούμε τα διεθνή δίκτυα. Υπάρχουν αυτά. Υπάρχουν και εκτός Ευρώπης. Μην το ξεχνούμε να το λαμβάνουμε υπόψη πάντα. Και έτσι να προχωρούμε με αυτόν τον τρόπο στην ενίσχυση του ευρωπαϊκού χώρου έρευνας σε σχέση με τους εξωτερικούς, τους εκτός Ευρώπης εταίρους μας. Υπάρχει σχέση μεταξύ έρευνας βάσης και εφηρμοσμένης έρευνας. Αν ε, προσέχουμε και τους δύο κλάδους, θα είναι πιο βιώσιμη η προσπάθειά μας. Πολύ σημαντικό να το προσέξουμε και αυτό. Και αυτό είναι και το ατού του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας. Ευχαριστώ. Έτσι ακούσαμε τους κοιόδης ηγητάς και τώρα έχω ακόμη συναδέλφους εγγεγραμμένους με την επισήμανση παρακαλώ στο δυνατόν πιο σύντομα. Ε, ο κύριος ε, Μπρεζίνα παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, να θα είμαι και εγώ σύντομος. Η συγγετρία έχει ιδιαίτερα δώσει έμφαση στην έρευνα, την κατάρτιση και ασφαλώς θα πρέπει να διευκολύνουμε τα πράγματα και γραφειοκρατικά, γιατί είναι μεγάλο το γραφειοκρατικό άχθος. Ε, θα ήταν καλό να εξασφαλιστεί μια ισορροπία μεταξύ εμπιστοσύνη και ελέγχου, δηλαδή του κινδύνου και του μετριασμού, αυτού του και μετριασμού του κινδύνου. Ε, και γι' αυτό έχω καταθέσει κάποιες τροπολογίες με βασικές αρχές όπως ε, αποδείξεις για κάποιες δαπάνες των πανεπιστημίων, ερευνητικών κέντρων κτλ. με πιο απλουστευμένες διαδικασίες και πιστεύω ότι Ίσως θα πρέπει να εξηγήσουμε γιατί η προσέγγιση που έχουμε για συγκεκριμένα αποτελέσματα χρειάζεται νέα, νέες λύσεις, απαιτεί νέες εφαρμογές. Αυτό όμως είναι μια λεπτομέρεια. Πάντως η έκθεση μου φαίνεται ευπρόσδεκτη και ιδιαίτερα στη στιγμή κατά την οποία περιμένουμε την ενδιάμεση αναθεώρηση του 7ου προγράμματος πλαισίου και κάνουμε, ξεκινάμε την προετοιμασία για το 8ο. Ευχαριστώ. Κυρία Εκ. Εγώ θα, θα συγχαρώ την εισηγήτρια, έξοχη δουλειά που έκανε, υπέροχη έκθεσή της. Να αναφερθώ σε κάποια σημεία που πρέπει να ξεκαθαρίσουμε σαν Επιτροπή. Αυτή η έκθεση πρωτοβουλίας είναι βάση των συζητήσεων. όταν συζητήσαμε και το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο και όταν σχεδιάζαμε το, πρόγραμμα, το 8ο πρόγραμμα πλαίσιο. Η προσέγγιση που έχει σαν στόχο το αποτέλεσμα είναι καλή, όχι μόνο επιστημονικά, αλλά και από πλευρά ελέγχου. Και είναι, εάν είχαν δηθεί χρήματα για να πάει κανείς από α στο β μεταξύ και βρει κανείς ότι είναι πιο γρήγορο και απλούστερο και φθηνότερο με λεωφορείο και δεν σου επιτρέπεται να πάει στο λεωφορείο. Έτσι μοιάζει ο έλεγχος που έχουμε σοφά την έρευνα και τα ερευνητικά προγράμματα. Και το να εργάζεται κανείς σε πανεπιστήμιο και να προσπαθεί να χειριστεί προγράμματα τέτοια είναι κάτι αδύνατον. Και φαίνεται διότι είναι δύσκολο το μεγάλο πανεπιστήμιο να συμμετάσχει όπως πρέπει και αν δείτε και το ποσοστό συμμετοχή της βιομηχανία μειώνεται εδώ και 15 χρόνια, όταν εμεί θέλουμε μεγαλύτερη συμμετοχή και δραστηριότητε στην Ευρώπη όσον αφορά την έρευνα. Επίσης έχουμε ένα σύστημα όπου τα πρότυπα ελέγχου ή τα λογιστικά πρότυπα αλλάζουν κατά τη διάρκεια του προγράμματος ή πριν τον τελικό έλεγχο και αυτό βάζει τον υπεύθυνο να αντιμετωπίζει απίθανα προβλήματα και τρομάζει τον κόσμο. Θα πρέπει να έχουμε μια τελική ημερομηνία για τον έλεγχο και επικροτώ και την πρόταση για ενία για, πιο, για συντονισμό των εφαρμογών πρέπει να επιληθούν τα φορολογικά προβλήματα. Όταν δημιουργείται μεγάλο ερευνητικό πρόγραμμα, ίσω χρειάζεται και ένα χρόνο για να επιληθούν τα προβλήματα πνευματικών δικαιωμάτων και σχετικέ συμφωνίε. Χρειαζόμαστε προδιαγραφέ λοιπόν για αυτή την προσέγγιση για τα πνευματικά δικαιώματα. Ένα χρόνο για να το λύσει αυτό, όταν ξέρει τι θε να κάνει, ξέρει τι δυνατότητε και τα τελικά ενδεχόμενα αποτελέσματα και κολλά στα πνευματικά δικαιώματα και τι σχετικέ διαπραγματεύσει είναι τρέλα. Επικροτώ και την πρόταση για ενία βάση ε, για τη, για τη συλλογή πληροφοριών και την ενημέρωση. Αυτό ήταν συγκεκριμένο πρόβλημα που αντιμετώπιζε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Τέλος, υπάρχει μια φράση που θα πρέπει να διευκρινιστεί. Αυτό που λέει η συγγήτρια δηλαδή, όταν αναφέρεται στη διοντολογία και τη συμμετοχή των κρατών μελών. Είναι σαφές ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να πούν δεν θέλουμε να συμμετάσχουμε, αλλά θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο ότι δεν μπορούν να σταματήσουν άλλους από το να συμμετάσχουν και αυτό θα πρέπει να αναφέρεται ρητά στο τελικό κείμενο. Διότι θυμηθείτε τη συζήτηση που έλαβε χώρα όσον αφορά την έρευνα για τα βλαστοκύτταρα. Όταν τα χρειαζόταν κάποιοι για να επιληθούν προβλήματα όπως διαβήτης και ο ρευματισμός, το ήθελαν οι ρευματισμοί, και κάποια άλλα κράτη-μέλη δεν το επιθυμούσαν. Το αντεπιχείρημα ε, για το πυρηνική ενέργεια. Δεν μπορούν τα κράτη-μέλη να σταματούν ε, άλλους από το να ερευνούν συγκεκριμένους τομείς. Αυτό χρειάζεται διευκρίνηση. Και τέλος, η πέμπτη ελευθερία, η, με, η μετακίνηση και της γνώσης και των ερευνητών. Αν εφαρμόζεται αυτό σε ένα πρόγραμμα, Μάλλον, εάν ε, λειτουργεί ένα πρόγραμμα, θα πρέπει να επιτρέπεται να συνεχίσετε το πρόγραμμα ακόμα και να αλλάξει το πανεπιστήμιο. Η Αγγέλικα Νίμπλερ έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχάς, θα συμφωνήσω κι εγώ με τους επένους των συναδέλφων για την έκθεση. Ήταν όντω εξαίρετη η έκθεση της κυρίας Καβάλιο. Ιδιαίτερα δεδομένου ε, και της πίεσης χρόνου που είχε για να ετοιμάσει το κείμενό της. Συγχαρητήρια λοιπόν. Κάποιες γενικές παρατηρήσεις καταρχάς. Ναι, και είχα την ευκαιρία να ζήσω και την προετοιμασία του 7ου προγράμματος πλαισίου, όπου πάλι μιλούσαμε για απλούστευση, πάλι μιλούσαμε για τις περιπλοκές διαδικασίες για την καταθέση των αιτήσεων, που πρέπει να απλουστεύσουμε, που πρέπει να επιταχύνουμε, πρέπει να καταθέσουμε πιο διαφανείς. Ναι, πρέπει νομίζω ότι όλα αυτά που λέμε πλέον να γίνουν πράξη. Τα λόγια τα έχουμε και τα έχουμε πει πολλές φορές, αλλά δεν υλοποιούνται δυστυχώς. Α κάνουμε άλλη μια προσπάθεια, εν πάση περιπτώσει, σε τα ίδια πράγματα και σε ελπίσουμε ότι η Επιτροπή και η αρμόδια υπηρεσία, αποκεντρωμένη υπηρεσία, θα βρει τον τρόπο να το πράξει. Ιδιαίτερα, δεν θα ήθελα να περάσω τώρα στην παρατήρηση, με ενδιαφέρει να πω ο, η ένταση επαλήθευση των ε, ερευνητικών προγραμμάτων θα πρέπει να μας απασχολήσει και με κριτήριο το μέγεθος ενός προγραμμάτος, δηλαδή να δούμε αν είναι ένα μεγάλο πρόγραμμα, ευρύ πρόγραμμα ή μικρό, ε, αναλόγως, χωρίς φυσικά αυτό να σημαίνει ότι θα έχουμε ε, λιγότερη ακρίβεια στην επαλήθευση τη στήριξη των όρων κτλ. Αλλά ένα πρόγραμμα το οποίο είναι μικρό και σε όγκο χρηματοδότηση περιορισμένο δεν θα πρέπει να το επιβαρύνουμε με πολύ μεγάλη και περιττή γραφειοκρατία. Να υπάρξει μια κάποια διαβάθμιση δηλαδή. Και πολύ ωραία το περιγράφετε και εσείς κυρία Καρβάλιο στην έκθεσή σας να ε, ακολουθεί η ένταση του ελέγχου των επαληθεύσεων το μέγεθος ή τον όγκο του προγράμματος. Νομίζω ότι μπορούμε να έχουμε διαφορετική ε, ανοχή, περιθώριο φάρματος ανάλογα με το μέγεθος του σχεδίου. Επίσης, αναφέρθηκε το Γαλιλαίος και το Ιτρι. Νομίζω ότι καλό θα είναι να αναγνωρίσουμε ότι έχουν προχωρήσει καλά τα είδου σχέδια και να αποφασίσουμε εάν θέλουμε να έχουμε τέτοια σχέδια. Νομίζω ότι συμφωνούν όλοι οι συνάδελφοι ότι και το ΙΤΟ και το Γαλλέος αξίζουν υποστήριξης. Ταυτόχρονα έχουμε πει ότι δεν θα πρέπει τα σχέδια που χρηματοδοτούνται να είναι ε, όχι διακυβερνητικά, ούτε εθνικά καθαρά, δηλαδή να αναπτύσσονται μόνο μέσα σε ένα κράτος, αλλά ε, να έχουν τον ευρωπαϊκό χαρακτήρα. Μόνο τότε αξίζουν τη χρηματοδότηση. Πρέπει να δούμε βέβαια και τις δομές διαχείρισης με ένα σχέδιο διαχειριστικό καθώς είχαμε πρόσφατα και τη σχετική παρουσίαση στην Επιτροπή μας. Και γι' αυτό με ενδεχόμενο τα προγράμματα αυτά, ε, με δεδομένο μάλλον θέλουμε να τα χρηματοδοτήσουμε τα προγράμματα αυτά, ίσως θα πρέπει να σκεφτούμε και το ενδεχόμενο να, να ενεργοποιήσουμε τα αποθηματικά. Ο κύριος Σουκαλάς έχει το λόγο. Ε, κύριε Πρόεδρε, να προσθέσω και τα δικά μου συγχαρητήρια στην αξιότιμη κυρία συνάδελφο, την κυρία Καρβάλιο για την πολύ καλή δουλειά της πράγματι, καθώς επίσης να ευχαριστήσω και τους κυρίους και κυρίες συναδέλφους που με τις παρατηρήσεις επισύρουν την προσοχή σε ζητήματα τα οποία ταλαιπωρούν την ευρωπαϊκή έρευνα και καινοτομία επί μακρά σειρά ετών. Πολύ φοβούμαι ότι όσο καλή και να είναι η έκθεση και όσες καλές να είναι οι παρατηρήσεις, έχουμε ένα σύστημα στην Ευρώπη το οποίο χρειάζεται να αποτελέσει αντικείμενο πραγματικά καινοτομικής δράσης για να αντιμετωπίσουμε με νέο μάτι το τι γίνεται σχετικά με την έρευνα και την καινοτομία, τη διαχείριση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων με εντελώ νέα προοπτική. Εχθές το απόγευμα είχαμε την ευκαιρία να ακούσουμε τη φωνή πέραν του Ατλαντικού υποδεικνύουσα διάφορα σημεία στα οποία η Ευρώπη διαφέρει από τους ανταγωνιστές μας. Διάφοροι συνάδελφοι επισήμαναν ήδη ότι το πεδίο της διεξαγωγής της έρευνας δεν είναι πια η Ευρώπη, είναι το παγκόσμιο σκηνικό και στο παγκόσμιο σκηνικό με παγκόσμια όπλα πρέπει να ανταγωνιστούμε εάν πρόκειται να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις που εμείς οι ίδιοι με τις εκθέσεις μας προδιαγράφουμε για το 2025. Είναι, ε, ε, θεώρησα τον εαυτό μου χαζό να μου υποδεικνύει ο, ο Αμερικάνος γερουσιαστής ότι δεν πήραμε ακριβώς είδηση τι κάνουν οι Κινέζοι με τις σπάνιες γέες και επίσης αισθάνθηκα χαζός όταν μου έλεγε ότι δεν χρειάζεται να κάνουμε επιτροπές των επιτροπών αλλά αυτοί ό,τι δουλειά έχουν να την κάνουν πηγαίνουν στα NSF και παίρνουν τα λεφτά τους. Δεν με ενδιαφέρουν αυτά που λέει ο Αμερικάνος. Με ενδιαφέρει τι λέει η πραγματικότητα. Και η πραγματικότητα είναι η ακόλουθη. Η Ευρώπη αποτελεί ένα μέρος όπου η επιστήμη, η τεχνολογία και ο πολιτισμός βρίσκονται στην κοιτίδα τους και δεν έχει βρεθεί ακόμα ο τρόπος και ο δρόμος ώστε η παραγωγή, δηλαδή οι ερευνητές, οι επιχειρήσεις και η βιομηχανία να συνεργαστούν με τον ομαλό, απρόσκοπτο και φυσιολογικό τρόπο που παράγει πρόοδο και πλούτο. Αυτό δεν φαίνεται να βοηθιέται από όλο ένα και πιο λεπτομερείς κανονισμούς που υποτίθεται ότι βελτιώνουν και απλουστεύουν τις διαδικασίες. Στη βάση όμως, επειδή πρόκειται για σύγκρουση δύο εξουσιών, δηλαδή του παραγωγού ερευνητή επιστήμονα και της ελέγχουσας διοικητικής αρχής, στη βάση της διαφάνειας και του εξορθολογισμού των δαπανών που τίθενται στην διάθεση των επιστημόνων, ανάγκη είναι επιτέλους να γίνει αυτό που και η κυρία Καρβάλιο αναγνωρίζει στην έκθεσή της, μια πολιτική εμπιστοσύνης η οποία δεν θα οδηγεί σε ατιμορρησία, αλλά θα οδηγεί σε διαφανή αποπομπή από το σώματος των ερευνητών εκείνων που παραβιάζουν τους κανόνες, αλλά και θα αφήσει ελευθερία και αναπνοή στους ερευνητές. Ευχαριστώ πολύ. Ο το λόγο. Ευχαριστώ και ευχαριστώ και την ε, εισηγήτρια. Νομίζω είναι ορθή η προσέγγιση να ε, έχουμε διαφορετική μεταχείριση για τα μικρότερα σχέδια. Πρέπει και οι δαπάνες βεβαίω να επαληθεύονται, αλλά και αυτό που θα έλεγα έσοδα, δηλαδή συγκεκριμένα το ότι προσφέρουν ε, ως πλέον έκτημα, ως κέρδος για την Ευρώπη τα προγράμματα αυτά κατά την εκτέλεσή τους. Θα πρέπει να μπορούμε να κάνουμε μια αποτίμηση δηλαδή των, ε, της αποτελεσματικότητάς τους και των πλέον εκτιμάτων που μας προσφέρουν. Και επίσης ε, για το, για το 8ο πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα για να κερδίσει αξιοπιστία θα πρέπει και ε, ο κόσμος βέβαια, οι Ευρωπαίοι, αλλά και οι αρχηγοί και κυβερνήσεων να αντιληφθούν τη σημασία του και έτσι όταν λαμβάνουν τι αποφάσεις για τη χρηματοδότηση να μην περικόπτουν τα κονδύλια. Το one-stop shop, η μονοθυριδική προσέγγιση, είναι επίσης κάτι που έχει αναφερθεί πολλές φορές. Σημαίνει δηλαδή γρήγορα και αποτελεσματικά να λαμβάνονται οι αποφάσεις ε, γιατί πολλές φορές μια απόφαση εάν κρατήσει έξι εβδομάδες μέχρι να ληφθεί, είναι πολύ αργά για ορισμένα σχέδια. Σύντομα λοιπόν περιθώρια για τη λήψη απόφαση και γρήγορη καταβολή των κονδυλίων, ώστε ιδιαίτερα μικρέ και μισέ επιχειρήσει να μπορούν να δραστηριοποιηθούν χωρί δυσκολίε. Και το ίδιο πιστεύω με το έντυπο το οποίο θα πρέπει να είναι στη διάθεση του ενδιαφερομένου σε μία γλώσσα κατανοητή. Ε, ενδεχομένως το έντυπο το ίδιο να είναι τυποποιημένο όπως ε, έχουμε, αλλά να υπάρχει ένα συνοδευτικό έγγραφο διαθέσιμο στην κάθε γλώσσα που θα εξηγεί το κάθε, η κάθε θέση, το κάθε τετραγωνάκι, το νούμερο 1, το νούμερο 2, τι πρέπει να συμπληρώσει. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Κοβίνσκα, έχει το λόγο. Ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω την συγγήτρια για αυτή την έκθεση που επισημαίνει διάφορα προβλήματα που αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει η επιστημονική κοινότητα. Είχαμε συζητήσει την απλούστευση στο 7ο πρόγραμμα πλαίσιο και θα έπρεπε να συζητήσουμε βέβαια και το 8ο πρόγραμμα πλαίσιο. Θα πρέπει λοιπόν να ζητήσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προβεί μια ανάλυση για να καταλάβουμε πώς κάποιες χώρες χρησιμοποιούν περισσότερο τους πόρους που διατίθενται και άλλες λιγότερο. Από τις πληροφορίες που διαθέτω, αυτό το πρόβλημα φαίνεται όλο και πιο σοβαρό και τα κράτη-μέλη, τα νέα κράτη-μέλη μάλλον, όμως ε, μαθαίνουν στα, νέα κράτη-μέλη επιστήμονε τι νέε διαδικασίε. Σε αυτή την έκθεση θα ζητήσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προετοιμάσει μία ανάλυση για να καταλάβουμε τι διαφοροποιεί τι χώρες μας και ποια είναι τα φράγματα, οι φραγμοί ε, που έχουν επισημανθεί στα διάφορα κράτη-μέλη για τη σωστή χρήση των διαδικασιών. Υπάρχουν προβλήματα για κάποιους που υποβάλλουν αιτήσει στην Πολωνία και στα άλλα κράτη-μέλη. Και ένα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζονται είναι από το result-based, από την προσέγγιση με στόχο τα αποτελέσματα, να περάσουμε ε, στο cost-based. Το λέω διότι αυτή είναι μια αλλαγή ε, νοοτροπίας και προσέγγισης και χρηματοδότησης και θα πρέπει να υποστηριχθεί. Όμως Πολλές αιτήσει που έρχονται από τα νέα κράτη-μέλη αφορούν τις βασικές έρευνες. Και λοιπόν θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε σαφώς ποια είναι τα αποτελέσματα που αναμένονται. Κατά την άποψή μου αυτό δεν είναι εφικτό. Όσον αφορά τον τομέα των διαφόρων βασικών ερευνών, το θέμα του κόστους δεν μπορεί να είναι το βασικό στοιχείο. Διότι διαφορετικά θα περιπλακεί πάρα πολύ η πρόσβαση στα προγράμματα. Δεν είναι σαφές πώς πρέπει να χρηματοδοτηθεί, ποιο θα είναι το αποτέλεσμα πριν ολοκληρωθεί ένα πρόγραμμα για να χρηματοδοτηθεί. Αυτή είναι η λύση που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υπάρχουν πιο πλούσια ιδρύματα, άλλα πιο φτωχά. Για τα πιο φτωχά ιδρύματα, τα ερευνητικά δεν μπορούν να περιμένουν πολύ για να επιστραφούν τα, οι δαπάνε, γιατί δεν θα τα καταφέρουν διαφορετικά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να χαιρετήσω το τεράστιο έργο που επετέλεσε η συνάδελφός μου, η κυρία Καρβάγιο, λέει ο κύριο Σοντή. Συγχαρητήρια. Και είναι δουλειά που περιμένει και τη δική μας Επιτροπή και την Επιτροπή Ελέγχου Προπολογισμών. Όσον αφορά το ΙΤΕΡ, ας μην το θεωρούμε υπεύθυνο για τα πάντα η επιστημονική φιλοδοξία και η έρευνα του ΙΤΕΡ περνάνε μέσα από διάφορους δημοσιονομικούς περιορισμούς και είναι λυπηρό. Βέβαια υπήρξε και κακή διαχείριση που τίθεται το πρόβλημα της διαχείρισης των μεγάλων προγραμμάτων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τόσο αφορά την σημερινή έκθεση, αν η συγγήτρια συμφωνεί, θα ήθελα να συμφωνήσουμε με μια τροπολογία για να ρυθμίσουμε την παρελθούσα κατάσταση ρυθμίζουμε το μέλλον εδώ, αλλά πρέπει να ρυθμίσουμε και του ελέγχου του παρελθόντο. Διότι αν δεν το κάνουμε αυτό διακριτικά, όλα θα βρεθούν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Θα δημιουργήσουμε έλλειψη δημοφιλία στα κράτη-μέλη τη στιγμή που χρειαζόμαστε για τις επόμενες δημοσιονομικές προοπτικές να δώσουμε μεγαλύτερη έρευνα σε ευρωπαϊκή κλίμακα. Θα προτείνω λοιπόν μια τροπολογία που εν γέννη θα στρέφεται γύρω από την εξή ιδέα. Να πούμε, εφαρμόζοντας την απλούστευση όπου έχει επιτευχθεί εκεί η πολιτική συνένεση στη διευθέτηση των παρελθουσών καταστάσεων. Αυτό προτείνω να πούμε για να στείλουμε ένα σήμα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αποδεχθεί ε, βάση ερεύνας και, αντιπαρα... και αντιπαραβολής να ρυθμιστούν τα παρελθόντα προβλήματα. Κύριος Μέσαρος, Kutatási programjaink főleg az oktatás területén kibővültek az idők során, melyet a jó pályázati lehetőségeknek is köszönhetünk. Azonban figyelembe kell venni azt is, Όσο πάμε και καλύπτουμε περισσότερα θέματα αυτά τα προγράμματα, καλύψαμε και θέματα παιδείας και θα πρέπει να διαρρονίσουμε τις καινούργιες δυνατότητες, θα πρέπει να δούμε πώς θα περιορίσουμε τη γραφειοκρατία, πώς θα περιορίσουμε τις αβεβαιότητες του συστήματος γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορέσουμε να συντονίσουμε τις διαδικασίες να προσέξουμε το 8ο πρόγραμμα πλαίσιο. Θεωρώ ότι θα πρέπει να εμπιστευτούμε περισσότερο τους ερευνητές. Θα πρέπει να λάβουμε περισσότερο υπόψη τις ανάγκες για την καινοτομία και να περιορίσουμε τη γραφειοκρατία. Βεβαίως και υπάρχουν οι οικονομικοί κίνδυνοι, αλλά δεν θα πρέπει να τους φοβόμαστε υπερβολικά. Επίσης, να σιγουρέψουμε το ότι αυτά τα προγράμματα είναι προσβάσιμα στα καλύτερα πανεπιστήμια, στους καλύτερους ερευνητές. να υπόψη και το κόστος αλλά και το αποτέλεσμα. Περισσότερη εμπιστοσύνη. Αυτό που είναι χαρακτηρίζει το καινούργιο σύστημα. Είναι πάρα πολύ καλή έκθεση, θεωρώ. Νομίζω ότι καλύπτει ό,τι χρειάζεται και πρέπει να ευχαριστήσουμε την κυρία Καρβάλιο πολύ για την εκθεσή της. Το σημαντικό είναι ακριβώς το πώς όλα αυτά θα τα εφαρμόσουμε, θα τα υλοποιήσουμε. Κυρία Χέρτσοκ, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να σας πω δύο-τρία πράγματα για την ε, έκθεση. Πρώτα απ' όλα συγχαρητήρια στην ε, εισηγήτρια, γιατί θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντική έκθεση, όμως θα πρέπει να αποφασίσουμε τι θα την κάνουμε. Να προετοιμαστούμε γιατί, ε, για το επόμενο πρόγραμμα πλαίσιο που είναι θέμα τη ΕΙΤΡΕ, αλλά επίση θα πρέπει να δούμε τι αλλαγέ θα γίνουν στο δημοσιογραφικό κανονισμό. Γιατί αν δεν αλλάξει ο δημοσιονομικό κανονισμό, τότε δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε βήματα προ τα εμπρό και άρα ε, δεν θα τηρήσουμε τι υποσχέσει που δίνουμε στου ερευνητέ. Άρα αυτό είναι το πρόβλημα. Ο δημοσιονομικός κανονισμός είναι κανονισμός που σημαίνει ότι περνάει από την ε, συναπόφαση. Και άρα η Επιτροπή Κλειδί εδώ είναι η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Συνάδελφε, όμως το Ελληνικό Συνέδριο δεν αποφάσισε για τους ε, κανόνες του ε, οικονομικού ελέγχου. Όλα αυτά ήταν αποφάσεις των τριών θεσμικών οργάνων. Επομένως θα πρέπει να δούμε πώς θα συνοηθούμε με τους συναδέλφους της ίδιας πολιτικής ομάδας της Επιτροπής Ελέγχου Προπολογισμού γιατί μόνο έτσι θα προωθήσουμε το θέμα. Να μιλήσουμε κυρία Γιάννη την κυρία Γκρέσλε, ε, οι πράσινοι στους πράσινους, αυτό θα βοηθήσει πάρα πολύ. Και να δούμε πώς θα τροποποιήσουμε το κείμενο και εγώ και ο κύριος Σοντή που είμαστε στην Επιτροπή εκείνη μπορούμε κάτι να κάνουμε. Κάτι άλλο τώρα το ανέφεραν οι συνάδελφοι, το ΙΤΕΡ και ο Γαλιλαίος είναι τα βασικά προγράμματα. Όμως αυτά δεν είναι θέματα ερευνητικά, είναι θέματα εδώ δημοσιονομικά. Ο λόγος που έχουμε αυτά τα προγράμματα στα πλαίσια του 7ου προγράμματος είναι το ότι το πολιτές ε, ε, πλαίσιο δεν ε, έχει τροποποιηθεί και είπαμε ότι έτσι δεν μπορούμε να τα βοηθήσουμε αυτά τα προγράμματα στην διάμεση αυτή περίοδο εν ώψη της επόμενης δημοσιονομικής ε, περίοδου και των προοπτικών. Και για το επόμενο μας θέμα έχουν σημασία αυτά. Θα σας τα ξαναπώ, θα επανέλθω. Γνωρίζετε ότι έχουμε 142 δις σαν προϋπολογισμό και από αυτά 8,5 δις πάνε στην έρευνα. Άρα μιλάμε για το 1% του ΕΠ. Και άρα για την έρευνα πάει το, το, το χιλιοστό. Μα θέλουμε μια οικονομία της γνώσης. Πώς είναι το να την έχουμε με, με τόσο λίγα χρήματα, με το 0,0006% ευμένως του ΕΠ μας. Άρα είναι πρόβλημα προπολογισμού και όχι διαχείρισης. Μ' άρεσε που χτες ο Βέλγος Υπουργός είπε ότι θα πρέπει να ε, τα καταφέρουμε καλύτερα, αλλά δεν είναι θέμα ποιότητα. Και εδώ πέρα θα πρέπει να το παρέψουμε με τα κράτη-μέλη και όσον αφορά τη διαχείριση θα πρέπει να δούμε πώς θα έχουμε ερευνητική υποδομή, κάτι δηλαδή που να εκμεταλλεύεται ότι είμαστε 27, 27 κράτη-μέλη. Να τι θα πει η υποδομή. Κάποια κράτη-μέλη συμμετέχουν αλλά δεν είναι όλοι. Έτσι θα πρέπει να προχωρήσουμε στην καλύτερη διαχείριση για να προχωρήσει και το ίτερ και το πρόγραμμα πλαίσιο το επόμενο. Όμως πρέπει να επενδύσουμε και μόνο τότε θα στραφεί επιτυχώς η έρευνα στην αγορά που αυτό είναι το σωστό. Για την Κλάρα Ντελατόρ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ την κυρία Καρβάγιο, την εισηγήτρια. Ευχαριστώ και την Επιτροπή που εξέτασε ενδελεχέστατα το θέμα της απλούστευσης και υποστήριξε εν γέννη τις ιδέες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα ήθελα να επιμείνω ε, επί της παρεμβάσεως της κυρίας Χέρτσοκ. Πράγματι δεν μπορούμε να πετύχουμε τους σκοπούς μας αν δεν συνδυάσουμε τις αποφάσεις όσον αφορά το πρόγραμμα με τις αποφάσεις για τον μουσιονικό κανονισμό και το ανεκτό ποσοστό σφάλματος, κάτι το οποίο θα αναφέρω αργότερα. Συμφωνεί πλήρως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την εισηγήτρια και τους άλλους ότι ο προπλησιασμός των μηχανισμών χρηματοδοτήσεως και των εφαρμοστικών φορέων είναι μια πηγή ε, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, στην πρόταση για το επόμενο πρόγραμμα πλαίσιο θα το λάβει δόντως υπόψη, θα προσπαθήσει να μειώσει τον περίπλοκο χαρακτήρα, θα προσπαθήσει να ενμονίσει τους διαφόρους μηχανισμούς παρέμβασης στο μέτρο του δυνατού. Και εμπιστεύεται το Κοινοβούλιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να μα βοηθήσει ο συνομοθέτη. Καλωσορίζουμε την υποστήριξή σα όσον αφορά την απλούστευση των κανόνων για τον υπολογισμό του κόστου, συμπεριλαμβανομένου και του ε, μέσου όρου του κόστου. Ε, που μας έχει πονοκεφαλιάσει και αυτό θα έχει ύψιστη σημασία για το επόμενο πρόγραμμα πλαίσιο. Όπως έλεγε η συγγήτρια, είναι αδύνατο να γνωρίζουμε πού θέλουμε να επιφέρουμε τις αλλαγές και πιστεύει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στην προσέγγιση μας και στις αλλαγές, διότι όπως γνωρίζουμε όλοι η σταθερότητα αποτελεί τμήμα στοιχείο. Δεν είναι η πλήρης απάντηση, στοιχείο για την απλούστευση είναι. Όμως οι εσδήποτε περιορισμένες αλλαγές στους κανόνες του 7ου προγράμματος πλαισίου 7 θα προταθούν αλλαγές εάν είμαστε πεπισμένοι ότι και ο συνομοθέτης συμφωνεί. Ίσως σχετίζονται οι αλλαγές με το μέσο προσωπικό ατομικό κόστος. Πολλοί, ο κύριος Χατζημαρχάκης, η κυρία Φόρντ, ο κύριος Οντί κλπ. αναφέρθηκαν στις ανησυχίες του σχετικά με τον υπερβολικό έλεγχο και τη μηδενική ανοχή στο σφάλμα από πλευρά Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και η συγγήτρια είπε όσον αφορά την αναδρομική εφαρμογή των κανόνων ότι ανησυχεί. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητά κατανόηση από εσά όσον αφορά αυτό το θέμα, διότι είμαστε σε πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Είμαι υποχρεωμένη να σας πω ότι ποτέ δεν αλλάξαμε αναδρομικά κανόνες, ούτε επανερμηνεύσαμε κανόνες. Όμως σχεδιάσαμε τον έλεγχο της στρατηγικής που συνάδει με την προσέγγιση του λεκτικού συνεδρίου για την ετήσια δήλωση και αυτή η στρατηγική, αυτές οι παράμετροι για ε, τη δήλωση αξιοπιστίας έχουν εγκριθεί από το Κοινοβούλιο. Αυτή η προσέγγιση απαιτεί να εφαρμόσει αυστηρούς κανόνες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκ των υστέρων, ανακτήσεις λοιπά. Και δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό όσον αφορά ε, διότι μας έχουν ε, δοθεί συγκεκριμένες παράμετροι ελέγχου. Γι' αυτό είναι σημαντικό πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπή να καθοριστεί το ανεκτό επίπεδο κινδύνου και γι' αυτό έχουμε εκδώσει σχετική ανακοίνωση. Και είναι σημαντικό το Κοινοβούλιο όπως υπόθηκε, να υποστηρίξει αυτή την έννοια του διαφορετικού ποσοστού ε, ανεκτού κινδύνου για τις πολιτικές. Ανησυχώ λίγο, διότι χτες, όπως γνωρίζετε, η Επιτροπή Ελέγχου Προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου ψήφισε την έκθεση του κ. Πατιτσέλο και νομίζω ότι η Επιτροπή Ελέγχου Προϋπολογισμού δεν ευθυγραμμίζεται πλήρως με αυτά που άκουσα εδώ για το ανεκτό ποσοστό σφάλματος. Είμαι σίγουρος, σίγουρη ότι αν ακολουθήσετε την πρόσκληση της κυρίας Χέτσο για να συνομιλήσετε με τους συναδέλφους της Επιτροπή Ελέγχου Προπολογισμού θα βρεθεί κάποια λύση. Όσον αφορά το χρόνο που πρέπει να διατεθεί η συγγήτρια ζήτησε μείωση ε, στο εξάμεινο να καθοριστεί το όριο αυτό και η συγγήτρια πρότεινε κάποιο σύστημα βαθμολόγησης. Συμφωνώ δεν μπορούμε να περνάμε τόσο χρόνο, να ξοδεύουμε τόσο χρόνο για τη σύναψη τη συμβάσεω και μεγάλο χρονικό διάστημα για την καταβολή των πληρωμών, όπω είπε και η Χέρτσοκ. Μπορούμε να επιφέρουμε βελτιώσει, μη λησμονώντα όμω ότι δεν πρέπει να είμαστε υπερβολικά αισιόδοξοι. Εξετάσαμε στοιχεία από τα διάφορα εθνικά συστήματα και για προγράμματα παρόμοια περιπλοκότητα, να μην το λησμονούμε ότι πάντα το περισσότερο χρονικό διάστημα ασχολούμαστε με προγράμματα στις οποίες συμμετέχουν πολλοί εταίροι για παρόμοιες προσπάθειες τα κράτη-μέλη έχουν περίπου 12 μήνες για να διαθέσουν τους πόρους και είναι σημαντικό για μας να μειώσουμε τον χρόνο μας αλλά να μην υπονομεύσουμε ταυτόχρονα την περίοδο αξιολόγησης και το σύστημα αξιολόγησης από ομολόγους που είναι και η βάση του συστήματός μας. το θέμα του χρόνου λοιπόν δημιουργεί προβλήματα και είναι θεμητό αυτό στους δικαιούχους, κυρίως του πανεπιστημιακού τομέα αν δεν εισαγάγουμε κατά αποκοπήν ποσά για προγράμματα, κατά αποκοπήν ε, ποσά λοιπόν, θα είναι αδύνατον να καταργήσουμε με κάποιο τρόπο ε, τη μέτρηση του χρόνου, διότι ο χρόνος είναι μια από τις παραμέτρους ε, των προγραμμάτων και πρέπει να μετράτε. Η πιο ριζοσπαστική πρόταση είναι να περάσουμε από την προσέγγιση βασίζεται στο κόστο στην προσέγγιση βασίζεται στο αποτέλεσμα. Και ακούσαμε στην αίθουσα αυτή να αναφέρονται διάφορα τον κύριο Λάμπερ, την κυρία Φόρ, την εισηγήτρια, Επίσης και από την κυρία Εκ διάφορες απόψεις για το θέμα που είναι δύσκολο. Δεν συμφωνούν όλοι σχετικά με τα δέοντα να γίνουν, αλλά θεωρήσαμε ότι η μετακίνηση προς το νέο σύστημα όπου καταβάλλονται κατά αποκοπήν ποσά βάση τη αξιολόγηση τη έρευνας που διεξάγεται στα πλαίσια του προγράμματος είναι κάτι το οποίο συμβάλλει στη λύση. Θα μπορούσε τουλάχιστον να μας επιτρέψει να μειώσουμε τους ελέγχους όσον αφορά τις δαπάνες, θα επιτρέψει μεγαλύτερη ευελιξία στα κονσόρτσια για την κατανομή των πόρων ανάλογα με τις επιστημονικές ανάγκες. Ευχαριστούμε την εισηγήτρια που αναφέρθηκε στην προσέγγιση που βασίζεται στην επιστήμη και όχι που βασίζεται στα αποτελέσματα. Ίσως αυτό θα πρέπει να το σκεφτεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ίσως λόγω της αυξημένης ευελιξίας και της ε, Γι' αυτό η Επιτροπή Ελέγχου Προπολογισμού, από ό,τι κατάλαβα χτε, έδωσε πλήρη υποστήριξη σε αυτή την προσέγγιση. Γνωρίζουμε τον κίνδυνο που υπάρχει όταν μετακινηθούμε προς ένα σύστημα όπου θα πληρώνουμε βάση αποτελεσμάτων και άρα μπορεί να υπάρχει διάκριση έναντι πιο επικινδύνων προγραμμάτων. Αυτή βεβαίως δεν είναι η πρόθεσή μας και γι' αυτό προσπαθούμε ε, να έχουμε κοινή αντίληψη όσον αφορά το αποτέλεσμα ή την εκροή ενός προγράμματος όσον αφορά την επιστήμη, διότι επουδενή δεν θέλουμε να ακολουθήσουμε μια προσέγγιση που θα δηλιάζει εναντί του κινδύνου ή που θα υποστηρίζει παρομοίως προγράμματα που έχουν χαμηλή δυναμικότητα. Όπως πρότεινε η συγγήτρια, και άλλοι αγορητές ίσως θα έπρεπε να προχωρήσουμε σε σχετικές πιλωτικές δράσεις. Να πω μερικά λόγια σχετικά με αυτά που είπε η κυρία Ριέρα όσον αφορά την πιστοποίηση. Είναι σαφές οι κανόνες πιστοποίησεως είναι αυστηρότατοι, αποθαρρύνουν πολλούς να ζητήσουν την πιστοποίηση, όμως ευθυγραμμίζονται πλήρως με τις παραμέτρους ελέγχου που προανέφερα. Αν αυτοί αλλάξουν θα μπορούσε να είναι πιο ήπια Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά τη διαδικασία πιστοποίησης. Και τέλος, προσπαθώντας να απαντήσω στο δύσκολο ερώτημα της κ. για τους διάφορες επιδόσεις των κρατών μελών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέλησε πολύ συχνά το θέμα, έγινε εσωτερική ανάλυση, δεν πρόκειται να εξηγήσει πλήρως τα όσα συμβαίνουν. Δύο πράγματα που έχουμε όμως υπόψη, ότι πάντα υπάρχει μια καμπύλη μάθησης όταν μπαίνουν νέα κράτη-μέλη στην Ένωση ή όταν νέες χώρες αρχίζουν να εφαρμόζουν το πρόγραμμα πλαίσιο, οπότε υπάρχει καμπύλη μάθησης. Αλλά υπάρχει σημαντικότερος παράγων, πολύ σημαντικότερος. Είδαμε ότι υπάρχει έντονος θετικός συσχετισμός μεταξύ εθνικής επενδύσεως στις επιστήμες και του επίπεδου συμμετοχής στο πρόγραμμα πλαίσιο. Και αυτό είναι κάτι που είναι σημαντικό, πρέπει να το γνωρίζουμε όλοι. Είναι κάτι που μπορεί να το λάβει υπόψη σε, άλλα, σε άλλες πολιτικές Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτά και ευχαριστώ Πρόεδρε. Έχει στήσει σύντομα το λόγο και ο κύριος Οντί. Μετά θα ξανακούσουμε την εισηγήτρια. Πολύ σύντομα Πρόεδρε. Χρόνια τώρα συζητούμε τον κανονισμό, τουλάχιστον από το 2007 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και όχι η Επιτροπή μας, ε, η Επιτροπή Ελέγχου του Προβολισμού, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει μία πάγια τακτική, χωρίς καμιά απόκληση μεταξύ των δύο επιτροπών μας, της Επιτροπής Βιομηχανίας και της Επιτροπής Ελευθερού Προπολογισμού και μάλιστα το Κοινοβούλιο στο σύνολό του με δύο απαλλαγές που ψήφισε το 2007-2008 και εσείς φαίνεται να λέτε ότι έχει αλλάξει το Κοινοβούλιο στάση κτλ. Όχι. Το Κοινοβούλιο θέλει οι εκρεμείς διαφορές να επιλύονται με φρόνηση, με περίσκεψη. Και δεν ξέρω, Πρόεδρε, ίσω θα ήταν καλό να έχει προσκληθεί και το ελεκτικό συνέδριο σήμερα. Ε, είχε προσδιορίσει το ελεκτικό συνέδριο ένα ποσοστό του 2%, δεν ξέρουμε πού το έβγαλε. Ε, κατά τους ελέγχους του, με, το, με την έκθεση λοιπόν για τη δήλωση αξιοπιστίας, παραβιάζει την ίδια τη συνθήκη, γιατί η συνθήκη ζητεί από το Ελεκτικό Συνέδριο μια συνολική γνωμοδότηση για τους λογαριασμούς Επιτροπής. Δεν το πράττει όμως το Ελεκτικό Συνέδριο για τους ετήσιους λογαριασμούς, ναι, αλλά όχι για τους συμπληρωματικούς. Γι' αυτό λοιπόν, και ζητώ συγγνώμη που ενοχλώ έτσι, αλλά εν πάση περιπτώσει μην ε, παραλαμβάνετε τα ίδια και τα ιδέα για το Ελεκτικό Συνέδριο. Ξέρω ότι από την Επιτροπή Σαντέρ αισθάνεται κάποια δυσφορία απέναντι στην Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αλλά εμεί αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι, είναι η χρηστή δημοσιονομική διαχείριση. Και θέλουμε να διαπραγματευτούμε με τα κράτη-μέλη για να ανεβάσουμε την πάρα και να εξευρωπαίσουμε την έρευνα. Κάντε όμως τους ελέγχους σας και προς όλες τις ε, μονάδες, τα ερευνητικά κέντρα κτλ. που κάνατε ελέγχους, τους, τους βάζετε στο εδόλιο του κατηγορουμένου, τους καταδιώκετε, τους φαίνεται την ΟΛΑΒ μέσα, τους αντιμετωπίσετε σαν εγκληματίες του κοινού ποινικού δικαίου. Εν πάση περιπτώσει αφήστε αυτό το 2%, κοιτάξτε την κοινή λογική, ρυθμίστε τα προβλήματα του παρελθόντος, έχετε κάποιους κανόνες που πρέπει να εφαρμόσετε, ε, λοιπόν εφαρμόσετε τους με περίσκεψη και με εδώ. Και γι' αυτό υπάρχουν ανεξάρτητες μελέτες ελέγχου, δημοσιονομικού ελέγχου, οι οποίες είναι το 1 τρίτο αυτών των τα οποία εσείς ισχυρίζεστε. Βρείτε λοιπόν ποιες είναι αυτές οι ανεξάρτητες μελέτες, κάντε τις ρυθμίσεις, τις διορθώσεις και ας αποφύγουμε να καταφύγουμε, στα, να φτάσουμε στα δικαστήρια για μια δεκαετία, γιατί εμείς θα σας στηρίξουμε σε αυτή την προσπάθεια. Ας μην κάνουμε περιτούς δικαστικούς αγώνες για ψηλουπίδημα και ζητώ συγγνώμη πρόεδρε που είμαι τόσο Όμω, αλλά νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Βούλιο πρέπει να δουν το ζήτημα, γιατί δεν είναι θέμα του ελεγκτικού συνεδρίου. Πρέπει μεταξύ μας να βρούμε τις, τον τρόπο, τον πολιτικό τρόπο επικοινωνίας για να βγούμε από το αδιέξοδο. Ευχαριστώ πολύ και για να κλείσει η κυρία Καρβάλιο, έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Θα είμαι πολύ συντομή. Ευχαριστώ πολύ τους συναδέλφου για τα πολύ ευγενικά τους λόγια. Ευχαριστώ για όλες τις ε, υποδείξεις τους, όλα αυτά ήδη τα που παρατηρήσανε τα έχουμε βάλει στην έκθεση, αλλά βεβαίως θα τα λάβουμε υπόψη ακόμη περισσότερο. Ιδιαίτερα σημειώνω την ε, παρατήρηση για το Ίτερ και το Γαλιλαίος και θα ήθελα ακόμα να συμπληρώσω κάτι για τις παρατηρήσεις σχετικές με τις διοντολογικές αξιολογίες. Το σύστημα το οποίο λειτουργεί σήμερα λειτουργεί ικανοποιητικά πιστεύω και μάλιστα εμένα ιδιαίτερα με ενδιαφέρει και το γνωρίζω γιατί ήμουν υπουργό τότε που το πρότεινα το 2006-2007 γιατί είχαμε μια διελκυστίνδα και ιστορική στην Πορτογαλία εν πάση περιπτώσει η χώρα η οποία δεν θέλει να το εφαρμόσει δεν είναι υποχρεωμένη να το εφαρμόσει αλλά από την άλλη δεν μπορεί και να απαγορεύσει σε κάποια άλλη χώρα που θέλει να εφαρμόσει το σύστημα αυτό να το πράξει. Λειτουργεί λοιπόν καλά, ικανοποιητικά το σύστημα και νομίζω θα πρέπει να το διατηρήσουμε όσα έχει. Και για το στόχο αυτό βεβαίω θα πρέπει να παρεμβούν τα κράτη-μελή, να παρεμβαίνουν όταν προκύπτουν δεοντολογικοί ε, αντίκτυποι, συνέπειες ενός σχεδίου. Και θα ακούσω, θα παρατηρήσω, θα παρακολουθήσω όλα τα όσα είπατε. Ε, θα καταλάβω λάβω υπόψη στην έκθεση. Ο Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ και για να κλείσουμε θα ήθελα να κάνω σύντομα τρεις παρατηρήσεις. Καταρχάς, πολύ σωστά επισημάνθηκε ότι είναι ένα θέμα που μας απασχολεί εδώ και πολύ καιρό. Μιλούμε όχι μόνο για αλλαγές, ε, δεν μιλούμε μάλλον μόνο για αλλαγέ, θέλουμε να τις υλοποιήσουμε, να τις δούμε στην πράξη. Έχουμε πραγματοποιήσει άριθμες ακροάσεις. Ε, μάλιστα ακολουθήσαμε και τον μη συνήθι δρόμο της ομάδας εργασίας, την οποία αναθέσαμε να παρακολουθήσει την ε, τις παρατηρήσεις και τη συνέχεια που δίνεται στα όσα έχουμε πει. Και θέλουμε και με την Επιτροπή Λάχτου του Προπολογισμού φυσικά, αυτές οι προτάσεις να μην είναι απλώς ωραία λόγια, αλλά να οδηγήσουν σε δεσμευτική δράση σχετική με τη διαδικασία. Δηλαδή να αλλάξουμε δεσμευτικά τη διαδικασία, υποχρεωτικά τη διαδικασία και νομίζω ότι πολλοί είναι συνάδελφοι. Κύριε Καρβάλιο, ίσω θεωρείτε ότι μπορείτε να συνεργαστείτε με την Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού. Δεν ξέρω αν είναι αρκετοί συνάδελφοι, νομίζω, οι οποίοι αναφέρθηκαν σε αυτή την, αυτή τη συνεργασία. Επίση, 14 Ιουλίου 2010, 12 ε, το μεσημέρι, προθεσμία καταληκτική για τι τροπολογίε και τελευταία προσωπική παρατήρηση αυτή τη φορά στα θέματα αυτά της ουσίας που συζητούμε τώρα, τα γενικά προβλήματα, όχι το ΙΤΡΕ ή το Γαλιλαίο, Σα μην τα μπερδέψουμε αυτά εδώ μέσα, γιατί είναι πολιτικά συστήματα τα οποία μπορεί κάνει να αξιολογεί διαφορετικά, αλλά πρέπει νομίζω σε αυτό το έγγραφο να μιλήσουμε για μια γενική πρωτοβουλία, αν θέλετε, μια γενική προσέγγιση, μια νέα προσέγγιση για την έρευνα. Ευχαριστώ πολύ για την καλή συζήτηση. Κλείνω το θέμα αυτό στην ημερήσια διάταξη και περνώ αμέσως στο προσεχές θέμα που είναι πάλι ε, θέματα οικονομικά, δημοσιονομικά με την κυρία Χέρτσοκ η οποία ασχολείται με τον προϋπολογισμό. Έχει αναλάβει ένα καθήκον που φέτο, αυτή το, η χρονιά θα είναι ακόμη πιο ε, δυσχερές. Παρακαλώ κύριε Χέρτσοκ. Πρόεδρε ευχαριστώ και πριν... Ε, ξεκινήσω την ε, ομιλία μου, θα θέλω να χαιρετήσω τους επισκέπτες από την Ουγγαρία και τη Σλοβακία που ήρθαν να παρακολουθήσουν ε, την συνεδρίασή μας. Καλώς ήρθατε. Είναι καλό να γνωρίζετε κι εσείς τα σχετικά με την Ευρώπη. Για το προϋπολογισμό. Ο προϋπολογισμός είναι πάντα άχαρο έργο. Κανείς δεν ε, ε, ακούει ευχάριστα θέσεις για τα χρήματα και για τα δημοσιονομικά, αλλά πρέπει βέβαια να τα συστούμε όλα αυτά. Βλέπουμε μια θετική εξέλιξη στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια, που όμως με δεδομένη την, την κρίση, μετά την κρίση, θα πρέπει να δούμε εάν θα μας αφήσει και χρήματα διαθέσιμα επαρκή για αξιοποίηση. Έτσι λοιπόν οι στόχοι για το 2011 θα πρέπει να στηρίξουμε την ευρωπαϊκή οικονομία και την ανάκαμψή της ε, από την ε, τελευταία κρίση και ο προπολογισμός του 2011 θα πρέπει να ακολουθεί τους στόχους της εφιούς αηφόρου και αποτελεσματικής ανάπτυξης όπως έχουμε ορίσει με βάση τους στρατηγικούς του 2020. Η Ήτρε λοιπόν τι μπορεί να κάνει, να στηρίξει την ανταγωνιστικότητα για την ανάπτυξη και την απασχόληση και τα χρήματα για τα οποία γίνεται λόγος για το 2011 είναι 34,42 δισεκατομμύρια ευρώ, δηλαδή 142,1 δις ε, είναι ο συνολικός προϋπολογισμός, είναι ένα μερίδιο από τον προπολογισμό 1% του αέπινο προπολογισμό, δηλαδή 0,001% είναι αυτά που ζητούμε για τη βιομηχανία. Και πρέπει να δούμε πώς κατανέμονται αυτά. Τα 85 εκατομμύρια πάνε στο 7ο πρόγραμμα πλαίσιο, ένα ποσοστό πάει στις υποδομές. 1,5 στο γαϊλαίο Ήτρε και αντίστοιχα προγράμματα τις υποδομές δηλαδή τα έχω βάλει για τον επόμενο χρόνο, για τους ανθρώπινους πόρους μιλάμε για 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ και για την ανάπτυξη και καινοτομία κατάρριξη των πυρηνικών κτλ. Έχουμε τα υπόλοιπα ποσά από τον προπολογισμό. Πρόκειται για κονδύλια που βρίσκονται στο επίκεντρο της οικονομικής, ε, του οικονομικού εξυγχρονισμού και έχουν πολύ μεγάλη σημασία για τα σχετικά προγράμματα. Επίσης, έχουμε να κάνουμε και με τις πρωτοβουλίες ε, τις σχετικές ε, με τη στρατηγική του 2020, καινοτομία, κινητικότητα των νέων πόρους στην Ευρώπη, θέση εργασίας, βιομηχανική πολιτική εν ώψη τη παγκοσμιοποίηση Ο προπολογισμό του 2002 έχει στρατηγικό χαρακτήρα. Διότι καταρχάς ε, νέε εξουσίες ε, που προβλέπει η συνθήκη της Λισαβόνα πρέπει να δοθούν σε εφαρμογή. Έχουμε την καταπολέμηση της εγκληματικότητα ε, και πολλούς άλλους τομεί. Έχουμε επίσης ζητήματα χρηματοδότησης ήδη εγκεκριμένων προγραμμάτων για το Κοσλοντού για το ΣΕΡΤ, για το Γαλιλαίος, προγράμματα τα οποία θα πρέπει να εγγραφούν στην ε, διαδικασία του προπολογισμού για το 2011. Τρίτον, η Ίντρε έχει στρατηγικό χαρακτήρα ως Επιτροπή για την εφαρμογή της στρατηγικής του 2020 και, και των 7 πρωτοβουλειών Φτάνουμε στο τελευταίο κομμάτι επίσης της ε, περίοδου 2007-2013 και θα πρέπει να ξεκινήσουμε την επεξεργασία, την προετοιμασία για τη συζήτηση για το προσεχές δημοσιονομικό πλαίσιο και δεν μπορεί να λησμονούμε ότι προβλέπεται πλέον νέα δημοσιονομική διαδικασία με τη συναπόφαση για πρώτη φορά στην ιστορία του Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει δικαίωμα να συμμετέχει στην διαδικασία, πολύ περισσότερο από ό,τι στο παρελθόν που απλώς γνωμοδοτούσε και έτσι έχουμε για πρώτη φορά την ε, δυνατότητα του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να συμφωνούν σε κάθε γραμμή του προϋπολογισμού μέσα από τη διαδικασία της ε, συνδιαλλαγής. Εγώ, ως ηγήτρια για την Επιτροπή Ήτρε αντιπροσωπώ ε, στις μελλοντικές συζητήσεις για το τριμερή διάλογο το θέμα της ε, καινοτομίας. Θα ήθελα λοιπόν επίσης να πω ποιοι είναι οι στόχοι μας, ε, καταρχάς με δεδομένες στις δινές οικονομικές ε, πολιτικές συνθήκες, ε, τις οποίες βλέπω ότι κάποια κράτη-μέλη θα αξιοποιήσουν ως πρόφαση για να περικόψουν τον προϋπολογισμό και η τελευταία πρωτοβουλία από το Συμβούλιο, μια ανώνυμη συμφωνία για περικοπή κατά 3,6 δισεκατομμύρια ευρώ του προϋπολογισμού αποτελούν μάλλον δυσάρεστες ειδήσει και μάλιστα για μας ένα δισεκατομμύριο πάει στο, στην ανταγωνιστικότητα από τη διαχείριση των προγραμμάτων ε, έρευνας που μόλις συζητήσαμε. Επίσης, ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι μικρός, προπολογισμό, μικρός προϋπολογισμός. Η αδίποτε ενίσχυσή του θα είναι μηδαμινής ε, απήξης, μηδαμινού αντίκτυπου ως προς το συνολικό προϋπολογισμό των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ κάθε περικοπή του μπορεί να έχει σημαντικές δυσμενείς επιπτώσεις για τη συνέχιση των ευρωπαϊκών πολιτικών στο μέλλον. Ας δούμε λοιπόν, ε, αυτό που ζητούμε εμείς είναι μια θαραλέα προσέγγιση και ε, να μην ακολουθεί η εύκολη επιλογή η Ευρωπαϊκή Ένωση να καθίσταται πάντοτε ο αποδιοπομπαίος τράγος. Πρέπει να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα, οι ελλείψεις, τα κενά και εμείς εδώ στην Ήτρη θα πρέπει να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διαρρήξουμε τα ταμπού στον ευρωπαϊκό προπολογισμό και να εξασφαλίσουμε ότι οι πολιτικοί στόχοι και ιδιαίτερα η στρατηγική του 2020 θα έχουν τη δυνατότητα να φέρουν αποτελέσματα πριν από το 2014. Δηλαδή, ήδη με τον προπολογισμό του 2011 θα πρέπει να ξεκινήσουμε. Ε, οι ευρωπαϊκές επενδύσεις θα πρέπει να κοιτούν μακροπρόθεσμα και να στηρίζονται στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, να έχουν επαρκή στήριξη δηλαδή και σε μια τέτοια χρονική στιγμή δεν μπορούμε να περικόπτουμε τις επενδύσεις ε, και ως εκ τούτου και ε, την προσθέμενη αξία που προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μια ε, συνολική λοιπόν ευρωπαϊκή βιομηχανική πολιτική για το μέλλον ε, χωρίς ε, την πολιτική για το διάστημα και το Γαλιλαίο δεν μπορεί να υπάρχει. Όπως δεν μπορεί να υπάρχει πολιτική για το μέλλον και βιομηχανική πολιτική χωρίς έρευνα και ανάπτυξη. Τι πρέπει να κάνουμε λοιπόν πρέπει οι πολιτικές προτεραιότητες της ΣΥΤΡΕ να μεταφραστούν σε συγκεκριμένε τροπολογίες στον προπολογισμό. Δύο τον αριθμό, πρώτος κύριος και σημαντικότερος στόχος, στη γραμμή όπου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει καταθέσει ικανοποιητικά νούμερα για την Ήτρε, να επαναφέρουμε τα ποσά αυτά εμείς με μία τροπολογία. Άρα εγώ προτείνω συνάδελφοι με μία γραμμή όπου το, όπου το Συμβούλιο προτείνει περικοπή σε σχέση με τις προτάσεις της Επιτροπής, εγώ να επαναφέρω τις προτάσεις της Επιτροπής στα θέματα που αφορούν εμάς, την Ήτρε δηλαδή, και στις... Ε, και στις ε, υποχρεώσεις και στις πληρωμές. Ε, δεύτερον, όπου βλέπουμε ότι χρειάζεται να προχωρήσουμε, και αυτό αφορά περισσότερο τις δεσμεύσεις, ε, σε διαφορετικά ποσά σε σχέση με την Επιτροπή, θα ήθελα να μου πείτε εσείς τι προτιμάτε. Πάντως το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο και το ανώτατο όριο του τίτλου 1α θα είναι το ε, όριο με βάση το οποίο, ο γνώμονας με τον οποίο θα προσανατολιστούμε. Εδώ έχουμε να κάνουμε μια διαφορά 50 εκατομμύρια ευρώ που ισοδυναμεί με τη θεωρητική μας δυνατότητα για εισαγωγή πολυπιλωτικών προγραμμάτων. Τώρα πρέπει να συμφωνήσουμε για τη στρατηγική και εγώ προτείνω να ξεπεράσουμε το όριο του τίτλου του 2011 γιατί με το γαριλαίο στο ε, πρόγραμμα πλαίσιο, το 7ο πλαίσιο ή της πρωτοβουλίας 2020 κτλ. Δεν μπορούμε να έχουμε προγραμματισμό ε, του, του δημοσιονομικού πλαισίου, δεν μπορούμε να περιοριστούμε δηλαδή στον προγραμματισμό του δημοσιονομικού πλαισίου και πρέπει να δείξουμε θάρρος για να ξεπεράσουμε και να στήσουμε περισσότερους πόρους. Και πρέπει Εν τω μεταξύ να αποστείλουμε ένα σεφέστατο πολιτικό μήνυμα ότι θέλουμε να διαφυλάξουμε το πρόγραμμα πλαίσιο, το 7 πρόγραμμα πλαίσιο και δεν δεχόμαστε περικοπές και ότι θέλουμε μια στρατηγική βιομηχανική στραμμένη προς το μέλλον. Και εδώ συμφωνώ με τους πράσινους συναδέλφους που λένε ότι το Έτερ και το Γαλιλαίος δεν μπορούν να αντικαταστήσουν ε, ή να απορροφήσουν το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο. Γι' αυτό θα πρέπει να πάμε να αγωνιστούμε ως Επιτροπή για τους στόχους αυτούς. Τώρα, τι δημοσιονομικά μέτρα θα μπορούσαμε να βρούμε ως λύση. Ίσως θα πρέπει να συμφωνήσουμε το Κοσλοντούι Β να χρηματοδοτηθεί για το 2011 πάνω από το περιθώριο, όχι με το μικρό αυτό ε, περιθώριο δηλαδή, γιατί το περιθώριο θα πρέπει να το χρησιμοποιούμε για τα πιλωτικά προγράμματα και τις προπαρασκευαστικές δράσεις και το Κοσλοντούι 2 να πάει ε, στο, όπως και το ίτερε ε, στο μέσον. Επίσης από τα, από τα 5 εκατομμύρια περιθώριο μπορούμε να έχουμε περίπου 120 εκατομμύρια ευρώ περισσότερα από το σχέδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις προτεραιότητές μας και για την τρομερή διάλογο. Επίσης και αυτή θα πρέπει να είναι κύριοι στόχοι μας δηλαδή το Γαλιλαίο, το ΖΙΠ, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, η ψηφιακή ατζέντα. και άλλα αντίστοιχα σημαντικά προγράμματα. Αυτά θα ήθελα να μου πείτε εσεί τι θέλετε να χρηματοδοτήσουμε από αυτά τα 120-125 εκατομμύρια. Ίσως θα πρέπει η Ήτρε να προσδιορίσει το συνολικό ποσό αυτών των προτάσεων, 10 με 15 εκατομμύρια ευρώ συνολικά και για τις τεχνικές λεπτομέρειες θα ήταν καλό να γνωρίζετε ότι έχει ανάξει το σύστημα με τη νέα συνδιαλλαγή. Υπάρχει μια ιστοσελίδα στο ίντρανετ. Μπαίνει εγχειρίδιο χειρίδιο περίπου 20 σελίδων, το οποίο λεπτομερώς περιγράφει πώς γίνεται η χρήση αυτής της διαδικασίας. Και ο κάθε ένας μπορεί να μπει στο ίντρανετ, να βάλει τις τροπολογίες του, να καταθέσει τροπολογίες του. Ε, τις οποίες μπορεί να βλέπει ο κάθε ένας εξημών και είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι η τελευταία προθεσμία είναι 18 Αυγούστου για την κατάθεση των τροπολογιών, καταλεκτική προθεσμία είναι 18 Αυγούστου. Και εν τέλει, συνάδελφοι, θα ήθελα να πω ότι η διαδικασία είναι συναπόφαση και ο εκ του το Κοινοβούλιο έχει μίζωνα βέβαια δικαιώματα, εξουσίες, αλλά πλειοψηφία δεν έχει. Άρα δεν μπορούμε χωρίς εκείνου που κάθονται εδώ στα πίσω έδρανα και οι οποίοι θα πρέπει να επιστρέψουν στις πατρίδες τους, στι πρωτεύουσε και να πείσουν τις κυβερνήσεις τους, γιατί πρέπει να ε, πείσουμε το Συμβούλιο για να μια πολιτική η οποία θα μας πάει μπροστά στον 21ο αιώνα και όχι πίσω στον, 20, ε, στον 20ο. Ευχαριστώ, λέει ο κύριος κύριο ροιλ Θα είναι πράγματι σκληρή συζήτηση. Ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ήδη στην Επιτροπή μου είμαι τακτικό μέλος, μίλησα στην ΑΦΚΟ, την συνταγματική και θα σας πω τα ίδια. Γιατί διαπιστώνω ότι οι ίδιες αρχές ισχύουν ή δεν ισχύουν ή δεν εφαρμόζονται θα πρέπει να είμεθα υπέρ της, των περικοπών στον προπολογισμό not, uh, για να δείξουμε αλληλεγγύη με τις κυβερνήσεις. Ποιος όμως θα αποφασίσει. Θα πρέπει να αποφασίσουμε όχι τώρα θα περικόψουμε ή όχι, αλλά το πού θα γίνουν οι περικοπές. Να ποια είναι η επιλογή διότι έχουμε ένα σωρό προτάσεις για περικοπές και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από το Συμβούλιο. Επομένως, Εμεί θα πρέπει να αποφασίσουμε πού δεν θα γίνουν περικοπέ. Μια υπάρχουν τόσε προτάσει για περικοπέ, αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο αφορά και την Ήτρε. Και θα πρέπει να δούμε ότι εδώ ο σκοπό είναι να κατοπολμήσουμε την κρίση. ο δικός μας προπολισμός γενικά δεν θα πρέπει να περικοπεί. Αυτό το μήνυμα πρέπει να στείλουμε. Βέβαια μπορεί να αλλάξει το μήνυμα. Και να δούμε τι γραμμή πλέψη θα ακολουθήσουμε. Τώρα όσον αφορά τις προτάσεις αύξησης του προϋπολογισμού, Εκεί θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ αυστηροί, θα πρέπει να είναι πολύ καλά τεκμηρωμένες τέτοιες προτάσεις. Το ίδιο πρέπει να και με τις περικοπές. Γενικά, συμφωνώ με την εισηγήτρια. Τα επιχείρηματά της είναι κρυστάλλινα, τα διάλεξε με προσοχή και άρα θα πρέπει να δώσουμε τη μάχη για τον προπολογισμό της ε, Ήτρε. Το μήνυμά μας είναι ότι εμείς θα πούμε όχι στις προτάσεις περικοπών της ε, Κομισιόν. Γενικώ και με εξαίρεση κάποια κονδύλια πολύ προσεκτικά επιλεγμένα. κάποιες διοικητικές δαπάνες, ίσως προτάσεις οικονομίας. Επομένως, συμφωνώ με την πρόταση της συζητήτριας να δοθεί αυτή η μάχη, είναι γνωστή η κατάσταση, αλλά προσοχή για τα προηγούμενα που δημιουργούμε δημιουργούν προηγούμενα κατά αυτόν τον τρόπο και ελπίζω να μην επαναληφθούν τα προηγούμενα με τον επόμενο προπολογισμό. Γιατί τώρα έχουμε συγκεκριμένε περιστάσει. Άρα δεν θα περικόψουμε κονδύλια πέραν της προσπάθειας να καταπολεμήσουμε την κρίση. Ε, κατά κάποιο τρόπο αυτό είναι, ε, να το πω και διπλωματικά, είναι, είναι, είναι λαϊκίστικο εγχείρημα. επόμενο. Λυπηρό είναι βέβαια σε τέτοια οικονομική κρίση να περικόπτουν τα κονδύλια από τα οποία περιμένουμε και τη μεγαλύτερη απόδοση, δηλαδή το πρόγραμμα πλαίσιο που φαίνεται να περικόπτεται κατά 35%. Πρέπει λοιπόν να γίνει μια συζήτηση σοβαρή για τις συνθήκες αυτών των περικοπών, διότι δεν μπορούμε να εξασφαλίσουμε ούτε φορεία ούτε οικονομική ανάπτυξη με τέτοιου περικοπές. Και ίσως το δημοσιονομικό πλαίσιο που έχει μακροπρόθεσμα να εξασφαλιστεί, να συμφωνήσουμε, να τηρείται και οι νέες δαπάνες που προκύπτουν, που απαιτούν περισσότερα νέα κονδύλια να συζητήσουμε πώς θα βρούμε τα κονδύλια, πού θα από πού θα τα χρηματοδοτήσουμε. Δεν δέχομαι όμως το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο ή άλλα σχέδια ή προγράμματα να περικόπτονται μαζικά. Χρειάζεται διαφάνεια. Μια άλλη παρατήρηση. Η προπαρασκευαστική δράση και για το low carbon refurbishment όσον αφορά τη δική μας επιτροπή απαιτείται να αναλυφθεί αυτή η πρωτοβουλία γιατί μην ξεχνάμε ότι υπάρχει μέρος του, των λαών μας που δεν έχουν τους πόρους να κάνουν την αναμετατροπή έτσι ώστε να φτάσουμε στα ποσοστά που επιδιώκουμε με το zero energy κτλ. Ίσως λοιπόν για μικρά σπίτια και μικρά διαμερίσματα θα μπορούσαμε να δώσουμε λύσεις διαφορετικές. Έχουμε με την τροπολογία 2 στην έκθεση Van Brent την την οικονομική υποστήριξη στον τομέα της ενέργειας και νομίζω ότι αυτό αντιστοιχεί σε αυτό το στόχο ε, έτσι ώστε να αναπτυχθεί ένα τέτοιο σχέδιο το οποίο θα έχει θετικές, θετικό αντίκτυπο. Επίσης το Εράσμους για τους επιχειρηματίες και τους δημοσιογράφους είναι χρήσιμο πιστεύω έτσι ώστε να προβληθεί περισσότερο η Ευρωπαϊκή Ένωση στο κοινό και ευχαριστώ εδώ πέρα και την εισηγήτρια, τη διαβεβαιώνω για την πλήρη μου υποστήριξη. Ασφαλώς Οφελεί τα συμφέροντα της Επιτροπής μας να προχωρήσουμε σε αυτές τις προτάσεις. Ευχαριστώ κυρία Νίπλερ. Ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ την εισηγήτρια. Ήταν ε, η ανάλυση της σαφής και εμπεριστατωμένη. Δεν θέλω να αφαιρθώ σε δύο σχέδια τα οποία με ενδιαφέρουν ιδιαίτερως και σχετίζονται και με την συζήτηση για την απλούστευση, τα αναφέραμε και νωρίτερα, το ίτερ και το Γαλιλαίο. Πρέπει να είμαστε σαφείς εάν τα θέλουμε ή όχι. Εάν τα θέλουμε λοιπόν αυτά τα σχέδια και πιστεύω ότι η ευρύτατη πλειοψηφία εδώ στο Κοινοβούλιο τα υποστηρίζει, θέλουμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση να συμμετέχουμε στο ΙΤΕ και θέλουμε και το σύστημα Γαλιλαίος ως δικό μας δορυφορικό σύστημα πλοήγησης θέλουμε να τον αναπτύξουμε. Άρα θα πρέπει στη συνεργασία με τα κράτη-μέλη και βέβαια με την εισηγήτρια να εξασφαλίσουμε τη χρηματοδότησή τους. Για το Γαλιλαίος έχουμε συζητήσει επί μακρόν και υπενθυμίζω ότι είχε τεθεί το ζήτημα να καταστεί διακρατικό εγχείρημα ή μόνο ευρωπαϊκό το Γαλιλαίος. Και εμείς είχαμε πει ως Κοινοβούλιο ξεκάθαρο ότι πρέπει να είναι μόνο ευρωπαϊκό εγχείρημα και γι' αυτό χρειάζεται και ευρωπαϊκή χρηματοδότηση και επίσης η έρευνα για τη σύνδεξη, ενεργειακή έρευνα, το Γαλιλαίος είναι ε, διαστημική έρευνα. Δεν μπορούμε λοιπόν ε, να πούμε ότι δεν έχουν θέση στο 1α. Παρακαλώ να επιμείνουμε να μην υπάρξει αποδοχή ασδήποτε περικοπής, να μην υπάρξει αλλαγή στην υπαγωγή στο 1α και να αφήσουμε ένα περιθώριο για την ουσιαστική εξασφάλιση τη ε, χρηματοδότηση των κονδυλίων των προγραμμάτων αυτών. Δεν ξέρω τα κράτη-μέλη τι θέση έχουν ω προς τη χρηματοδότηση των δύο αυτών ε, σχεδίων. Ίσως να σκοπεύουν να την εγκαταλείψουν 100% πράγμα το οποίο είναι απαράδεκτο φυσικά. Είχαμε δει και στο παρελθόν, είχαμε προσπαθήσει παραδείγματι να βρούμε τα κονδύλια από άλλες κατηγορίες όταν είχαμε προβλήματα ως προς τους σπόρους, στο Γαλλιός, αν δεν θυμάμαι, αν καλά, ε, είχε χρηματοδοτηθεί από την κατηγορία 5 και σε ένα βαθμό από γεωργικά κονδύλια που με κάποιο τρόπο είχαν χαρακτηριστεί κατάλληλα για τη χρηματοδότηση του Γαλιλαίου. Ε, αυτό πρέπει να το αποφύγουμε. Πρέπει να έχει τη δική του χρηματοδότηση και είναι βέβαιο ότι ο πιο σημαντικό στόχο είναι να διαφυλαχθεί η λειτουργία των προγραμμάτων αυτών. Ω Κοινοβούλιο, εμεί έχουμε παρακολουθήσει τη διαχείριση του προγράμματος. Μάλιστα για το ITER, για το είχαμε και μία μια παρουσίαση που αποδεικνύει ότι είχε καλά αποτελέσματα, έχει λειτουργήσει ικανοποιητικά. Και παρακαλώ να ασχοληθούμε εντατικά με τα θέματα αυτά στην Επιτροπή μας και πώς προχωρούν τα ε, σχέδια και ποια είναι η αποτελεσματικότητά τους. Αποτελεσματικότητα και ως προς το κόστος και ως προς την παραγωγή αποτελέσματος. Ευχαριστώ κυρία Έκα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ την εισηγήτρια. Σαφέστα τις πληροφορίες που δίνει και τοποθέτησή της επίσης. Υποστηρίζω τις απόψεις της όσον αφορά το ίτερ. Λοιπόν, δεν μπορεί να τριπλασιάσει κανένα πρόγραμμα του, το, να τριπλασιάσει τα το κονδύλια του. Το θέμα δεν είναι να σταματήσει ή να συνεχίσει το πρόγραμμα. Θα πρέπει να τηρήσει τα, τον προπολογισμό που, να συμμορφωθεί τον προπολογισμό που έχει αποφασιστεί. Αν δεν μπορεί να γίνει αυτό θα πρέπει να επανεξεταστεί το θέμα. Δεν δίδεται επιταγή εν λευκό για τα πάντα μια απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή μια απόφαση δημοσιονομική στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θυμηθείτε τη συζήτηση που είχαμε πριν από δεκάλεπτο για τα ερευνητικά προγράμματα και πώς προσπαθούμε να τα ελέγξουμε και πώς μπορούμε να ελέγξουμε επιστήμονες ή γεωργούς ή μικρομεσές επιχειρήσεις. Ένα ερευνητικό πρόγραμμα σαν και αυτό θα πρέπει να μείνει εντός προϋπολογισμού. Διαφορετικά δεν θα γίνεται σεβαστή αδίποτε απόφαση περί προπολογισμού του Κοινοβουλίου. Και δεν είμαι έτοιμη ακόμα να πω όχι στο ίτερ, αλλά είμαι έτοιμη να υποστηρίζω τους δημοσιονομικούς κανονισμούς και για αυτό το πρόγραμμα. Θα μπορούσα να τα πω πιο χοντρά, αλλά σε εγώ με τον πρόεδρο. η συντριπτική πλειοψηφία υποστηρίζει τις προτεραιότητες του ψηφίσματος για την Ευρωπαϊκή Ένωση του 2020 που ψηφίστηκε πριν από 15 μέρες. Είναι πολύ καλό το ότι η συγγήτρια θέλει να γίνει σεβαστή και αυτή η απόφαση. Πρέπει να επενθυμίσουμε και στα κράτη-μέλη και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι υπάρχει η κρίση και ότι χρειάζεται κάτι να κάνουμε για να βγούμε από αυτή και ότι ο προπολογισμό είναι ένα πάρα πολύ ζωτικό εργαλείο για κάτι τέτοιο. Αν δείτε κάποιε από τι Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα δείτε ότι δεν ευθυγραμμίζονται με τη στρατηγική Ευρωπαϊκή Ένωση του 2020. Αντιθέτω, είναι σχεδόν αντίθετε με κάποιε από τι πολιτικέ που συμφωνήσαμε στον τομέα αυτό. Θα πρέπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση να μπορέσουμε να εξετάζουμε ποιες είναι οι διασυνδέσεις διαφόρων τομέων ε, πολιτικής και ανάμεσα σε αποφάσεις που έχουμε πάρει. Ε, κυρία Γαστίγιο, για να μην επαναλάβω πολλά από τα πράγματα που υπόθηκαν, πρώτα απ' όλα θα ήθελα να συγχαρώ την εισηγήτρια, διότι τα εξήγησε πάρα πολύ καλά και βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου όπως αναφέρθηκε, εξετάζουμε το θέμα της ε, προσαρμογής του πλαισίου. Αντί του να ζει κανείς ή να μην ζει του Σέξπιρ, είμαστε στο να περικόψει κανείς να μην περικόψει. Αυτό είναι το δίλημα. Ε, αναφέρθηκε το θέμα της συναπόφασης και εφόσον ακολουθούμε τη διαδικασία της συναπόφασης, έχουμε πραγματικά τη δυνατότητα να επηρεάσουμε τα αποτέλεσμα. Και για να το κάνουμε αυτό βέβαια, για να επηρεάσουμε τα αποτέλεσμα, ε, πρέπει να λάβουμε κάτι υπόψη που είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι θα πρέπει να, είμαστε, να είναι όσο πιο, δυνα, πιο συνενετική η θέση στην οποία θα καταλήξουμε, να συμφωνούν οι περισσότεροι. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα πρέπει να έχουν μια κοινή θέση όλες οι πολιτικές ομάδες, διότι αυτό θα επηρεάσει τα αποτελέσματα στη διαδικασία της συναποφάσεως. Και υπάρχει και κάτι άλλο που είναι πάρα πολύ σημαντικό και θέλω να αναφέρω, βλέπω πολλούς τομείς όπου μπορούν να γίνουν περικοπές. Αλλά δεν θέλω να με κυνηγήσουν συνάδελφοι από άλλες επιτροπές, αλλά κάτι μου έρχεται στο μυαλό όταν το σκέφτομαι το θέμα. Όμως εδώ είμαστε ακριβώς στο επίκεντρο του θέματος. Η Ήτρε αφορά βασικά θέματα για να ξεφύγουμε από την κρίση, αλλά και πέρα από αυτό, ούτω ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να μπορεί να είναι ανταγωνιστική οικονομικά στο παγκόσμιο προσκήνιο. Αυτά είναι θέματα με τα οποία ασχολείται η Ήτρε. Και αυτό θα πρέπει να είναι το βασικό επιχείρημα που θα χρησιμοποιείτε. Δεν μπορούν να γίνουν περικοπέ στο ίτερ και σε άλλα προγράμματα. Θα πρέπει να εξεταστεί η χρηματοδότησή του βέβαια και ε, η διαχείριση των ποσών που διατίθεται, αλλά δεν θέλουμε υπονομεύσουμε την συνέχεια των προγραμμάτων αυτών εις βάρος του προγράμματος πλαισίου ή εις βάρος της ανταγωνιστικότητας. Αυτό πρέπει να κάνουμε πρώτα απ' όλα είναι να είμαστε σίγουροι ότι έχουμε κοινή και ομόφωνη θέση όσον αφορά τα προγράμματα ITER και δεύτερον να τονίσουμε ε, τον σημαντικό παράγοντα. Ότι αυτά είναι προγράμματα για το μέλλον της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης των διαφόρων κοινών προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από αυτό το κοινό προπολογισμό. Είναι βασικά πολιτικές με τις οποίες ασχολείται η Επιτροπή μας, εκτός από κάποιες. Και αν περικοπεί η χρηματοδότησή τους δραστικά, δεν θα έχουμε κοινέ ευρωπαϊκέ πολιτικέ που μπορούν να επηρεάσουν τη μελλοντική ανάπτυξη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να επενθυμίσω δύο πράγματα όσον αφορά το ΙΤΕΡ. Εγώ θα ήθελα να πούμε ότι υπάρχει μεγάλη υποστήριξη ευρωπαϊκή για το ΙΤΕΡ. Είδα μια απόφαση του Συμβουλίου χτε ότι τα κράτη-μέλη δεν θέλουν να προσθέσουν χρήματα. Αυτό είδα. Υποστηρίζουμε αλλά δεν προσθέτουμε χρήματα. Λοιπόν, ο υφιστάμενος υπολογισμό και το εκτελεστικός κλάδος πρέπει να χρηματοδοτήσει. Άρα πρέπει να σχετικοποιούμε τα πράγματα όσον αφορά την υποστήριξη των κρατών μελών προς το ΙΤΕΡ. Όχι την ιδέα του ΙΤΕΡ, αυτό που έγινε το πρόγραμμα με αυτόν τον προπολογισμό και το κόστος του. Δεύτερον, εγώ θα έλεγα ότι η πολιτική ευθύνη ε, δεν είναι κάτι που παραμένει μόνο στην αρχή όταν υποστηρίζεται ένα πρόγραμμα, αλλά κατά τη διάρκεια ζωή του προγράμματο. Είναι η δική μα πολιτική ευθύνη από τη στιγμή που το πλαίσιο άλλαξε εντελώ. Είναι αυτό τη ε, χρηματοδοτική κρίσεω, δημοσιονομική κρίσεω των κρατών, τη ενεργειακή κρίσεω, τη κλιματική κρίσεω, που δεν, είναι στο δεν ήταν στο επίκεντρο τη επικαιρότητα όταν ε, βγήκε το ίτερ μετά από τον ψυχρό πόλεμο, όταν βγαίναμε από τον ψυχρό πόλεμο. Άλλαξε το πλαίσιο και είναι πολιτική μας ευθύνη να επαναξιολογήσουμε αυτό το πρόγραμμα βάσει των αναγκών, συναρτήσει των αναγκών της Ευρώπης, συναρτήσει των ανάγκης εξόδου από την κρίση για τη δημιουργία θέσης απασχόλησης και ε, τις προσπάθειες που χρειάζεται να βγούμε από την κλιματολογική κρίση ε, και την ενεργειακή κρίση. Χρειάζεται επαναξιολόγηση λαμβάνοντας υπόψη αυτές τις ε, διάφορες πτυχές. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Η Επιτροπή έχει στήσει να λάβει σύντομα το λόγο, δεν ξέρω ποιο από εσά, αλλά παρακαλώ πολύ σύντομα γιατί έχουμε πίεση χρόνου πλέον. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εκμεταλλεύουμε την ευκαιρία της συνεδρίας αυτής να υπενθυμίσω ότι οι πιστώσει πληρωμών ζητήθηκαν από τον προϋπολογισμό, για το σχέδιο προϋπολογισμού 2011 και το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο και είναι κονδύλια που προβλέπονται και για περιοδικές πληρώμες για υπάρχουσε υπάρχουσες συμβάσεις και για προχρηματοδοτήσεις για τις νέες συμβάσεις που θα υπογραφούν το 2011. Εάν οι περικοπές του Συμβουλίου, οι σημαντικές περικοπές υλοποιηθούν, αυτό θα έχει διτή συνέπεια. Πρώτα απ' όλα θα υπάρχει σημαντική καθυστέρηση των περιοδικών πληρωμών, των συμβάσεων που ήδη είχαν υπογραφεί από το 2007 μέχρι σήμερα και συνέπεια για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα είναι ότι θα, έχει πολλά, θα πληρώσει πάρα πολλά, πολλούς τόκους ε, για καθυστερήσεις πληρωμών 2011-2013 και περικοπές θα έχουν συνέπεια όσον αφορά την υπογραφή συμβάσεων ερευνητικών ε, για το 2011 με υποχρεώσεις που είχαν ληφθεί για το 2011. Η υπογραφή αυτών των συμβάσεων θα πρέπει να καθυστερήσει εθελοντικά για να μετατεθεί η προχρηματοδότηση για το 2012. Οπότε οι αιτήσει για το σχέδιο προπολογισμού του 2012, μάλλον οι απαιτήσει του σχεδίου προπολογισμού του 2012 ε, θα είναι πάρα πολύ αυξημένε. Και αυτό θα έχει συνέπειε και για την έρευνα. Ε, και δεν βοηθούν όλα αυτά την οικονομική ανάκαμψη. Θα δώσω το ε, λόγο τώρα στη Διευθυντή της Υπηρεσίας ΡΕΑ για την έρευνα για να αναφέρω κάτι που τόνισε και ο συνάδελφος. Αυτό που προτείνεται είναι 11% περικοπή στις πιστός πληρωμών για τις δράσεις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτό είναι αρκετά κακό. Θα μπορούσαμε να τα καταφέρουμε μέσω καθυστερήσεως της, της υπογραφής των ε, συμβάσεων και να μειώσουμε την ε, προχρηματοδότηση. Για να απορροφήσουμε αυτές τις περικοπές ε, θα πλήξουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και αυτού του είδους οι πελάτες δεν μπορούν να αντέξουν έτσι καθυστερήσεις των πληρωμών. Όμως, επίσης προσέξτε και το εξής. Υπάρχει μικρότερη περικοπή του 5,5 εκατομμύρια για διοικητικές δαπάνες για την υπηρεσία μου που χειρίζεται τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις αλλά αυτό είναι το 15% του ε, διοικητικού προϋπολογισμού της υπηρεσίας μου. Μέχρι τώρα μειώναμε τον χρόνο για να εγκρίνουμε προγράμματα και για να πληρώσουμε. Αν αυτή η περικοπή τελικά υλοποιηθεί, όχι μόνο δεν θα μπορώ να προσλάβω προσωπικό για να χειριστεί τα περισσότερα χρήματα που θα έχω του χρόνου, αλλά να απολύσω προσωπικό, διότι δεν θα μπορέσω να πληρώσω τους μισθούς του χρόνου. Εάν δεν μπορώ να κρατήσω το προσωπικό μου, όταν υπάρχει μεγάλη ανάπτυξη και αύξηση στον ετήσιο προπολογισμό, ξεχάστε κάθε στόχο όσον αφορά το πότε θα εγκρίνονται προγράμματα και πότε θα καταβάλλονται τα χρήματα. κυρία Έκαρτ, σύντομη παρακαλώ, οι συνέπειες λοιπόν που αναφέρθηκαν είναι πάρα πολύ σοβαρές και θα ήθελα να ζητήσω από την γραμματεία να περιγράψει γραπτό την κατάσταση για το ίτερ σε συνδυασμό με τις περικοπές του προπολογισμού και με όσα μας περιέγραψε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή του στα μέλη της Επιτροπής να τα έχουν όλα αυτά μπροστά τους γραπτός για να τα λάβουν υπόψη όταν θα συζητήσουμε τα διάφορα ζητήματα. Καλώς λάβαμε την πρόταση κύριε Χέρτσκοκ και παρακαλώ πολύ στόμα γιατί Έχουμε μόνο μισή ώρα για το τελευταίο σημείο στην ημερήσια διάταξη που επίση έχει μεγάλη σημασία. Παρακαλώ κυρία Χέρτσοκ. Ναι πρόεδρε, πολύ σύντομα. Αναφερθώ σε διάφορα θέματα όσον αφορά τα κονδύλια. Έχουμε ετοιμάσει όλους τους πίνακες, μπορούμε να τους αποστείλουμε. Μπορούμε να προχωρήσουμε. Δεν θα αναφερθώ σε όλες τις ερωτήσεις, δεν έχω χρόνο. Προς την κυρία Εκ να πω στον τομέα της έρευνας, αν καθυστερήσει το πρόγραμμα, τριπλασιάζεται το κόστος. Συμβαίνει αυτό. Το ίδιο θα γίνει και με το Γαλιλαίο. Αν δεν δοθούν τα 500 εκατομμύρια φέτος, εντάξει. Καθυστερήσει, αλλά του χρόνου θα είναι ένα δισεκατομμύριο ή παραπάνω το κόστος για να παραγγελθούν τα διάφορα μηχανήματα και τα ανταλλακτικά. Δεν είναι σαν να αγοράζει κάτι από την υπεραγορά. Εκρήγνεται το κόστος και σχετίζεται με κακέ αποφάσει όσον αφορά τον προπολογισμό, χρονισμό, καθυστερήσει. Και γι' αυτό είμαστε κατά. Όσον αφορά το ITER, το ITER δεν θα ισχύσει το 2000, για τον προπολογισμό του 2011. Δεν είναι άμεση πληρωμή. Πρέπει να είμαστε ενωμένοι. Διότι ετοιμαζόμαστε για το νέο δημοσιονομικό πλαίσιο και πρέπει να είμαστε πολύ ξεκάθαροι στο τι θέλουμε. Συμφωνώ πλήρω με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τι είδαμε στο έγγραφο του Συμβούλιο όσον αφορά την τροποποίηση του προπολογισμού. Περιέκοψαν το, τις δαπάνες για το management, για τη διαχείριση. Αν δεν αλλάξει τους κανόνες, ισχύουν οι κανόνες, αλλά η εφαρμογή των κανόνων αλλάζει λόγω περικοπών. Και είναι βάρος των προγραμμάτων. Οι συνέπειες μπορεί να είναι τεράστιες. Γι' αυτό συμφωνούμε ότι πρέπει όλα αυτά τα κονδύλια να αποκατασταθούν παρόλο που είναι διοικητικό κόστος, φαίνονται σε διοικητικό κόστος. Δεν μπορούν να λειτουργήσουν οι υπηρεσίες εάν γίνουν αυτές οι περικοπές. Πρέπει να είμαστε ενωμένοι, πρέπει να στείλουμε πολύ ισχυρομένοι στο το Συμβούλιο ότι στη διαδικασία συναπόφασης εμείς θα πολεμήσουμε προς όφελος όχι της Επιτροπής Βιομηχανίας αλλά προς συμφέρον της Ευρώπης. Συμφωνώ με αυτά που είπε και ο Ζούμπιχ και άλλοι. Εμεί θέλουμε να είναι ανταγωνιστική Ευρώπη και θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί το δέον δημοσιονομικό εργαλείο και να μην το σκοτώσουμε. Ευχαριστώ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρέπει επίση να ε, λέει ότι θέλει να λάβει τον λόγο, αλλά άρα είναι απολύτω απαραίτητο αν έχετε κάτι καινούργιο να μα προσφέρετε φυσικά. Κοιτάξτε, θα ήθελα να μιλήσω εκ μέρους του Ευρω... της εκτελεστικής υπηρεσίας του Ευρωπαϊκού Συμβούλιου Ερεύνας. Στην πρώτη προπολογισμού που είδα, εμείς είμαστε στόχος των μεγαλύτερων περικοπών, 100 εκατομμύρια επιστώσεις πληρωμών. Και το Ερευνητικό Συμβούλιο είναι μία από τις επιτυχίες του 7ου προγράμματος πλαισίου. Θα καταστραφούμε τώρα εάν γίνει αυτή η περικοπή. Δεν θα μπορέσουμε ακόμα να αναλάβουμε νέε υποχρεώσει με αυτά τα χρήματα, διότι καθυστερούμε πάρα πολύ την εκτέλεση του προπολογισμού. Απευθύνω έκκληση. Κοιτάξτε, έχουμε προγράμματα που ίσως δώσουν τις λύσεις όλα τα σημερινά προβλήματα και αν γίνουν οι περικοπέ, οι θετικέ εξελίξει θα σταματήσουν. Και αυτό θα είναι πάρα πολύ μεγάλη καταστροφή για μα αν γίνει αυτή η περικοπή σημαντική. Αυτά ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ, Λεπρόεδρο. Νομίζω ότι για τα θέματα αυτά δεν μπορούμε να προχωρούμε αν ο καθένα προεξαγγέλει καταστροφέ για το θέμα που τον ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Όχι, πρέπει να συμβάλλουμε στο να αποφεύγονται οι καταστροφέ. Είναι κάτι πολύ δύσκολο και συγχαίρω του συναδέλφου που επεξεργάζονται το θέμα αυτό. Πρέπει να κάνουμε τη δουλειά μα με προσοχή και το Κοινοβούλιο βέβαια και η Επιτροπή, αλλά και το Συμβούλιο πρέπει να συμβάλλει. Ζητώ συγγνώμη που πιέζω. Έχουμε όμως ακόμη το θέμα του σχεδίου δράσης για την αργιακή απόδοση. Ο κύριος Μπέντσεν, ο συντάκτης της έκθεσης πρωτοβουλίας, με πολλή υπομονή, παρακολούθησε όλες τις σημερινές συζητήσεις. Ήρθε η ώρα να ακούσουμε τι έχει να μας πει. 18 Αυγούστου είναι η προθεσμία για την κατάσταση τροπολογιών για το θέμα αυτό το τελευταίο στη μερίσια μας διάταξη. Παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καταρχάς θέλω να ευχαριστήσω τους και ηγητές. Πάρα πολύ καλή ήταν η συνεργασία μας. Και μετά συνεχίσω στη μητρική μου γλώσσα μετά την αγγλική. Έχουμε να κάνουμε μια πολύ σημαντική υπόθεση. Μπορούμε να κάνουμε κάτι για την Ευρώπη. Ζούμε σε ένα παγκοσμιοποιημένο κόσμο. Εξαρτόμαστε και από τη δυνατότητά μας να ανταγωνιστούμε σαν Ευρώπη. Είναι σημαντικό λοιπόν να φροντίσουμε ούτω ώστε η ενέργεια να μπορεί να συμβάλλει ε, στην προστασία και του περιβάλλοντος και στην ανταγωνιστικότητα. Όταν μιλάμε για ανταγωνιστικότητα και για το κλίμα θα πρέπει να θεωρήσουμε ότι η ενεργειακή απόδοση θα πρέπει να έχει νέα θέση, η ενεργειακή αποδοτικότητα, σημαντική θέση. Εμείς εισάγουμε πετρέλαιο ε, από άλλες χώρες. Αυτό που θα πρέπει να κάνουμε είναι να προσπαθήσουμε να βρούμε νέες πηγές ενεργειακές αλλά και να προσπαθήσουμε να εξοικονομήσουμε ενέργεια και να βελτιώσουμε την αποδοτικότητα. Είναι σημαντικό όταν δισεκατομμύρια ευρώ διατίθεται στην Ευρώπη να, να τα χρησιμοποιήσουμε ή να βοηθήσουμε τον καταναλωτή αλλά και να βοηθήσουμε να υπάρχει μεγαλύτερη ενεργειακή αποδοτικότητα. Αυτές οι οικονομίες μπορεί να είναι πάρα πολύ σημαντικές για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης. Είναι σημαντικό να μιλάμε όλοι με κοινή φωνή, το Συμβούλιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Κοινοβούλιο όσον αφορά το θέμα αυτό. Πιστεύω ότι όταν μιλάμε για τυποποίηση θα πρέπει να είμαστε πιο αποφασιστικοί στο συγκεκριμένο τομέα. Μεταξύ άλλων είναι σαφές ότι θα πρέπει να προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε τη δουλειά που κάνουμε όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση. Θα πρέπει να πετύχουμε το στόχο που είχαμε καθορίσει για το 2020. Για αυτό θα μας βοηθήσει να δημιουργήσουμε θέσεις απασχόλησης και να βοηθήσουμε και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η χώρα μου διπλασίασε το ΑΕΠ ε, κυρίως μέσω της, του ενεργειακού τομέα, σε σχέση, εν συγκρίση με αυτά που κάναμε πριν από δεκαετίες, έγιναν πολλές παρεμβάσεις σε διάφορους τομείς, στις διάφορες περιφέρειες. Πρέπει να κάνουμε περισσότερα όμως, διότι υπάρχει μετά κέρδος. Μία επένδυση στην ενεργειακή αποδοτικότητα αποσβαίνεται μετά από δύο μέχρι πέντε χρόνια και δίνει κέρδη. Αυτό είναι σημαντικό να το έχετε υπόψη. Εγώ πιστεύω ότι η έκθεση θα πρέπει να περιγράφει ε, τι πόροι διατίθεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να υπάρχει καλύτερη υλοποίηση των ιδεών που υπάρχουν. Όχι διότι δεν αποφασίζονται σωστά πράγματα στην Ευρώπη, όμως μετά χρειάζεται σωστή εκτέλεση, σωστή εφαρμογή στα κράτη-μέλη όλων αυτών των ιδεών και των αποφάσεων. Διαβάζοντας το σχέδιο δράσης για την ενεργειακή απόδοση βλέπω ότι υπάρχουν κάποιες παράγραφοι, υπάρχουν κάποια παραρτήματα με πάρα πολλές προδιαγραφές και διατάξεις που θα πρέπει να εφαρμόζονται. Είχαμε το 2007, 2008, 2009, 2010. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να είμαστε πολύ προσεκτικοί θα πρέπει στην πράξη να ε, εφαρμόζεται αυτό που ε, αποφασίζουμε. Χρειάζεται και επίσης και μια αναθεώρηση της Energy Service Directive, της οδηγίας και τις ενεργειακές υπηρεσίες και θα πρέπει επίσης να ε, εξετάσουμε και το τι γίνεται με το θέμα της θέρμανσης εξ αποστάσεως και να αφορμόσουμε και την οδηγία για την ετικετοθεσία, την Energy Labeling Directive θα πρέπει να συζητήσουμε την εξοικονόμηση ενέργειας που μπορεί να προκύψει και από μια προσαρμογή και ε, των υφιστάμενων οικοδομών και θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και την ε, ποσότητα των παλιών οικοδομών, τον αριθμό των παλιών οικοδομών και πως αυτή η προσαρμογή των παλαιών κατοικιών μπορεί να οδηγήσει σε δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης. Μπορούμε να δημιουργήσουμε μια αγορά, πιστεύω. Ε, αναφέρομαι και στις ε, δημόσιες αγορές smart metering, smart risk για τους ευφυείς μετρητές κλπ. Χρειάζεται περισσότερη δράση, χρειάζεται καλύτερη εκτέλεση, καλύτερη εκτέλεση των ιδεών και υλοποίησή τους και να υπάρχει και υψηλότερο ποσοστό υλοποίηση των ιδεών και στις μεταφορές. Και εκεί θα πρέπει να υπάρχει περισσότερη καινοτομία για τα μεταφορικά μέσα. Να είναι πράσινα τα μεταφορικά μέσα που χρησιμοποιούνται. Πιστεύω λοιπόν ότι η ενέργεια χρησιμοποιείται σε πάρα πολλούς τομείς και μπορούμε να κάνουμε πολλά για το μέλλον στο οικονόμηση ενέργειας. Το θέμα είναι ότι μας λείπει ε, η χρηματοδότηση. Θα πρέπει να επαναξετάσουμε τα διαθωτικά μας ταμεία. Ε, είναι σημαντικό επίσης να υπάρχει πρόσβαση και στο ιδιωτικό κεφάλαιο για αυτή την προσπάθεια. Πάνω απ' όλα για τις επιχειρήσεις μας, οι οποίες επιχειρήσεις έχουν μείνει πάρα πολύ πίσω όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα που συζητάμε. Είναι απαραίτητο λοιπόν να υπάρξουν επενδύσεις και από τον ιδιωτικό τομέα, μεταξύ άλλων, όπως είπα, σε δύο-τρία χρόνια θα υπάρχουν κέρδη και αποσβηση των επενδύσεων και μετά θα υπάρχει και κέρδη. Μπορούμε με κάποιες εγγυήσει να βοηθήσουμε την ανάπτυξη αυτού του τομέα και τις εξελίξεις. Σε αυτό το τομέα ήταν δυνατό τον να παρέμβουμε και με ενισχύσεις, κυρίως στις ε, εταιρείε του τομέα της ενέργειας. Τώρα θα πρέπει να πληρώσουμε τους λογαριασμούς του παρελθόντος ε, λόγω ελλείψεως επενδύσεων, καταλήλων επενδύσεων στο παρελθόν. Έχουμε συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα μπροστά μας ε, υπάρχουν προβλήματα μεταφράσεως των εφόρων κειμένων κλπ. Το Σεπτέμβριο θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρουσιάσει κάτι. Μετά θα υπάρξει και μια συνάντηση στη Σύνοδο Κορυφής που θα συζητηθεί το θέμα το Φεβρουάριο. Είναι σημαντικό λοιπόν να είμαστε έτοιμοι για τότε. Ίσως αυτή η έκθεση μπορεί να έχει και κάποια επιρροή όσον αφορά το εγγύς μέλλον. Βεβαίως είναι ανοιχτή η θέση μου, περιμένω να ακούσω σχόλια και σίγουρα θα υπάρξει πάρα πολύ καλή συνεργασία μεταξύ μας ε, μέχρι ότου καταλήξουμε στο τελικό κείμενο της εκθέσεως. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Και εγώ ευχαριστώ. Μας έχουν στις έξι συναδελφοί τον λόγο και θα σας παρακαλώ όλους να είστε πολύ σύντομοι. Ας ακούσουμε πρώτα τους και οδησηγητές, αν δεν έχετε αντίρρηση. Κύριε Χόλ, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον εισηγητή. Γιατί ήταν πάρα πολύ θετική η προσέγγιση του και η συνεργασία του με τους και ηγητές και όλοι συμφωνήσαμε ότι εδώ υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλες δυνατότητες να πετύχουμε την αποτελεσματικότητα την ενεργειακή, κάτι που δεν το έχουμε καταφέρει ακόμα και άρα θα πρέπει να έχουμε στάση ανοιχτή όσον αφορά κάποιες δυνατότητες που προσφέρονται για να μπορέσουμε να προωθήσουμε την υπόθεση αυτή, κάτι το οποίο θα πρέπει να καλύπτει και το πώ μπορεί να έχουμε νομοθεσία που, που να συντείνει προσπαθίε μας από άλλου ε, τομεί και να, να, να δούμε πώς με νομοθεσία θα πετύχουμε εκεί που δεν πετύχαμε με άλλου ε, λιγότερο αυστηρού τρόπους και να δούμε πώς ε, και από την πλευρά της προσφοράς κάτι θα κάνουμε εκτό από την πλευρά προσφορά. Τι κράτα λέει ο συγκεκριτής. Να κοιτάξουμε τι προβλέπουν και διατάξει τη οδηγία για τι υπηρεσίε, να δούμε του εθνικού στόχου και ενδεχομένω ίσω μπορούμε να έχουμε και τα κράτη-μέλη κάποιου στόχου για να ανανεώσουμε τα όσα προβλέπονται, που δεν είναι ακόμα δεσμευτικά και σύμφωνα με τον εισηγητή ότι μπορούμε να πετύχουμε περισσότερα όσον αφορά ε, τα προϊόντα που αναλώνουν ενέργεια. Εκεί τελευταία έχουμε κάποια προβλήματα και να δούμε τα κράτη-μέλη τι κάνουν και έτσι το χρονοδιάγραμμα να προχωρήσει. Έχουμε κάποιους εφραγμούς σημαντικούς. Πρώτα-πρώτα τι γίνεται με την αναθεωρημένη για τα κτίρια. Χρειάζεται να υπάρχει κάποιο κυλιόμενο ταμείο, κεφάλαιο. Χρειάζονται επενδύσεις παρά το ότι αυτό χρηματοδοτείται κατά κάποιο τρόπο η ενεργειακή αποτελεσματικότητα. Χρειάζεται κάποια κατάρτιση, εκπαίδευση, γιατί πολλές φορές είναι κάποιοι τοπικοί ηλεκτρολόγοι, μάστοροι, ε, αυτοί που ασχολούνται και για να είναι πιο αποτελεσματικά τα κτίρια, χρειάζεται κατάρτιση. Συμφωνώ για τις μεταφορές, συμφωνώ για τη γεωργία, τομείς που δεν τους καλύψαμε. Και Εκεί να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε καλύτερο για την ενεργειακή αποτελεσματικότητα, να δούμε τις υπάρχουσες δυνατότητες, πώς με έρευνα και τεχνολογία θα έχουμε καινούργια προσέγγιση. Υπάρχουν επαναστατικές μέθοδοι, βελτίωση του φωτισμού γραφείων. Μέχρι 50% μπορούμε να πάμε. Αντί για καθοδικές τεχνίες και παραδοσιακούς τρόπους, να πάμε στο φωτισμό με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και είναι τεράστιο τότε το όφελος. Γιατί τραβάει πολύ ενέργεια το, ο φωτισμός. Άρα να δούμε και αυτές τις καινοτόμες προσεγγίσεις εκτός από όλα τα άλλα. Τόμσον. Και εγώ, Πρόεδρε, να ευχαριστήσω τον εισηγητή και τους σκιώδεις εισηγητές και εισηγήτρες Είναι λιθαράκι αυτό στην στρατηγική για το 2020 και για την μείωση των εκπομπών του διοξίδιου. Να τονίσουμε το ότι αυτή η αποτελεσματικότητα είναι προϋπόθεση για την επιτύχηση των στόχων του 2020. Δυστυχώς, όπως οι εκπομπές και ενώσεις πηγές ενέργειας θα πρέπει να είναι δεσμευτικός στόχος και η ενεργειακή αποτελεσματικότητα, γιατί εάν δεν κάνουμε κάτι, τότε για τους στόχους του 2020 θα πρέπει να παράξουμε περισσότερη ενέργεια, να κάνουμε μεγαλύτερε επενδύσεις, άρα και για την αποτελεσματικότητα θα πρέπει ο στόχος να είναι δεσμευτικός και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Επίσης, είπε ο ότι το πρόγραμμα δράσης για την αποτελεσματικότητα δεν εφαρμόστηκε και γι' αυτό δεν πιάσαμε το στόχο. Όχι βέβαια. Γιατί στο κοινοβούλιο τι γίνεται. Όταν οι στόχοι δεν είναι δεσμευτικοί, δεν επιτυγχάνονται. Να και άλλο ένα ώστε να είναι δεσμευτικός ο στόχος τούτος. Ποια είναι τα αντεπιχειρήματα τώρα, ότι θα είναι πολύ ακριβό αυτό, αλλά και η ανάλωση ενέργειας είναι πολύ δάπανο πράγμα. Να δούμε την κοινωνική πτυχή. Θα δούμε τι γίνεται με την ενεργειακή παινία όσον αφορά την νίκηση της στέγαση. Γιατί πάρα πολλά λεφτά πάνε εκεί. Είναι σε επίπεδο παράδεκτα αυτή η ενεργειακή παινία για τις κατοικίες. Θα πρέπει να την καταπολεμήσουμε. Είναι πολύ σημαντικό Και θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε ιδίω στα κράτη-μέλη. Τα νέα που το πρόγραμμα είναι ε, οξύτερο. Στα αυτά τα πλαίσια θα πρέπει να καλύψουμε και να εμπλέξουμε κυρίως το Ταμείο Συνοχής και τα διαρθωτικά ταμεία. Και να μην το κάνουμε αυτό σαν σύσταση, να επιμείνουμε ότι οι πόροι από εκεί θα πρέπει να επενδυθούν στην ενεργειακή αποτελεσματικότητα. αυτό να καλυφθεί και από το πρόγραμμα πλαίσιο το επόμενο και από το τρέχουν τώρα πρόγραμμα που δεν το καλύπτει, καλύπτει μόνο κάποιες μορφές τεχνολογικών εφαρμογών. Για έχουμε τους στόχους μας θα πρέπει να θεωρηθεί στόχος του 2020 η αποτελεσματικότητα. Άρα σας παραπέμπω στο ψήφισμα του Στρασβούργου. Θα προχωρήσετε για το 2020 η βοήθεια και την απασχόληση και όπως είπε και η κυρία Χόλ, ε, αυτό είναι κάτι το οποίο ε, εστιάζει την προσοχή μας στις δεξιότητες και τα είπαμε και στην Επιτροπή Απασχόλησης. Θέλουμε πράσινες θέσεις εργασίας ευρωπαϊκή χρηματοδότηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί, να πάμε σε ισοβία κατάρτιση, το κοινωνικό ταμείο μπορεί να βοηθήσει. Και κατά αυτόν τον τρόπο μπορούμε να έχουμε την καινούργια πράσινη οικονομία και να έχουμε και θέσει εργασία. Ζαντού. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όπως και οι προγραλήσαντες και εγώ να πω τι ωραία που δούλεψε ο εισηγητή και πόσο καλή και ευχάριστη ήταν η συνεργασία του με τους σκιώδες εισηγητές. Αυτή είναι μια με φιλοδοξία μας, να έχουμε μια συλλογική δουλειά για κάποιες ε, ε, εκθέσεις. Θέλω και εγώ λοιπόν στον εισηγητή να τονίσω το ότι ακόμα απέχουμε από αυτά που μπορούμε να πετύχουμε όσον αφορά την ενεργειακή αποτελεσματικότητα. Και γι' αυτό και θα συμφωνήσω με την κυρία Χόλ και την κυρία Τόμσεν ότι δηλαδή θα πρέπει να κινηθούμε προς το να είναι το 20% ή υποχρεωτικό. Γιατί μόνο έτσι και με, με πολιτική τέτοια απόφαση μπορούμε να φτάσουμε σε αυτό το οποίο θέλουμε. Και έτσι να πετύχουμε αυτό που θέλουμε τα, τα επίπεδα που θέλουμε. Και αυτό δεν είναι μόνο θέμα ε, πολιτικού αιτήματο. Το αυτό το θέλει και βιομηχανία. Αν κάθετε και διαβάσετε ε, τον Ιούνιο τι είπε το Βιομηχανικό Φόρουμ, ε, τα ηλεκτρονικά, ε, ο κατασκευαστικό τομέα, όλοι, όλοι, όλοι οι κλάδοι της οικονομίας ζητάνε να υπάρχει στόχο δεσμευτικό που να μπορεί να τους δώσει μια, μια προβολή, μια δυνατότητα του τι να περιμένουν. Επίσης, για το πώ θα πρέπει εύστοχα να γίνει η συμμόρφωση και η εφαρμογή αυτών των μέτρων. Compliance στα αγγλικά. Η αναθεώρηση τη οδηγίας όσον αφορά τις ενεργειακές υπηρεσίες είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό γιατί έτσι η Κομισιόν ε, θα αποκτήσει έναν ρόλο εποπτικό. Με όλες τις οδηγίες μπορεί να καταλάβει τι γίνεται στα κρατημέλη, τι γίνεται στους ε, οικονομικούς συντελεστές τους operators. Το είπε ο εισηγητής και συμφωνώ μαζί του. Θα πρέπει να διατυπώσουμε κάποιες προτάσεις όσον αφορά την οικονομική στήριξη και η οικονομία στην ενέργεια στην αποτελεσματική χρήση της ε, να υλοποιηθούν και να δούμε τι μπορεί να γίνει όσον αφορά τα κτίρια για να μπορέσουμε να βρούμε έναν σωστό τρόπο για να στηρίξουμε τις ε, πολιτικές της ε, ανακαίνησης των κτίριων. Πολύ σημαντικό. Να πως να συνδέσουμε τα νέα χρηματοοικονομικά μέσα με την ανακαίνιση των κτίριων. Τα είπε χτες ο κύριος Μανιέτ και άλλοι συναδέλφοι όσον αφορά την ενεργειακή παινία Ε, κοινωνικέ κατοικίε, ε, όλα αυτά τα συνδέουμε. Γι' αυτό και νομίζω ότι οι προτάσεις οι σχετικές είναι πολύ εύστοχε. Τέλος, σε σχέση με αυτά που είπε ο κύριος Μπένσαν όσον αφορά την αναθεώρηση της ε, οδηγία για την κατοθεσία την ενεργειακή, νομίζω ότι έτσι θα μπορούσαμε να έχουμε μια άλλη λύση με τον ορίζοντα του 2012 να μπορέσουμε το eco το, την οικονοτολογική ετικέτα, όλα αυτά να τα συστρατεύσουμε και να έχουμε ε, μια, μια, μια ρύθμιση για τα προϊόντα και με όλα αυτά να μπορέσουμε να αναδείξουμε μια πολιτική για τα προϊόντα ε, δυναμική και ταυτόχρονα αυτό να βοηθήσει και την συμμόρφωση και την εφαρμογή της οδηγίας και στα κρατημέλη. Οπότε έτσι έχουμε και διοικητική επιτυχία. Ευχαριστώ κυρία Εκ, αλλά παρακαλώ να είμαστε πιο σύντομοι. Ευχαριστώ. Είναι πολύ σημαντικός, πολύ σημαντικό το θέμα αυτό. Πρέπει να το λύσουμε φυσικά. Όλοι γνωρίζουμε τι σημαίνει αποτελεσματικότητα ε, ενεργειακή, απόδοση ενεργειακή. Όλοι προσπαθούμε να βρούμε καλές λύσεις. Δεν τα έχουμε πάει και τόσο άσχημα. Αλλά μας έχουν ξεφύγει πολλές ευκαιρίες στην ε, αξιοποίηση αυτής της μεθόδου εργασίας για την ενεργειακή απόδοση. Φέρει πίν. Προσπαθούμε να προχωρήσουμε στις συμφωνίες για τις ανταλλαγές ε, ε, εκπομπών, αλλά δεν τα καταφέραμε λόγω του Συμβουλίου. Και σε άλλα ζητήματα το ίδιο. Με τις επενδύσεις στην βαριά βιομηχανία που περιμένουν την απόδοσή τους σε 3, 4 και 5 χρόνια να τη δουν να ξεκινάει, τότε ίσως θα πρέπει η βιομηχανία να επενδύσει σε τεχνολογία κατά τον ίδιο τρόπο. μπορεί η απόδοση να είναι τριετής ενώ ιστορική ε, κανόνες ε, μιλούν ε, για περισσότερα διαστήματα. Νομίζω ότι και για την αντιγωνιστικότητά μας, το περιβάλλον της θέσης εργασίας, πρέπει η νομοθεσία που θα ορίσουμε να πιέζει τη βιομηχανία προς τέτοιου είδους επενδύσεις. Οι δυνατότητες είναι τεράστιες και στην Σουηδία το βλέπουμε, αλλά λίγα μόνο εργοστάσια έχουν ε, αναδιαμορφωθεί κατά τον τρόπο αυτό και βέβαια και στα νέα κράτη-μέλη όπου είναι τεράστιο το κέρδος που μπορούν να προσμένουν από τέτοιες αλλαγές. Σε πολλούς τομείς ισχύει αυτό και νομίζω ότι θα πρέπει να βρούμε στόχους φιλόδοξους για την ενεργειακή απόδοση και τα κράτη-μέλη θα πρέπει να καταλήξουν σε γενικέ απόψει για τα θέματα αυτά με αξιοποίηση τη ομοθεσία που ήδη υφίσταται αλλά και με συμπλήρωση των κενών που υπάρχουν. Είναι πολύ μεγάλη σημασία η συνεργειακή απόδοση. Πρέπει να συστήσουμε τα θέματα τη γεωργία, όλα αυτά που δεν έχουμε συστήσει μέχρι τώρα. Τι μπορούμε να κάνουμε. Τα πιστοποιητικά που αποτελούν μία δυνατότητα και εν τέλει, ναι, συζητήσαμε τον προπολογισμό και πάλι θα το συζητήσουμε. Θα κοιτάξουμε τον προπολογισμό για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ισοδύναμο παγκοσμίου πολέμου το εγχείρημα ε, εξασφάλιση χρηματοδότηση για την ενεργειακή απόδοση, παρότι κερδίζουμε σε τρία μέτωπα εάν την εξασφαλίσουμε. Εθνική δεσμευτική στόχη λοιπόν. Αυτό πρέπει να συζητήσουμε. Και εκεί πρέπει να συμπληρώσουμε τα κενά για να κερδίσουμε όπως ξέρουμε ότι μπορούμε να κερδίσουμε. Ευχαριστώ κύριο Κάρενς. Ευχαριστώ πρόεδρε. Και θέλω καταρχάς να ευχαριστήσω τον κύριο Μπέντσεν. Κάνετε πολύ καλή δουλειά. Ανακοινήσατε πολύ σημαντικά ζητήματα. Θα ήθελα να αντιδράσω σε αυτά που είπαν διάφοροι συνάδελφοι σχετικά με τους δημευτικούς στόχους. Είναι συνεχιζόμενη η συζήτηση στο Κοινοβούλιο. Διάφορες πολιτικές ομάδες έχουν διαφορετική αντίληψη ενδεχομένως όσον αφορά τους δεσμευτικούς ε, στόχους θα πρότεινα να αλλάξουμε κάπως τη συζήτηση, να μην συζητάμε τόσο πολύ κατά πόσο χρειαζόμαστε δεσμευτικούς στόχους, διότι τι λέμε μέσω δεσμευτικών στόχων, ότι θέλουμε ενεργειακή αποδοτικότητα με δόντια, θέλουμε αποτελέσματα. Α, θα πρέπει να εστιαστούμε περισσότερο στο πώς οι αδίποτε στόχοι θα ε, επιτευθούν και ποιοι πόροι που να διατεθούν για την επίτευξη των στόχων, διότι ποικίλουν οι καταστάσει στα διάφορα κράτη-μέλη. Έχουμε κράτη-μέλη τα οποία είναι πλουσιότερα, άλλα που είναι φτωχότερα, κράτη-μέλη που είναι πιο αποτελεσματικά, άλλα που είναι λιγότερο. Και πριν βρούμε ποια είναι θέση του Κοινοβουλίου, πρέπει να υπάρχουν δεσμευτικοί στόχοι. Δεσμευτικοί στόχοι, οποιαδήποτε στόχοι θα πρέπει να ταιριάζουν με ρεαλιστική χρηματοδότηση για την επιτευξή του προ όφελο όλων. Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να είμαστε δημιουργικοί. Ο κύριο Μπένσον αναφέρθηκε στα θετικά ταμεία, ίσως το Ταμείο συνοχή, είναι ενδεχόμενοι ενδεχόμενε πηγέ χρηματοδοτήσεω. Α μην συζητούμε λοιπόν αν χρειαζόμαστε ή όχι δεσμευτικού στόχου, αλλά πώ μπορούμε να του πετύχουμε του στόχου μέσω ρεαλιστικής χρηματοδοτήσεως. Και από πού θα προέρχεται αυτή η χρηματοδότηση. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Ντεκαστήγιο έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και εγώ θέλω να συγχαρώ τον συνάδελφο Μπέλσεν για όσα έκανε. Γιατί με το έργο του κατάφερε να υπάρξει μια προσέγγιση συλλογική μαζί με τους άντρους, μαζί με όλες τις πολιτικές πτέρυγες και είναι πολύ σημαντικός αυτός ο στόχος για πολλούς λόγους. Πρώτα πρώτα βασικός λόγος είναι ότι οι ενεργειακοί πόροι βρίσκονται σε σπάνιδα και επομένως αποτελεσματική λύση της ενέργειας είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεύτερος λόγος είναι ότι τώρα έχουμε το θέμα της υπερθέρμανσης του πλανήτη, οπότε και για αυτό το λόγο χρειάζεται να υπάρχει ενεργειακή ασφάλεια. Βλέπουμε επομένως ότι έχουμε συνέπειες θετικές πάσης υφής. Εγώ πάντως θέλω να τονίσω κάτι που το είπε ο κύριος Κάρνης. Το θέμα της δεσμευτικότητας. για κάποια μέτρα. Δηλαδή, θεωρούμε ότι άμα γίνει ένα μέτρο υποχρεωτικό θα λύσει κάποια κοινωνικά προβλήματα. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δεν θα ε, φτιαχτούν θέσει εργασία και ανταγωνιστικότητα. Μπα και γίνεται το ανάποδο. Η ανάπτυξη και η ανταγωνιστικότητα οδηγεί σε κοινωνική ευημερία και σε ε, απασχόληση. Δεν έχουν θαυματικό, θαυματουργό χαρακτήρα τα υποχρεωτικά μέτρα. Αλλά, άρα εδώ δεν τα βλέπουμε σωστά τα πράγματα. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε κάποιους πόρους, κάποια κοινωτικά ταμεία και ακόμα έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας για να πετύχουμε την ε, αποτελεσματικότητα. Γι' αυτό σας λέω θα πρέπει να επιμείνουμε στο να χρησιμοποιήσουμε όχι την υποχρεωτικότητα των νόμων, αλλά την πιο προωθημένη τεχνολογία. Και έτσι να πετύχουμε ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα που θα φέρει τις λύσεις. Άρα, η πληροφορική, αυτή η κόμβη, η IC της πληροφορικής θα φέρουν τις λύσεις. Έχουμε και την ψηφιακή ατζέντα. Τις προτάσεις του Κοινοβουλίου και της Κομισιόν που σχετίζονται με τις i-cities, τις πόλεις της πληροφορικής και αυτά όλα θα μας βοηθήσουν για αυτήν τη διαδρομή που έχουμε να διανύσουμε μέχρι να πετύχουμε την αποτελεσματικότητα στη χρήση της ενέργειας. Προσέχετε λοιπόν αυτή την διάσταση. Ευχαριστώ. πολύ, Πρόεδρε. Βλέποντας ότι πέρασε η ώρα, θα προσπαθήσω να είμαι συντομότατη. Ευχαριστώ καταρχάς, κύριε Μπένσεν, και εσάς και όλους τους συναδέλφους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για αυτή την πρωτοβουλία. Για την έκθεση αυτή για την ενεργειακή αποδοτικότητα. Πάρα πολύ επίκαιρο θέμα. και από πλευράς χρονισμού θα συμβάλλει θετικότατα στην ανάπτυξη ευρωπαϊκών πολιτικών για την ενεργειακή αποδοτικότητα. Το επόμενο βήμα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υποβάλει γενική πολιτική για την ενέργεια, θέμα προσυζήτηση και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αρχές του επόμενου έτους θα συζητηθεί. Θα συμπεριλαμβάνεται και σημαντικό στοιχείο για την ενεργειακή αποδοτικότητα. Ποιος είναι ο σχεδιασμός για την ώρα. Για πρώτη φορά μια τέτοια γενική ενεργειακή στρατηγική θα αξιολογήσει και τη ζήτηση την ενεργειακή. Οπότε μπαίνει στο επίκεντρο των πολιτικών η ενεργειακή αποδοτικότητα. Πρόκληση για όλους. Η ενεργειακή ζήτηση, η ενεργειακή αποδοτικότητα, η εξοικονόμηση ενεργείας, όλα αυτά ε, είναι στα όρια της ε, επικουρικότητας και δεν είναι εύκολο να καλυφθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σήμερα πιστεύει ότι θα πρέπει να αναπτύξουμε άκρος φιλόδοξη ευρωπαϊκή πολιτική για την ενεργειακή αποδοτικότητα, ούτω ώστε να συμμετάσχουν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς. Εκείνοι κυρίως που θα εφαρμόζουν αυτή την πολιτική, κυρίως τα κράτη-μέλη και η τοπική αυτοδίκηση στα κράτη-μέλη. Στην πράξη λοιπόν χρειάζεται στρατηγική που θα καλύπτει το ζήτημα και οριζόντια αλλά θα πρέπει να αναπτυχθούν ακριβείς και φιλόδοξες πολιτικές όσον αφορά τους βασικούς τομείς κατανάλωσης. Θεματικές πολιτικές δηλαδή, για τα κτίρια. Ποιος ο ρόλος της ανακαίνησης των κτιρίων, μεταφορές, τι μπορεί να γίνει εκεί, για να συγκρατήσουμε την κατανάλωση στον τομέα των μεταφορών, κατανάλωση ορυκτών καυσίμων, βιομηχανία και ενεργειακές βιομηχανίες. Ξεκινάει η συζήτηση, Πρόεδρε. Θέλω να είμαι σύντομη και περιμένω περαιτέρω συνεργασία μαζί σας. Σας ευχαριστώ. Παίξαν για άλλη μια φορά για να κλείσουμε. Πολύ σύντομα θα πω απλώς ευχαριστώ για όλα τα σχόλια. Θα εργαστούμε όσο δυνατόν πιο σκληρά. Και στις διακοπές μας. Καλώς λέει ο Πρόεδρος. Μια παράκληση καταρχάς προς την ε, γραμματεία. Θα ήθελα να ρωτήσω εάν έχουμε υπόψη ακριβώς το τι έχει επιτύχει η βιομηχανία, γιατί πολλές φορές γίνονται ε, πρόοδοι που δεν είναι πάντοτε γνωστές. Μια άλλη παρατήρηση. 2 Σεπτεμβρίου έχουμε την επόμενη μας συνεδρίαση, δηλαδή μεσολαβούν οι διακοπές. Σας εύχομαι πολύ καλές διακοπές. Κύριε Μπένσεν, και για σας καλή ξεκούραση. Mm. Καλή δουλειά το καλοκαίρι και ευχαριστώ και τους διερμηνείς, λέει ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ.